Ladies and gentlemen. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας, σε όλους. Ας ξεκινήσουμε τη συνεδρίασή μας της Υποεπιτροπής Ασφάλειας και Άμυνας. Θα ήθελα να σας ανακοινώσω ότι για τη διερμηνία φυσικά δίδεται η προτεραιότητα στις γλώσσες των τακτικών μέλων της υποεπιτροπής μας. Όπως πάντα η συνεδρίασή μας δι... μεταδίδεται στο διαδίκτυο. Ας περάσουμε στην έγκριση της μέσης διάταξης. <clears throat> Εάν δεν υπάρχουν αντίλησεις μπορούμε να θεωρήσουμε ότι έχει εγκριθεί. Εντάξει, ευχαριστώ. απουσία σχολείων και αντιρρήσεων θεωρούμε ότι η μέρηση διάταξη έχει εγκριθεί και επιτρέψτε μου και ας περάσουμε στα πρακτικά εάν θέλετε της 1 η Οκτωβρίου 2015 Εάν έχετε κάποιες παρατηρήσεις ε, ή αντιρρήσεις Πρέπει να το πράξετε μέχρι το τέλος της συνεδριασής μας σήμερα, εάν δεν υπάρξουν τέτοιες αντιρρήσεις ή παρατηρήσεις και τα πρακτικά θα θεωρηθούν ότι έχουν εγκριθεί. Περνάμε τώρα στο πρώτο σημείο της ημερησίας διαταξής μας που είναι η παρουσίαση της μελέτης που έχουμε ζητήσει να εκπονηθεί τον Ιούνιο, αν θυμάμαι καλά, και το θέμα της ε, μελέτης αυτής είναι η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ασφάλειας και Άμυνας με, με τα υπάρχοντα μέτρα και διαδικασίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το, το κύριο Ινστιτούτο το οποίο ανέλαβε αυτή τη ε, μελέτη ήταν το κέντρο του Λουβέν για την ε, ε, ε, για τα θέματα συνολικής σφαιρικής στρατηγικής αντιμετώπισης. Ο κύριος ε, Κολεαράουμπε είναι αυτός ο οποίος θα παρουσιάσει αυτή τη μελέτη. Και η μελέτη αυτή έχει εκπονηθεί με τη βοήθεια εξεχόντων ε, πανεπιστημίων, το Νιούκας η και το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο, συγγνώμη, Κοίμπρα, όχι Πράγα, το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο των Βρυξελών, το οποίο εκπροσωπείται από τον κύριο που είναι ο δεύτερος ομιλητής μας, κυρίες και κύριοι λοιπόν, χωρίς περαιτέρω περιστροφές, θα δώσω το λόγο στον δόκτορα Ράουμπε και μετά στον κύριο Φίατ. Το λόγο κύριε Ράουμπε. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Η μελέτη αυτή για την υποστήριξη <clears throat> της Ευρωπαϊκής ε, ε, Άμυνας και Ασφάλειας με τα μέσα που είναι στη διάθεσή μας αντιμετωπίστηκε από το κέντρο του Λουβέν για, την, ε, για τις μελέτες σφαιρικής διακυβέρνησης Έχουμε κάνει αυτή τη μελέτη σε συνεργασία με πολλούς συναδέλφους από διάφορα άλλα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια που τα βλέπετε αυτά στην διαφάνεια αυτή. Οι εμπειρογνώμονες και οι ερευνητέ αυτοί μας φέρανε την εμπειρογνωμοσύνη τους σε διάφορους τομείς πολιτικής. Κάναμε διάφορες συνεντεύξεις με εκπροσώπους της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Φορέα Άμυνας, και η μελέτη μας εξετάζει το πώς η, η ΕΠΑ μπορεί να αντιμετωπίσει την, ε, τις ανάγκες της ασφάλειας και άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τονίζει ότι αυτό μπορεί να γίνει μονάχα σε συνεργασία με άλλους φορές και άλλες πολιτικές. Τούτου δεδομένου, τα άλλα εργαλεία τα οποία δεν είναι τα εργαλεία της ε, κοινή εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας θα πρέπει να παίξουν ένα υποστηρικτικό ρόλο. Δείχνει η μελέτη ότι τα περαιτέρω αυτά όργανα και οι πολιτικές μπορούν να παίξουν ένα ρόλο συνέργειας μεταξύ τους και με την εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας. Αν δούμε την επόμενη διαφάνεια. Η επόμενη διαφάνεια παρακαλώ. Βλέπετε ότι η εστίασή μας είναι στην ανάλυση του πολιτικονομικού πλαισίου της ε, κοινή εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας και βλέπουμε ότι είναι ένα ευρύτερο τμήμα της Γενικής Πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης δίνει στρατιωτικές και μη στρατιωτικές ικανότητες όπως ξέρετε υπάρχουν τα εργαλεία για την εσωτερική συνεργασία σε θέματα άμυνες που η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλιώς δεν θα είχε ούτε για τα θέματα εσωτερικής ολοκλήρωσης ούτε για την εξωτερική της δράση. Αλλά η μελέτη καταδεικνύει επίσης τι είδου μορφή έχει η κοινή αυτή πολιτική, ότι έχει ένα διακυβερνητικό χαρακτήρα και επομένως τονίζει ότι μια συνολική προσέγγιση που συνδέει αυτή την πολιτική με άλλες πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι απαραίτητη. Η μελέτη καταδεικνύει ότι το άρθρο 21 της ε, Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπογραμμίζει την ανάγκη να υπάρξει συνεκτικότητα μεταξύ των διαφορετικών τομέων πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρέπει να υπάρχει συνοχή και συνεκτικότητα σε ό,τι αφορά την εξωτερική και εσωτερική διάσταση της ΚΕΠΑ. Όλα αυτά μπορεί να οδηγήσουν και σε μεγαλύτερη συνεκτικότητα μεταξύ των θεσμικών οργάνων όταν δούμε τα προβλήματα για, την, το συντονισμό των πολιτικών μέσα στα πλαίσια της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης. Περαιτέρω προσπαθούμε να δούμε ποιο είναι το δυναμικό το οποίο δεν έχει τύχει εκμετάλλευσης ε, για την πολιτική αυτή, όπως παραγωγός η ειδική πλειοψηφία σε ό,τι αφορά ε, τα μία νεόφυτα για την ε, χρηματοδότηση τέτοιων ενεργειών ή την δημιουργία μόνιμης διαθρωμένης συνεργασίας. Επίσης, μας ενδιαφέρει αυτή η μόνιμη διαθρωμένη συνεργασία. Θεωρούμε ότι δεν έχουμε εξαντλήσει το δυναμικό αυτής της διαδικασίας και μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα η ρήτρα αμοιβαία υποστήριξης για αμυντικά θέματα. Για τις συστάσεις, και εδώ έχουμε στην επόμενη διαφάνεια, εδώ θέλουμε να εστιάσουμε στο στόχο της ε, συνεκτικότητος και την συνολική προσέγγιση που θα είναι τα οδηγά νήματα στην εξωτερική πολιτική μας ώστε να μπορέσουν οι διάφοροι εμπλεκόμενοι και τα διάφορα εργαλεία να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν όλες τις πτυχές των ενεργειών της ΚΕΠΑ. Επίσης τα, οι θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να γνωρίζουν ότι με τον τρόπο αυτό η ΚΕΠΑ πρέπει να οδηγήσει σταδιακά σε μια κοινή πολιτική άμυνα και επίσης οι νομικές ρήτρες και ευκαιρίες που δίνονται από τη Συνθήκη της Λισαβόνας θα πρέπει να διευκρινιστούν περισσότερο. Στην μελέτη αυτή περαιτέρω εστιάζουμε περισσότερο σε ειδικού τομείς πολιτικής ε, αφού έχουμε εξετάσει το νομικό πολιτικό πλαίσιο ε, εστιάζουμε ιδιαίτερα στην εξωτερική και την εσωτερική διάσταση για την, για την πολιτική κίνηση ασφάλειας και άμυνας. Και εδώ θέλω να αναφέρω ορισμένα θέματα σε σχέση με την ευρωπαϊκή πολιτική γειτονία σε ό,τι αφορά τις εσωτερικές πολιτικές, την ανάπτυξη και συνεργασία και ο Δανίλο, συναδελφό μου, θα πει περισσότερο για τι περιφερειακές πολιτικέ και τι πολιτικέ εμπόριου. Στην, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονιάς, γειτονίας η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ορισμένα εργαλεία που δεν εμπλέκονται στην ΚΕΠΑ και στην κοινή πολιτική άμυνα και ασφάλειας. Αυτό περιλαμβάνει την πρόθεση της ασφάλεια και της σταθερότητα και έχουμε μια σειρά από εκπροσώπους και αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ασχολούνται με τα θέματα αυτά. Δείχνει η μελέτη όμως ότι γενικά τα πολιτικά τμήματα τη αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πολύ μικρά, έχουν μονάχα ένα ή δύο άτομα και γενικά θα πρέπει να χρησιμοποιούνται περισσότερο <clears throat> τα πολιτικά τμήματα γιατί μπορούν να είναι εστιακά σημεία για περισσότερη πληροφόρηση και συντονισμό. Χρειάζεται επίσης περισσότερη χρηματοδοτική υποστήριξη από το εργαλείο για την πολιτική γειτονία τη Ευρωπαϊκή Ένωση για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε καλύτερα τα θέματα ασφάλεια. Και η συνθήκη τη Λισαβόνα έχει δώσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ισχυρά εργαλεία τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν και τα οποία θα πρέπει να τύχουν συντονισμού από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα όλο ένα και περισσότερο. Όταν έλθουμε τώρα στις συστάσεις, τονίζουμε ότι η συνεχιζόμενη αναθεώρηση της πολιτικής γειτονίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να οδηγήσει σε ένα οικονομικό και πολιτικό όραμα για να αντιμετωπίσουμε την ε, επίλυση συγκρούσεων και στην Μεσόγειο αλλά και στις χώρες της ανατολικής γειτονίας. Αυτή η αναθεωρημένη πολιτική θα πρέπει να αντιμετωπίσει την πολιτική και οικονομική λογική των συμφωνιών <clears throat> αναφερόμαστε ιδιαίτερα στις ε, ευρωμεσογειακές τέτοιες συμφωνίε σύνδεση και πρέπει να υπάρξει μια πιο ε, γενναιόδορη προσέγγιση προς την γεωργία. Η πολιτική μας λοιπόν στην Μεσόγειο και στην ε, Ανατολική Ευρώπη, εάν εγκριθούν, θα πρέπει να συνοδεύονται από πολιτικο-οικονομικά εργαλεία και επίσης εστιάζουμε ιδιαίτερα στην, στο θεσμικό συντονισμό μέσα στα πλαίσια αυτά και τονίζουμε ότι οι εμπειρογνώμονες ασφάλειας της ευρωπαϊκής αντιπροσωπείας είναι ένα πάρα πολύ χρήσιμο εργαλείο προς αυτή την κατεύθυνση. Σε ό,τι αφορά τώρα την συνεργασία για την ανάπτυξη, τονίζουμε ότι μπορούν να υπάρξουν συνέργειες μεταξύ των <clears throat> εργαλείων πολιτικής και ασφάλειας και τονίζουμε ότι η ευρωπαϊκή πολιτική άμυνα και ασφάλεια έχει αντιμετωπιστεί ω αποπέδη πολλέ φορέ στο παρελθόν, απομονωμένη, αλλά αυτό δεν ανταποκρίνεται στι πραγματικέ συνθήκε. Δεν υπάρχει, όπω ξέρετε, έλλειψη εργαλείων για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε κοινέ αναλύσει και αξιολογήσει για τα θέματα αυτά. <clears throat> και είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθούν όλα αυτά τα εργαλεία από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια τη πολιτική ασφάλεια. Υπάρχει εδώ η σύσταση ότι πρέπει να αναθεωρήσουμε την εμβέλεια και τη διευκόλυνση για την ειρήνη στην Αφρική και του εργαλείου που συμβάλλει στην ειρήνη και σταθερότητα. Πρέπει να εξετάσουμε λοιπόν και τα δύο αυτά εργαλεία, ενώ συγχρόνω χρειαζόμαστε ένα νέο χρηματοδοτικό εργαλείο, το οποίο ήδη είναι υποσυζήτηση. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να ενισχύσουμε τα πολιτικά τμήματα τη αντιπροσωπείες τη Ευρωπαϊκής Ένωσης για να μπορέσουμε να συντονίσουμε την εκπόνηση κοινών αναλύσεων που συνδυάζουν την ανάπτυξη και την ασφάλεια ώστε να υπάρξει πιο άμεση διάδραση με τις υπηρεσίες ανάπτυξης. Μπορούμε να δούμε επίσης ότι το προσωπικό που ασχολείται με την ανάπτυξη θα πρέπει να έχει μεγαλύτερη επίγνωση των προβλημάτων ασφάλειας του κράτους δικαίου κτλ και έρχομαι τέλος στις εσωτερικές πολιτικές. Εδώ έχει μια μεγάλη εργαλειοθήκη η Ευρωπαϊκή Ένωση για να αντιμετωπίσει την πολιτική ασφάλειας. Παραδείγματος χάρη είναι ενισχυόμενος ο ρόλος της Frontex στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ασφάλειας και μπορούμε να εστιάσουμε και στην συνολική προσέγγιση ως εργαλείο για να μπορέσει να συνδυάσει αυτά τα διαφορετικά εργαλεία σε σχέση με τις συστάσεις μας πρέπει να εστιάσουμε στην ανάγκη να ενεργοποιήσουμε όλα τα σχετικά εργαλεία τα οποία βρίσκονται στη διάθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να αντιμετωπιστούν οι εσωτερικές απειλές και επίσης η Ευρωπαϊκή Συνολική Στρατηγική θα πρέπει να διευκρινίσει καλύτερα τη στρατηγική προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να μπορέσει να γεφυρώσει καλύτερα τις εσωτερικές με τις εξωτερικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά. And now I pass on... Και δίνω το λόγο στον συνάδελφό μου τώρα, στον Daniel Field. Yes, please, floor is Έχετε το λόγο, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Ας δούμε την επόμενη διαφάνεια που αναφέρεται στην περιφερειακή πολιτική. Θα αναφερθώ σε δύο συγκεκριμένα τμήματα της μελέτης. Το πρώτο έχει να κάνει με την περιφερειακή πολιτική και το άλλο με την πολιτική στο τομέα του εμπορίου. Θα σας δώσω μια γενική περιγραφή των πολιτικών αυτών όπως έκανε ο συναδελφός μου και συνέχεια θα προχωρήσω σε κάποιες συγκεκριμένες συστάσεις στις οποίες καταλήξαμε στα πλαίσια της μελέτης μας. Εξ αρχής βέβαια πρέπει να σας πω ότι εγώ συνέταξα μόνο το τμήμα αυτό που είχε να κάνει με την πολιτική εμπορίου, ενώ άλλο συνάδελφο ασχολήθηκε με την περιφερειακή πολιτική. Θα ξεκινήσω πάντω με αυτή, με την περιφερειακή πολιτική. Όπω ξέρετε, η περιφερειακή πολιτική και τα διαρθρωτικά ταμεία μπορούν να διαδραματίσουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο όσον αφορά την έρευνα στον τομέα τη ασφάλεια και τη άμυνα. Και ήδη έχει γίνει αυτό από τη δεκαετία του 80. Βέβαια υπάρχουν συγκεκριμένες παράμετροι όσον αφορά τη χρήση των διαθροτικών ταμείων για την ε, έρευνα στον τομέα της άμυνας. Εδώ υπάρχουν πολύ συγκεκριμένοι κανόνες. Ουσιαστικά έχει γίνει μια έρευνα μόνο χρησιμοποιώντας τα ταμεία αυτά για τα είδη διπλής χρήσης. Θεωρούμε εμείς πάντως ότι θα πρέπει να δοθούν περισσότεροι πόροι και για άλλες μελέτες, πέρα από αυτές δηλαδή που έχουν γίνει μέχρι στιγμής, που έχουν να κάνουν κυρίως με τη μη στρατιωτική πτυχή. Δεν έχω επικεντρωθεί, δηλαδή, επικεντρωθεί αρκετά στην αμυντική διάσταση των ε, ερευνών αυτών και βέβαια αυτό οφείλεται σε διάφορους πολιτικούς λόγους. Πέρα όμως από τους πολιτικούς αυτούς λόγους βλέπουμε ότι όλο και περισσότερες από τις στρατικές ικανότητες που αναπτύσσουμε παγκοσμίω έχουν μια διπλή διάσταση, μια διάσταση διπλής χρήσης και αλληλοσυνδέονται όλο και περισσότερε οι εσωτερικές και εξωτερικέ δραστηριότητε Ευρωπαϊκή Ένωση, Πράγμα που σημαίνει ότι πολλά αγαθά ή πολλέ τεχνολογίε μπορούν διτά να χρησιμοποιηθούν τόσο για την εσωτερική όσο και την εξωτερική ασφάλεια. Για παράδειγμα, όσον αφορά τις τηλεπικοινωνίες ή τους δορυφόρους, βλέπετε ότι εκεί μπορεί να έχουμε εφαρμογέ που έχουν να κάνουν τόσο με την στρατιωτική όσο και τη μη στρατιωτική τεχνολογία. Αυτή τη στιγμή έχουν ξεκινήσει κάποιες προπαρασκευαστικές δράσεις για τα διευθυντικά ταμεία προκειμένου να επικεντρωθούμε περισσότερο στην αμυντική διάσταση των ειδών διπλής χρήσης. Τώρα, όσον αφορά την δική μας την μελέτη, εμείς επικεντρωθήκαμε περισσότερο στα υφιστάμενα κοινωνικά και διευθυντικά ταμεία που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας. Ξέρουμε αυτή τη στιγμή ότι το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Κοινωνικό Ταμείο χρησιμοποιούνται για την αμυντική μετάβαση, δηλαδή προκειμένου να περάσουμε από παλιά παρχημένα στρατόπεδα σε κάποιες πιο μοντέρνες μονάδες που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την βιώσιμη ενέργεια ή για την παραγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Το κοινωνικό επίση ταμείο έχει χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν και για λόγους αποκατάστασης ή υποστήριξης βετεράνων πολέμου. Βλέπετε δηλαδή ότι υπάρχει μια διαφορετική χρησιμοποίηση των ταμείων αυτών ήδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η υποστηριξη βετερανων πολεμου βλεπετε δηλαδη οτι υπαρχει μια διαφορετικη χρησιμοποιηση των ταμειων αυτων ηδη στην ευρωπαικη ενωση η συναδελφος μου που ασχολήθηκε με τον κλάδο αυτό μα είπε ότι εφόσον, ότι, έχουμε τα μέσα αυτά, δεν τα έχουμε χρησιμοποιήσει επαρκώ και δεν έχουμε επαρκή επικοινωνία και συντονισμό ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο που είναι αρμόδια για τον προπολογισμό, προκειμένου να έρχονται σε επαφή με τις εθνικές αρχές για να χρησιμοποιούν τους πόρους αυτούς από τα ταμεία αυτά, προκειμένου να βοηθηθούν τα κράτη-μέλη. Υπάρχει λοιπόν μεγάλη απόσταση ανάμεσα σε αυτά τα οποία θεωρητικά έχουν αποφασιστεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Κοινοβούλιο και αυτά τα οποία όντως υλοποιούνται από τα κράτη-μέλη. Και ξέρετε ότι πολλέ φορέ όταν λέμε εθνικέ αρχέ αναφερόμαστε και στι περιφερειακέ αρχέ, καθότι πρέπει και αυτέ να εγκρίνουν τη χρησιμοποίηση κάποιων διαφορετικών ταμείων. Η χρησιμοποίηση πάντω των διαφορετικών ταμείων και του κοινωνικού ταμείου είναι πολύ σημαντική, διότι ακόμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν ορισμένα κράτη-μέλη τα οποία χρησιμοποιούν παλιές υποδομές, παλιές στρατιωτικές υποδομές, οι οποίες ε, δεν ευθυγραμμίζεται με τις εξελίξεις ή τις ανάγκες που έχουμε στα πλαίσια της άμυνας και της ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ας μην ξεχνάμε ότι κάθε φορά που μετατρέπουμε παλιά στρατόπεδα σε νέες μονάδες, κάθε φορά που χρησιμοποιούμε τον κοινοτικό προπολογισμό για την κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας, επηρεάζονται και οι δραστηριότητες μετά του ΝΑΤΟ, γιατί ξέρετε ότι υπάρχει μια έντονη σύνδεση, συσχέτιση ανάμεσα στα όσα κάνουμε εμεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τι δραστηριότητε που αναλαμβάνει το ΝΑΤΟ. Θεωρούμε λοιπόν ότι θα πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη υποστήριξη από τα θεσμικά όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου οι περιφερειακέ αρχέ να μάθουν ότι υπάρχουν αυτά τα δραστηριακά ταμεία και ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διάφορου σκοπού. Ξέρω ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη έχουν εκπονήσει κάποιες μελέτες για το πώς θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για λόγους άμυνας ή διπλής χρήσης στα διαφορετικά ταμεία. Οι μελέτες αυτές είναι καλές. Ωστόσο, εμεί στι δικέ μα συστάσει λέμε ότι θα πρέπει να υπάρχει μια γενικότερη ευαισθητοποίηση και δεν θα πρέπει να, να παραμείνουμε μόνο σε κάποιε εκθέσει και μελέτε. Α περάσουμε τώρα στην πολιτική εμπορίου και εδώ έχω πλέον την πλήρη ευθύνη των όσων θα πω, γιατί έχω εγώ συντάξει το τμήμα αυτό της μελέτης. Η πολιτική εμπορίου είναι ένα σημαντικό τμήμα της κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας. Είναι ένα ζήτημα το οποίο έχουμε αντιμετωπίσει στο παρελθόν και ουσιαστικά έχουμε πει και παλιότερα ότι όντω η πολιτική εμπορία επηρεάζει την ασφάλεια και την άμυνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρετε ότι από ρυθμιστική πλευρά γίνεται μια διάκριση ανάμεσα στι εξαγωγέ όπλων και τι εξαγωγέ ειδών αγαθών διπλή χρήσεω. Έχουμε λοιπόν δύο ξεχωριστά καθεστώτα εξαγωγών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη μελέτη αυτή προσπάθησα να επικεντρωθώ περισσότερο στον αντίκτυπο που έχουν οι ε, εμπορικές συμφωνίες στην κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας. Ασχολήθηκα καταρχάς με το TTIP, με τη Διατλαντική Σχέση Εμπορίου και Επενδύσεων, όπου είπαμε ότι στα αρχικά στάδια, δηλαδή πριν από κάποια χρόνια, αν είχαμε συμπεριλάβει την άμυνα στο TTIP, τότε αυτό θα είχε ένα αντίκτυπο προφανώς στον τομέα της άμυνας στην Ευρώπη, όσον αφορά για παράδειγμα τις δημόσιες συμβάσεις στον τομέα της άμυνας. Από ό,τι φαίνεται όμως ο κλάδος αυτός δεν πρόκειται να υπαχθεί στο TTIP. Παρόλα αυτά υπάρχουν κάποιοι τομείς που έχουν να κάνουν με τις τεχνολογίες διπλής χρήσης και που θα μπορούσαν να υπαχθούν στο TTIP. Σε μια σύσταση που κάνουμε εμεί στη δική μα τη μελέτη, λέμε ότι θα πρέπει να υπάρχει μια καλύτερη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για τον αντίκτυπο που έχουν οι συμφωνίε ελευθέρου εμπορίου στον τομέα τη άμυνα. Και δεν αναφέρομαι μόνο στο TTIP, αναφέρομαι και στην εμπορική συμφωνία για τι χώρε του ειρηνικού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προφανώ δεν συμμετέχει στην TPP, δεν συμμετέχει επίσης και η Κίνα, αλλά ένα μεγάλο τμήμα της Ασίας συμμετέχει στην συμφωνία αυτή και αυτή η συμφωνία, η TPP, αντιστοιχεί περίπου στο 40% του παγκόσμιου ΑΕΠ. Αν αυτό συνδυαστεί με το ότι οι περισσότερες επενδύσεις στον τομέα της τεχνολογίας γίνονται πλέον στην Ασία και αν τα δούμε αυτά στα πλαίσια της γενικότερης προσπάθειας εξισορρόπησης που κάνουν οι Ηνωμένε Πολιτείες όσον αφορά τον ρόλο και την επιρροή που θέλουν να έχουν στην Ασία, τίθενται διάφορα ζητήματα εμπορίου και ανταγωνισμού όσον αφορά αυτή την πλευρά του πλανήτη. Επίσης ε, υπάρχουν και κάποιες ε, άλλες συμφωνίες όπως η Συμφωνία για το Εμπόριο Προϊόντων της Τεχνολογίας των Πληροφοριών σύμφωνα με την οποία καταργούν τη δασμή για κάποιους ε, σημαντικούς τομείς των νέων τεχνολογιών Η ημιαγωγή, GPS, αναφέρομαι γενικότερα σε τεχνολογίες και προϊόντα υψηλής τεχνολογίας και για τα οποία προβλέπεται πλέον ότι δεν θα επιβάλλονται δασμοί στα πλαίσια του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Και νομίζω ότι από ευρωπαϊκή πλευρά θα πρέπει να εξετάσουμε και αυτή τη συμφωνία και να δούμε τελικά ποια θα μπορούσαν να ήταν τα ωφέλη ή το κόστος το οποίο δημιουργείται για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι είμαστε πλέον σε θέση να γνωρίζουμε τι αντίκτυπα έχουν όλες αυτές οι συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου στον τομέα της άμυνας. Αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τον παγκόσμιο ανταγωνισμό, αλλά ουσιαστικά μπορεί να βοηθήσει την ε, λεγόμενη τεχνολογική αμυντική βάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για άλλη μια φορά επηρεάζονται και οι δραστηριότητε του ΝΑΤΟ. Ξέρετε ότι αυτέ οι συμφωνίε εμπορίου δεν επηρεάζουν μόνο την Ευρωπαϊκή Ένωση, επηρεάζουν ουσιαστικά τα κράτη-μέλη, επομένω κατά επέκταση και το ΝΑΤΟ. Λέμε λοιπόν εμεί ότι θα πρέπει να γίνονται γενικότερε μελέτε και αξιολογήσει για το πώ τελικά αυτέ οι συμφωνίε ελευθέρω εμπορίου μα επηρεάζουν. Και ολοκληρώνω σε αυτό το σημείο. Ωραία, σας ευχαριστώ. Έχω μόνο τον κύριο... Δύο μάλλον ομιλητές έχουν ζητήσει το λόγο. Κύριο Βενχάρτεν, αν δεν διαφωνείτε να μιλήσετε δεύτερος. Σας ευχαριστώ. Είναι πολύ χρήσιμη και ενδιαφέρουσα η έκθεση που μας παρουσίασαν οι συντάκτες προς το τέλος, νομίζω να δείξετε ένα σημαντικό θέμα. Και αν κάποιος ήθελε να κάνει μια κάποια επικριτική κρίση για την έκθεση αυτή είναι ότι δεν έχουμε λάβει υπόψη μας αρκετά τη σχέση μας με άλλους οργανισμούς. Είναι κάπως εσωστρεφής. Κοιτάμε μόνο τι συμβαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν ετέθη οπουδήποτε το ερώτημα κατά πόσον τελικά η ΚΕΠΑ είναι απαραίτητη σε συγκεκριμένους τομείς. Συχνά ακούμε ότι μια συνεκτική προσέγγιση είναι η καλύτερη δυνατή, αλλά θα πρέπει να δούμε νομίζω σε μεγαλύτερο βάθος τη σχέση μεταξύ της πολιτικής, ε, ε, των γενικών πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της στρατιωτικής τους διάθεσης. Έχουν πραγματικά μια σχέση συνέργειας. Ε, πώς λειτουργούν στην πράξη οι σχέσεις τους. Και κυρίως είναι απαραίτητο να υπάρχει σχέση μεταξύ αυτών των δύο πτυχών της πολιτικής η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει στη διάθεσή τους τους πόρους που τους έχουν δώσει τα κράτη-μέλη και επίσης κάποιες ικανότητες στρατιωτικές τις οποίες έχουν προσφέρει. Αλλά επίσης η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είχε τη διάθεσή τη δυνατότητα μάλλον, να υποστηριχθεί από μια σειρά πολυμερών οργανισμών, διεθνών οργανισμών. Και με εξέπληξε μία από τις συστάσεις ότι θα χρειαζόταν να αυξηθεί το προσωπικό στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πιο συγκεκριμένα στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Εγώ θεωρώ ότι είναι υπερβολικά ε, πολύ άριθμο το προσωπικό αυτών των υπηρεσιών, ενώ υπάρχει ε, επικάλυψη των αρμοδιοτήτων τους με τις δραστηριότητες άλλων οργανισμών. και στο κοινοβούλιο θα μπορούσε κανείς να πει ότι μπορούμε να κάνουμε οικονομία ιδίως στα θέματα του προσωπικού, αλλά η κατάσταση είναι ακόμα χειρότερη σε άλλες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άλλα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα την Επιτροπή. Πιθανώς να υπάρχουν άλλες προτεραιότητες, ε, νέες προτεραιότητες. Εκεί η συνήθιση αντίδραση είναι να προσλαμβάνεται νέο προσωπικό. Έτσι αυξάνεται διαρκώ το προσωπικό. Και εγώ αμφισβητώ ότι αυτό είναι το σωστό. Πολλέ από τις ε, δραστηριότητε αυτέ στρατιωτικού χαρακτήρα είναι δραστηριότητε τι οποίε αναλαμβάνουν τα κρατημέλη ε, εδώ και πάντα και άλλοι διεθνεί οργανισμοί Επομένω, θα έλεγα ότι η έκθεση σα μα δίνει τροφή για σκέψη. Έχετε συγκεντρώσει διάφορε ενδιαφέρουσε πληροφορίε. Ε, στόχος σας εξάλλου ήταν να δώσετε, να παρουσιάσετε τα ευεργετήματα, τα, θετικά στοιχεία της ε, ευρωπαϊκής πολιτικής. Έχω την αίσθηση ότι ξεκινήσατε από αυτό και αργότερα αναζητήσατε πληροφορίες για να υποστηρίξετε αυτήν την θέση. Ευχαριστούμε κυρία Γκόμες. Σας ευχαριστούμε για τη μελέτη που μας παρουσιάζετε. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα και ιδιαίτερα για τα κράτη-μέλη, για τους υπουργού Άμυνα, για να έχουν κάτι στα χέρια τους που θα τους διευκολύνει να σκεφτούν. Πώς θα αντιμετωπίσουν ακριβώς αυτές τις προκλήσεις που σας περιγράψατε. Γιατί κατά την άποψή μου το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η έλλειψη πολιτική βούληση στο επίπεδο των κρατών μελών να υιοθετήσουν αυτή την ολιστική προσέγγιση, να αποδεχτούν ότι μπορούν να λειτουργήσουν ε, συνεργατικά αυτές τις πολιτικές, να δημιουργήσουν συνέργειες. Και αυτό φαίνεται ακόμα περισσότερο σε καταστάσεις κρίσης όπως η προσφυγική και η μεταναστευτική κρίση. όπου διαπιστώνουμε ότι πρέπει να κινητοποιηθούν πολλών ειδών διαφορετική και ικανότητε διαφορετική πόροι, ενώ δυστυχώς αυτό που βλέπουμε και το διαπιστώνουμε τώρα με τη σύνοδο στη Βαλέτα, ότι η λύση που προκρίνεται είναι απλώς να ρίχνουμε λεφτά και να θεωρούμε ότι αυτό θα λύσει το πρόβλημα. Με κάποιον τρόπο οι άνθρωποι θα σταματήσουν να έρχονται προς την Ευρώπη. Και φυσικά αυτό δεν σημαίνει. Επομένως πιστεύω ότι η προσέγγιση που περιγράφεται, το όραμα αν θέλετε που περιγράφεται είναι ακριβώς αυτή που θα έπρεπε να έχουμε εμείς, όχι μόνο οι Υπουργοί Άμυνας, αλλά και εμείς για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να χρησιμοποιούνται οι δυνατότητες που έχει στη διάθεση της Ευρώπη. Και φυσικά αυτό πρέπει να ξεκινήσει από τα υψηλότερα κλιμάκια και δυστυχώς δεν υπάρχει τέτοια πολιτική βούληση, τουλάχιστον στα περισσότερα από τα κράτη-μέλη στις κυβερνήσεις τους δεν υπάρχει αυτή η πολιτική βούληση. Σε ορισμένα κράτη-μέλη αυτό οφείλεται σε άγνοια. Σε άλλα κράτη-μέλη δυστυχώς έχουν επιλέξει να μην επιτρέψουν στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση να λειτουργήσει. Και μιλώ κυρίως για τη Βρετανική κυβέρνηση εδώ, η οποία υπονομεύει την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Άμυνας, υπονομεύει την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική άμυνα εν τέλει. Και είναι λυπηρό ιδίω όταν γνωρίζουμε την επεμβαίνει ω βουλευτή από τη Μεγάλη Βρετανία. Πιστεύω ότι αυτό που λέτε δεν ισχύει. αντιθέτω, η συνεισφορά μα είναι δυσανάλογα μεγάλη. Η πρόεδρος επεμβαίνει Τζέφρι δεν είχατε το λόγο. Να τελειώσει η κυρία Γκόμε. και μετά αν θέλετε να πάρετε το λόγο. Κυρία Γκόμες. Ναι, λοιπόν, όπω έλεγα, ε, πράγματι είναι ακριβώ τραγικό επειδή η Βρετανία θα είχε, το Ηνωμένο Βασίλειο θα είχε τη δυνατότητα ε, να συνεισφέρει πολύ περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον, από οποιοδήποτε άλλο κράτο μέλο, επειδή έχει ήδη μια στρατιωτική δομή στη διάθεσή του που ακολουθεί την ολιστική προσέγγιση και ταιριάζει με αυτή την προσέγγιση, αλλά οποτεδήποτε τίθεται το θέμα στο ευρωπαϊκό ε, πλαίσιο απέχει. Και αυτό είναι τραγικό για όλου μα. Επίσης θέλω να σταθώ στη σημασία των θεμάτων που αναφερθήκατε σε σχέση με το εμπόριο. Όπως είπατε και εσείς, έχει τεράστιες επιπτώσεις ο τρόπος με τον οποίο εξελίσσεται το διεθνές εμπόριο. Ο λόγος που η TTIP δεν καλύπτει τις εξαγωγές όπλων δεν είναι για τον καλύτερο ή ερενικότερο λόγο, είναι επειδή δεν θα καλύπτεται συμφέροντα των ΗΠΑ κάτι τέτοιο δεν θα τα εξυπηρετούσε. Επίση, ο λόγος για τον οποίο δεν ε, ασχοληθήκαμε ιδιαίτερα με την TIPP είναι ακριβώς ο ίδιος λόγος με τον, για τον οποίο δεν ασχοληθήκαμε με το τι συνέβη τα τελευταία δεκαετία της ιδιωτικοποίηση και την διαρκή λιτότητα η οποία οδήγησε να έχουν στα χέρια τους πλέον δυνάμεις ε, ε, με στρατηγικά συμφέροντα να έχουν πλέον στα χέρια τους στρατηγική σημασίας υποδομές των ευρωπαϊκών κρατών και να σας δώσω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα επισκεφτήκα πρόσφατα την Κίνα και ο τρόπος, με, με εντυπωσίασε ο τρόπος με τον οποίο η Microsoft έχει αξιοποιήσει την βοήθεια του Αμερικανικού κράτους για να εδραιωθεί στην Κίνα. Αναρωτιέμαι Πώς έχουν αξιοποιηθεί για παράδειγμα δυνατότητες αυτές για την δημιουργία δικτύων επικοινωνιών διπλής χρήσης. Νομίζω έχουμε τις αποδείξεις στα χέρια μας που δείχνουν ότι τίποτα δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε και εξετάζονται στην έκθεση σας το καταλαβαίνει αυτό κανείς. ενέκριναν αυτή την κοινή θέση όσον αφορά τις εξαγωγές όπλων. Η Πρόεδρος ε, ζητώ συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά έχουμε και κάποιο περιορισμό χρόνου. Ε, ε, φτάστε καν στο συμπέρασμά σας. Τα είπα όλα. Εντάξει. Θα δώσω το λόγο στον ταξίαρχο Τζέφρι Φανόρντεν. Απλώς, εν συντομία Τζέφρι, για να απαντήσω σε αυτά που είπε η Άννα. Άννα, δυστυχώς, το Ηνωμένο Βασίλειο συμβάλλει υπεραναλογικά στις ενέργειες ε, της πολιτικής ασφάλειας και άμυνας, παραγωγικά χάρη στην επιχείρηση Αταλάντα. Έχουμε κάνει λοιπόν πάρα πολύ σημαντική συνεισφορά για τις ενέργειες στην Μεσόγειο. Δεν λέω ότι συμφωνώ με αυτό το οποίο γίνεται, απλώς θέλω να διαμφισβητήσω αυτό το σημείο. Ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν συμβάλλει Πράγματι συμβάλλει το Ηνωμένο Βασίλειο. Εγώ διαμφισβητώ τον τρόπο με τον οποίο συμβάλλει, αλλά αυτό είναι ένα διαφορετικό θέμα το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσω με τη δική μας κυβέρνηση. Δεν είπα ότι δεν συμβάλλει, λέει η Αναγκόμης. Λέω ότι μποϊκοτάρει, οπότε το βολεύει το Ηνωμένο Βασίλειο τις κοινέ ενέργειες. Εντάξει, λέει η Ο κύριος... Ε, θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω <clears throat> την ε, πρόεδρό μας τους και τους δύο ομιλητές και θέλω να σας ευχαριστήσω και για την παρουσίαση που μας έχετε δώσει. Η έρευνα αυτή έχει φυσικά σημαντικό περιεχόμενο και εκπαιδευτικό περιεχόμενο. Είναι απαραίτητο να αναλύσουμε καλύτερα την κατάσταση που έχουμε ενώπιόν μας. Και η κατάσταση είναι αυτή. Ότι οι συνθήκες της Λισαβόνα αναφέρεται στην αναγκαιότητα να υπάρχει κοινή πολιτική άμυνας και ασφάλειας, αλλά δεν έχουμε μια τέτοια πολιτική, έχουμε ψήγματα μονάχα αυτής της πολιτικής. Και νομίζω ότι θα πρέπει να συζητήσουμε για το γεγονός αυτό, ότι δεν έχουμε παρά μόνο ελάχιστα στοιχεία αυτής της πολιτικής. Μια συζήτηση που έγινε πριν από λίγο καιρό βλέπετε ότι υπάρχει μια σημαντική διαφορά απόψεων μεταξύ των κρατών μελών για τα θέματα αυτά. Θα ήθελα όμως να επιστήσω την προσοχή σας σε ένα άλλο θέμα, το οποίο είναι θέμα μεθοδολογίας. Όταν αναλύουμε την κοινή πολιτική ασφαλείας και άμυνας, κανονικά δίνουμε έμφαση σε θέματα άμυνας και σε στρατιωτικά θέματα. Όχι, αυτό είναι σφάλμα. Μια τέτοια προσέγγιση είχε χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν. Σήμερα όμως <clears throat> είναι αδύνατον να υπάρξει σωστή συζήτηση για την ασφάλεια της Ευρώπης χωρίς να αντιμετωπίσουμε τρία συγκεκριμένα ζητήματα. Πρώτον, η ασφάλεια ενέργειας. Πολύ ασθενικό σημείο, ένα από τα δύνατα σημεία της Ευρώπης. Ξέρουμε ότι η Ευρώπη εξαρτάται από πόρους ενεργειακούς που έρχονται από εκτός της Ευρώπης και εκεί δεν υπάρχει κοινό συμφερόντων, δεν υπάρχει κοινό πολιτικών το North Stream παραδείγματος χάρη. Έχει δείξει ότι υπάρχουν τέτοια προβλήματα. Ένας δεύτερος χώρος έχει να κάνει με τις κυβερνοεπιθέσεις και το κυβερνοέγκλημα. Και τρίτον έχουμε και μια κρίση προσφύγων. Και τα αποτελέσματα αυτής της ε, κρίσης επηρεάζουν την ασφάλεια της Ευρώπης. Έχω ακούσει την ανάλυση που παρουσίασαν οι ομιλητές μας σήμερα βλέπω δύο ζητήματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Πρώτα απ' όλα, να δούμε ποια στοιχεία ικανότητος ελείπουν και μας εμποδίζουν να έχουμε μια πραγματική πολιτική άμυνας και ασφάλεια σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα κράτη-μέλη έχουν αυτές τις απαραίτητες ικανότητες. Το πρόβλημα είναι όταν θέλουμε να δράσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τι λείπει λοιπόν, τι μας εμποδίζει να δράσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεύτερον, Ξέρουμε πολύ καλά ότι είναι ατελής ο μηχανισμός μας για τη λήψη αποφάσεων. <clears throat> Ενώ ξέρουμε ότι οι αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται με μεγάλη ταχύτητα. Βλέπετε τι γίνεται τώρα. Κάθε μήνα συνεδριάζει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και είναι να εξελίξει η κρίση των προσφύγων και χρειαζόμαστε να έχουμε μια πιο αποτελεσματική δράση. Τι μπορεί λοιπόν να αλλάξει αυτό το θέμα. κύριο Ε, θα ήθελα να πω κάτι το οποίο νομίζω ότι συμπληρώνει αυτά που είπε ο Πολωνός προλαλής σας. Δεν έχω να πω πολλά πράγματα περισσότερο καταρχήν γιατί είπε αυτά τα οποία ήθελα να πω και εγώ. Απλώς ήθελα να πω ότι τα θέματα ασφάλειας είναι θέματα κυριαρχικότητας. Δεν υπάρχει ευρωπαϊκή κυριαρχικότητα και γι' αυτό το λόγο δεν υπάρχει ευρωπαϊκή ασφάλεια και άμυνα. Το μόνο πράγμα το οποίο μπορούμε να κάνουμε είναι συνεργασία μεταξύ εθνικών κρατών. Αυτό προβλέπουν και οι συνθήκες, μια μορφή συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας με ενισχυμένα εργαλεία, όπως είναι η ενισχυμένη συνεργασία κτλ. Για όλα αυτά είναι απαραίτητο να δούμε τα κοινά σημεία για τα οποία μπορεί να λειτουργήσει αυτή η συνεργασία και να προσφέρει υποστέμενη αξία. Τεχνολογικά παραδείγματο χάρη μπορούμε να σκεφτούμε τα αεροσκάφη τα οποία τα μεταφορικά αεροσκάφη που θα οδηγήσουν σε μια αυτονομία της Ευρώπης, τα πυρηνικά υποβρύχια, του δορυφόρους. Να δούμε λοιπόν βασιζόμενοι σε κάτι τέτοιο, βασιζόμενοι στην έννοια της ανεξαρτησίας και της αυτονομίας της στρατιωτικής δράσης της Ευρώπης. Το ερώτημα είναι Πώ θα μπορέσουμε να το επιτύχουμε, γιατί είναι απαραίτητο να έχουμε αυτή την αυτονομία και ανεξαρτησία τη Ευρώπη σε ένα πολυπολικό κόσμο, να μην βασιζόμαστε ούτε στου Αμερικανού ούτε σε άλλε εξωτερικέ δυνάμει, να βρούμε με ποιο τρόπο μπορούμε να ενισχύσουμε την αυτονομία τη Ευρώπη και την ανεξαρτησία τη από ξενέ δυνάμει. Θα πρέπει να καθορίσουμε καλύτερα του τομεί όπου μπορούμε να συνεργαστούμε. Προφανώς υπάρχει το πρόβλημα της ενέργειας, των κυβερνοεπιθέσεων, επιθέσεων, τα προβλήματα αντιμετώπισης της τρομοκρατίας και φύλαξης των συνόρων μας. Όλα αυτά λοιπόν μου φαίνεται ότι δεν μας οδηγούν πουθενά αν δεν έχουμε μια πραγματική ευρωπαϊκή άμυνα. Δεν θέλει κάτι τέτοιο το Βασίλειο, στην πράξη ούτε και η Γαλλία θέλει κάτι τέτοιο. Λοιπόν, σταματήστε να ονειροπολείτε για κάτι το οποίο δεν γίνεται. <clears throat> Σε ένα τομέα λοιπόν που μπορούν τα κράτη-μέλη να συνεργαστούν, εκεί κάτι μπορούμε να κάνουμε, αλλά και πάλι επανέρχομαι σε αυτό που είπα, θα πρέπει να κάνουμε μια διάκριση μεταξύ των σημείων όπου η συνεργασία οδηγεί σε μια προσθέμενη αξία και εδώ κυρίω στα θέματα έρευνα και τεχνολογία. Εκεί μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλέ κοινέ και συμπληρωματικέ προσπάθειε. Μπορούμε να ξεκινήσουμε για κοινά προγράμματα που έχουν να κάνουν με μια ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια. Αλλιώ δεν θα έχουμε ποτέ ευρωπαϊκή προσθέμενη αξία και το ΝΑΤΟ θα είναι πάντα πιο ισχυρό από μια ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια. Τρίτο θα πρέπει να βρούμε όπου πραγματικά υπάρχει ανάγκη συνεργασία και όπου η συμπληρωματικότητα είναι απαραίτητη. Ευχαριστώ. Μέρση ε, λέει η πρόεδρος. Θέλε... Θέλω και εγώ να κάνω κάποιες παρατηρήσεις. Και εγώ θέλω να Συμφωνήσω απόλυτα με τον κύριο Ζέμκα για τα θέματα ασφάλειας στον ενεργειακό τομέα. Είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά. Πρέπει επίσης να σκεφτούμε ποια μέτρα, ποιε διαδικασίες θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε για να ενισχύσουμε την ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια. Θα πρέπει να δούμε από πού έρχονται οι απειλέ προς την ασφάλεια και την άμυνά μας και να δούμε πώς μπορεί να γίνει σωστή χρήση των μέτρων και των πολιτικών μας. Κύριε Χάουμπε, είπατε στην αρχή την ανατολική εταιρική σχέση. Αποτελεί ένα πρόβλημα. Αν δούμε τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης όπως στην Ουκρανία. Τα θέματα είναι πάρα πολύ σαφή. Όταν λάβουμε υπόψη επίσης την Λευκορωσία ή την Αρμενία, τα πράγματα είναι ασαφέστερα λιγάκι. Πρέπει λοιπόν να έχουμε μια ποικιλία μέτρων και πολιτικών για να αντιμετωπίσουμε τα θέματα αυτά, για να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε καλύτερα σε πολιτικό επίπεδο τα προβλήματα αυτά. Έχετε το λόγο λοιπόν, κύριε Χάουμπε. Και κύριε έχετε το λόγο. Thank you, thank you very... Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ για όλες αυτές τις παρατηρήσεις και όλες αυτές τις ερωτήσεις που θέσατε. οι οποίες βασίζονται στην σημερινή παρουσίαση. Να απαντήσω καταρχάς στις ερωτήσεις, τουλάχιστον να απαντήσω σε αυτές που θεωρώ ότι απευθύνονται σε μένα. Κύριε Βανόρδεν, θα ήθελα να τονίσω ότι στη μελέτη μας αυτή όντως λέμε ότι μπορεί να υπάρχουν δυνατότητες συνεργασίας με άλλους οργανισμούς. Αυτό όμως δεν είναι το βασικότερο, ουσιαστικότερο ζήτημα της έκθεσης. Λέμε όμως ότι θα μπορούσε να δημιουργηθεί μια άτυπη ομάδα συντονισμού διαχείριση κρίσεων στα πλαίσια του ΝΑΤΟ ή του ΟΑΣΕ. Προσπαθούμε δηλαδή να τονίσουμε τη διάσταση αυτή της διοργανικής συνεργασίας και προφανώς ξέρουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ο μόνος φορέας που παρέχει ασφάλεια και άμυνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ακριβώς για αυτό το λόγο πρέπει να υπάρχει συνεργασία και συντονισμός και με άλλους οργανισμούς όσον αφορά το προσωπικό στο οποίο αναφερθήκατε. Θα ήθελα να πω ότι αν δούμε τις ε, αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταρχάς και κυρίως το πολιτικό τμήμα των αντιπροσωπείων αυτών, όντως υπάρχουν πολύ λίγοι υπάλληλοι από τον πολιτικό τομέα σε σχέση με άλλα τμήματα των αντιπροσωπείων αυτών. Το ερώτημα που τίθεται λοιπόν είναι πώς θα μπορούσαμε εμείς να βελτιώσουμε το συντονισμό ανάμεσα το τμήμα της ασφαλείας, τον κλάδο ασφαλείας και άμυνας και τον κλάδο εκείνο, τα τμήματα εκείνων που έχουν να κάνουν με το εμπόριο για παράδειγμα και αναφέρουμε πάντα σε αντιπροσωπείες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μία λοιπόν από τις συστάσεις της μελέτης μας είναι ότι θα πρέπει να αναλύσουμε λίγο περισσότερο την πολιτική προσωπικού για τους υπαλλήλους των αντιπροσωπιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είπαμε ότι πρέπει να αυξηθεί αναγκαστικά το προσωπικό, απλώς είναι καλύτερα να γνωρίζουμε ποιος κάνει τι. Δηλαδή, ποιοι είναι οι υπάλληλοι εκείνοι οι οποίοι εργάζονται για ζητήματα αναπτυξιακής συνεργασίας και οι άνθρωποι αυτοί γνωρίζουν πώς εξελίσσεται το τομέα της άμυνας και της ασφάλειας και από την άλλη πλευρά θα πρέπει να δούμε αν οι ίδιες οι αποστολές κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας γνωρίζουν για όλα αυτά τα εργαλεία αναπτυξιακή συνεργασίας τα οποία διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό προσπαθούμε να πούμε ουσιαστικά με τη μελέτη μας, να καταφέρουμε να εμβαθύνουμε, να επικεντρωθούμε σε όλες αυτές τις διαφορετικές διαστάσεις. Όσον αφορά τώρα το ποιες ικανότητες θα πρέπει να έχουμε προκειμένου να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί σε ευρωπαϊκό τουλάχιστον επίπεδο και έρχομαι εδώ πέρα στο ερώτημα του κύριου Ζέμκε. Ως προς αυτό, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται στη συνεργασία και στο συντονισμό στον τομέα της κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας. Προφανώς η κυριαρχία παραμένει εθνική, παραμένει στα κράτη-μέλη, αλλά αυτό το οποίο λέμε στη μελέτη αυτή είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να παρουσιάσει ένα συγκεκριμένο αφήγημα στα κράτη-μέλη, να καταφέρει κατά αυτόν τον τρόπο να προσδώσει μια ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία σε όλα αυτά τα εργαλεία, σε όλες αυτές τις ικανότητες που έχουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα μπορούσε κατά αυτόν τον τρόπο να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα της δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατά αυτόν τον τρόπο θα είχαμε αν θέλετε και ένα όραμα, ένα αφήγημα εντό αγωγικών το οποίο θα μπορούσαμε να παρουσιάσουμε προς τα κράτη-μέλη και κατά αυτόν τον τρόπο θα τα κινητοποιούσαμε να συνεργαστούν και να συντονιστούν περισσότερο σε ευρωπαϊκό επίπεδο και δεν θα πρέπει να επικεντρωθούμε μόνο στην κοινή πολιτική ασφάλεια και άμυνα ως μεμονωμένη, αποκομμένη πολιτική αλλά ως πολιτική η οποία αρμονικά διασυνδέεται και συντονίζεται και με άλλα μέσα, τα λεγόμενα κοινοτικά μέσα νομίζω πλέον ότι θα πρέπει να τα ονομάζουμε μέσα ασφαλείας της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθότι επιτελούν και αυτό το ρόλο. Και μία τελευταία παρατήρηση τώρα όσον αφορά την ανατολική εταιρική σχέση. Προφανώς λέμε στη μελέτη και το τονίζουμε αυτό ότι υφίστανται πολλά προβλήματα στα πλαίσια της πολιτικής αυτής και όντως το έχουμε εντοπίσει αυτό στη μελέτη ότι ε, τα πάντα εξελίσσονται Σύντομα θα έχουμε μάλιστα και μία αναθεώρηση της ε, πολιτικής αυτής. Λέμε λοιπόν ότι ε, θα πρέπει εδώ πέρα να επανεξετάσουμε την όλη προσέγγιση που έχουμε στα πλαίσια της ανατολικής εταιρικής σχέσης. Και κυρία Πρόεδρε, με την άδειά σας, ε, μία τελευταία παρατήρηση. Νομίζω ότι θα πρέπει να εστιαστούμε περισσότερο και στο Αζερβαϊτζάν. Ξέρετε ότι η χώρα αυτή σχεδιάζει να αποχωρήσει από την Euronest, από το φόρουμ συνεργασία της Euronest και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, θα προκαλέσει περαιτέρω προβλήματα στην ανατολική εταιρική πολιτική. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Φιώτορ έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι ένα από τα γενικότερα βασικά θέματα που έχουμε εδώ πέρα δεν είναι να γίνει μια διχοτόμηση μεταξύ διαφορετικών οργανισμών, Ευρωπαϊκή Ένωση, ΝΑΤΟ και το καθεξής. Το πιο ουσιαστικό ζήτημα που εντοπίσουμε στη μελέτη δεν είναι τόσο πολύ τα θεσμικά όργανα και το πώ λειτουργούν, αλλά πώ λειτουργούν τα ίδια τα κράτη-μέλη. Αναφερθήκατε στην κυριαρχία των κρατών μελών. Εμα νομίζω ότι τα κράτη-μέλη συνειδητοποιούν όλο και περισσότερο ότι ο όρο άμυνα είναι πλέον ένας αδιέρετος όρος. Αναφερθήκαμε αυτή τη στιγμή στην ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, στην ενεργειακή ασφάλεια. Ξέρετε ότι Υπάρχουν όλες αυτές οι πτυχές στην ασφάλεια, υπάρχει καθαρή στρατιωτική ασφάλεια με την οποία ασχολείται το ΝΑΤΟ, υπάρχουν πάρα πολλοί τομείς όμως που επηρεάζουν πλέον την ασφάλεια των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θεωρώντας λοιπόν ότι η ασφάλεια και άμυνα είναι έννοιες αδιέρετες, λέμε στη μελέτη αυτή ότι ήδη υπάρχουν αυτή τη στιγμή ικανότητες, εργαλεία, μέσα, τα οποία δεν έχουν να κάνουν μόνο και αποκλειστικά με την κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας, αλλά μπορούν να επηρεάσουν θετικά και τα ίδια τα κράτη-μέλη, αν χρησιμοποιήσουν αυτά τα εργαλεία. Δεν λέμε αυτή τη στιγμή ότι πρέπει να δημιουργηθούν περισσότερα εργαλεία, δεν λέμε ότι θα πρέπει να τροποποιηθούν οι ίδιε οι συνθήκε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Λέμε απλώ ότι τα κράτη-μέλη ήδη έχουν αποδεχθεί μία δέσμη μέτρων, την οποία δεν έχουν αξιοποιήσει πλήρω ακόμα. Αυτό ουσιαστικά λέμε στη μελέτη. Καταγράφω λοιπόν όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία θίξατε, ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, ενεργειακή ασφάλεια και το καθεξής. Και ακριβώς επ' αυτού θεωρώ ότι δεν είναι μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή που θα πρέπει να αναλάβει δράση, αλλά θα πρέπει να ζητήσουμε ακόμα και από τους εταίρους μας στο ΝΑΤΟ να μας πούνε ποια είναι η δική τους άποψη, γιατί όντως επικεντρώνονται περισσότερο στην αμυντική πλευρά των πραγμάτων, αλλά γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι δεν μπορεί κανείς να εξετάσει την ε, αμυντική ασφάλεια ή τη στρατιωτική ασφάλεια μεμονωμένα και ξεχωριστά από οποιαδήποτε άλλη πολιτική που άπτεται και αυτή της ασφάλειας. Επομένως, είναι σημαντικό να πούμε ότι υπάρχουν εργαλεία και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που μπορεί να υποφελεί τόσο για την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και για άλλου οργανισμού όπω το ΝΑΤΟ. Ξέρω ότι υπάρχει μια έντονη πολιτική διάσταση στον τομέα αυτό, ξέρω ότι υπάρχουν αρκετοί πολιτικοί ενδιασμοί, ο Γενικός Γραμματέας Στόλτεμπερκ, η ε, ύπατη εκπρόσωπος Μογκερίνη έχουν προωθήσει την ε, σφαιρική αυτή χρησιμοποίηση των εργαλείων αυτών και ακριβώς αυτό λέμε και εμείς στη μελέτη μας, ότι θα μπορούσε να υπάρξει ένας καλύτερος συντονισμός και περισσότερες συνέργειες, Κύριε Γκόμες, ε, όσον αφορά το ζήτημα της ευρωπαϊκής πολιτικής εμπορίου. Συμφωνώ με τα όσα είπατε και πρέπει να πούμε και κάτι ακόμα. Έχουμε εδώ, θέλετε, ένα διτό πρόβλημα. Από τη μία πλευρά έχουμε επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση που παράγουν αμυντικό εξοπλισμό και που ιδίω ε, κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου είχαν μια πολύ υψηλή και σταθερή ζήτηση από τις κυβερνήσεις τους. Αυτή τη στιγμή όμως μιλάμε όλο και περισσότερο για μεταφορά τεχνολογίας στο εξωτερικό, για το γεγονός ότι υπάρχουν πάρα πολλές ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που χάνουν την ανταγωνιστικότητά τους αυτό γίνεται ακριβώ επειδή εμεί δεν καταναλώνουμε αρκετά αμυντικά, αν θέλετε, προϊόντα, αμυντικού εξοπλισμού πλέον στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένω, πρέπει να αναζητήσουν μια αγορά στο εξωτερικό επιχειρήσει αυτέ. Η όλη αμυντική βιομηχανία έχει επίση παγκοσμιοποιηθεί και νομίζω ότι και αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μα. Εξετάζοντα όμω την κατάσταση ω έχει στον κόσμο αυτή τη στιγμή και επικεντρώμενο περισσότερο στα όσα βλέπουμε στην Ουάσιγκτον, βλέπουμε ότι υπάρχει μια διάδοση των αμυντικών τεχνολογιών παγκοσμίω και όντω αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να είμαστε όσο στρατηγικά θα θέλαμε όσον αφορά το ζήτημα αυτό της αμυντικής στρατηγικής εξάρτησης. Ξέρετε ότι εδώ πέρα όντως υπάρχει μια πολύ έντονη πολιτική διάσταση. Πάλι εδώ πέρα θα πρέπει να δούμε ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε βρίσκονται στην πρώτη γραμμή κάθε φορά που λένε ότι θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση από στρατηγική πλευρά να γίνει πιο αυτόνομη, να αναλάβει περισσότερε αυτόνομε στρατηγικέ πρωτοβουλίε. Όταν λέω λοιπόν, όταν αναφέρομαι στην αυτονομία αυτή και την ανεξαρτησία αυτή, δεν λέω ότι δεν χρειαζόμαστε το ΝΑΤΟ, αλλά χρειαζόμαστε καλύτερη συνεργασία με το ΝΑΤΟ. Turkey in the EU, e good news. Χαίρομαι που βλέπετε συνεργασία και με άλλους ε, οργανισμούς εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καλά τα αυτά. Σας ευχαριστώ κύριε για αυτή τη συζήτηση και για την παρουσίαση της μελέτης σας. η οποία πραγματικά πιστεύω ότι πρέπει να τη υπόψη του οι κυβερνήσει των κρατών μελών τη Ένωση. Σίγουρα προσωπικά θα προσπαθήσω ο Πολωνός Υπουργό Άμυνα να τη λάβει υπόψη του. Γιατί φύγεται και ενδιαφέροντες τομεί, όπω για παράδειγμα τη χρήση των διαρθρωτικών ταμείων ή ακόμα και την ε, κοινωνικά προβλήματα, επίλυση κοινωνικών προβλημάτων, όπως για παράδειγμα τα προβλήματα των βετεράνων. Μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο σημείο τη μέρης διάταξη. Well, Φαίνεται ότι η Αταλάντα δεν είναι τόσο συναρπαστική όσο νόμιζα. Θα πρέπει να υπομισθώ εγώ το έργο του να σας παρουσιάσω τα θέματα της Αταλάντας. Αυτό είναι το επόμενο σημείο της ημερησίας διάταξης. Είναι η ε, απόδοση πεπραγμένων σε σχέση με την αποστολή της ε, Επιτροπής μας στο Northwood, στο στρατηγείο της ε, Αταλάντα που έγινε στις 24 Σεπτεμβρίου. Ήταν μια μικρή αποστολή με τρία άτομα, τρεις βουλευτές συνολικά. Εγώ ως πρόεδρος της υποεπιτροπής, τον κύριο Φανόρδεν, και τον κύριο Κίρτσο. Δυστυχώ δεν είναι παρόντα τα άλλα δύο μέλη αυτής της ε, αντιπροσωπεία. Γι' αυτό θα σας πω εγώ εν συντομία πώς πήγε αυτή η αποστολή. ναι, πράγματι ήταν μια πολύ ατυχή στιγμή που εμπόδισε την κυρία να έρθει σε αυτή την αποστολή και αυτή η ιδέα. Πράγματι ήταν μια σύντομη μονοήμερη επίσκεψη στο Northwood ήταν πάρα πολύ σημαντική γιατί συνέπεσε με την εκκίνηση της ε, ε επιχείρησης Σοφία της ε, EUNAFOR Σόφια λοιπόν η κυρία Μογκερίνη ως αντιπρόεδρος της ε, Κομισιόν ήταν στη Ρώμη την ίδια μέρα στα αρχηγεία της επιχείρησης Σόφια και ήταν εκεί και ο διοικητής της ε, Αταλάντα για να μεταλαμπαδεύσει την εμπειρία του στα πλαίσια αυτής της ε, ενέργειας σε αυτούς οι οποίοι θα συμμετείχαν στην ε, επιχείρηση Σόφια. Μας υποδεχτήκανε φυσικά ο αναπληρωτής διοικητής της Αταλάντα Ο υπονάβαρχος, ο οποίος είναι ο αναπληρωτής λοιπόν, Ήταν πολύ καλά λοιπόν. Μια πολύ καλά προετοιμασμένη ενημέρωση που μας δόθηκε για να μας παρουσιάσει όλες τις πτυχές της επιχείρησης Αταλάντα. Με ποιο τρόπο γίνεται η συλλογή πληροφοριών πώς γίνεται η διάδραση με τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η συνεργασία επίσης με τον επιχειρηματικό κόσμο ήταν κεφαλαιώδης για την επιτυχία της επιχείρησης γιατί προφανώς η Αταλάντα ήταν η πιο επιτυχημένη ευρωπαϊκή επιχείρηση στην περιοχή αυτή μαζί με άλλες επιχειρήσεις, άλλες δύο επιχειρήσεις. Είχε μεγάλη επιτυχία. Για να μπορέσει να εξαλείψει ή τουλάχιστον να μειώσει τις τρομοκρατικές ενέργειες στο κέρας της Αφρικής και ιδίως την πειρατεία. Και είχε μεγάλη επιτυχία για να φέρει τους ε, εγκληματίες αυτούς που είχαν κάνει αδικήματα κατά των επιχειρήσεων αυτών ενώπιον της δικαιοσύνης. Ήμασταν ιδιαίτερα Ευήκοη σε αυτά που μα παρουσίασαν από την επιχείρηση Αταλάντα για να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε καλύτερα τι μελλοντικέ δράσεις τι οποίε μπορεί να εμπλακεί η EU, EU Nav for Med. Σα υπενθυμίζω ότι από, πρώτη, από την 1η ε, Δεκεμβρίου θα έχουμε τον ε, διοικητή της ε, Σόφια εδώ στην Επιτροπή μα κάποια στιγμή. Είναι πολύ σημαντική η εμπειρία λοιπόν αυτή που θα αποκομίσουμε και στο Northwood μπορέσαμε να επισκεφτούμε το αρχηγείο της Μάρκομ του ΝΑΤΟ, το κέντρο ναυτικών επιχειρήσεων του ΝΑΤΟ και να ακούσουμε και τη δική τους άποψη για το θέμα αυτό. Επειδή ο κ. Σίκλατ είναι ήδη εδώ και έχουμε πολύ σημαντικές συζητήσεις πρέπει να κάνουμε για την κεντροαφρικανική δημοκρατία. Μπορούμε να σταματήσουμε εδώ με την Αταλάντα. Δεν ξέρω τώρα αν κάποιο μέλος θέλει να πει κάτι, ο κ. Λαντσπέργης, ο κ. Φουντσουλίτσα, η κυρία Γκόμης θέλουν να πούν κάτι. Όχι, δεν θέλουν να πούνε κάτι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ λοιπόν. Και θα περάσουμε στο επόμενο σημείο που είναι η ανταλλαγή απόψεων με ένα γνωστό μας ε, τον ε, Κλόντι από την ε, Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και έχει να κάνει με το ζήτημα της επιχείρησής μας στην Κέντρο Αφρικανική Δημοκρατία και χωρίς περαιτέρω περιστροφές Ξέρετε ότι είναι πολύ πολύπλοκη και η δύσκολη κατάσταση εκεί για πολλούς λόγους. Δίνω το λόγο στον κύριο Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα σε όλους. Ζητώ συγγνώμη που αργοπόρησα και λίγο. Ιδιαίτερος χαρούμενος που μπορώ να σας μιλήσω σήμερα εδώ για τις επιχειρήσεις μας στην κεντρική κεντροαφρικανική δημοκρατία. Προσπαθώ να εξετάσω το θέμα από πλευρά κοινή εξωτερικής πολιτικής έναντι της χώρας αυτής. Η EU-MAM είναι τα αρχικά της Ευρωπαϊκής ε, Στρατιωτικής ε, Αποστολής. Θα ξεκινήσω από μια παρουσίαση σχετικά με αυτή και αργότερα ε, θα ήθελα να συζητήσουμε πώς μπορούν να εξελιχθούν τα πράγματα στο μέλλον, πώς θα μπορέσει να παρασχεθεί ε, διαρκής υποστήριξη στην κεντροαφρικανική δημοκρατία, κυρίως όσον αφορά την εκπαίδευση των στρατιωτικών της δυνάμεων και επίσης να σκεφτούμε ε, ορισμένα από τα διδάγματα που μπορούμε να αντλήσουμε από την EU 4 Car, την επιχείρηση στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία δηλαδή, όπου διαπιστώσαμε ότι τα Ηνωμένα Έθνη ε, θα ήθελαν να χρησιμοποιήσουν τον τρόπο δόμησης της ε, επιχείρησης αυτής ως υπόδειγμα. για τον τρόπο με τον οποίο μια περιφερειακή ένωση μπορεί να ε, λειτουργήσει στον ενδιάμεσο χρόνο μέχρι να καταφέρουν να αναπτυχθούν μεγαλύτερες δυνάμεις και ανώκρονο σε μια περιοχή. Όπως θα θυμάστε, η επιχείρηση αυτή ξεκίνησε μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της EU 4 Car, EU, EU λοιπόν, καθυστέρησε η λήξη της, η παράδοση της κοιτάλης προς τα δυνάμεις του ΟΗΕ είχε προγραμματιστεί να γίνει πέρυσι το Δεκέμβριο, αλλά μετά από αίτημα του Προέδρου της χώρας ε, και εξαιτίας ορισμένων δυσκολιών ε, καθυστέρησε η παράδοση και έγινε τον Μάρτιο. Ήταν μικρή η δύναμη, ε, με 60 άτομα προσωπικό η ενώ συγκριτικά η η u 4 ήταν 450. Στόχος ήταν η στενή συνεργασία με τις δυνάμεις του ΟΗΕ που έχουν αναπτυχθεί εκεί, στην περιοχή. Και είχε διτό στόχο. Πρώτον, να παράσχει συμβουλές προς την κυβέρνηση και τις αρχές της κεντροφυκρανικής δημοκρατίας, συγκεκριμένα το Υπουργείο Άμυνας, για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να δομήσει και να οργανώσει τις ένοπλες δυνάμεις ε, της χώρας. Και δεύτερον, να υποστηρίξει και να προετοιμάσει μια διαδικασία SSR Ε, υποστήριξη στον τομέα της ασφάλειας. Βεβαίως υπήρξε στενή συνεργασία με την αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία και όλες, όλα αυτά τα προγράμματα ε, συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας και άμυνας έχουν δώσει δυνατότητα στην αποστολή της Ένωσης να ε, γνωρίζει πώς βοηθάμε τη χώρα αυτή στον τομέα αυτών. Η εμπειρία λοιπόν που αποκομίσαμε από αυτή την αποστολή είναι η εξή. και μια προσέγγιση από, κάτω, από πάνω προς τα κάτω. Δηλαδή, να ε, δημιουργηθεί, να στηθεί ένα ε, ε, σύστημα ιεραρχίας, ε, στρατιωτικής ιεραρχίας, ε, λειτουργικό από πάνω προς τα κάτω. Αυτό έλειπε ε, απολύτως στις κεντροαφρικανικές ένοπλες δυνάμεις. Επομένω ήταν απολύτως απαραίτητο να δημιουργηθεί πριν ξεκινήσει οποιαδήποτε προσπάθεια αναδιοργάνωσης των ενόπλων δυνάμεων. Πριν ξεκινήσει οποιαδήποτε προσπάθεια αναδιοργάνωσης πρέπει να είναι ξεκάθαρος ποιος θα είναι ο ρόλος του καθενός στο σύστημα, στην ιεραρχία που δημιουργείται. αρχικά της στάδια η ε, αποστολή εστίασε στο να παρέχει συμβουλές κυρίως στο Υπουργείο Άμυνας αλλά αργότερα επεκτάθηκε ε, στο Γενικό Επιτελείο και σε άλλες ε, υποστηρικτικές μονάδες. Ε, ξεκινώντας από πάνω προ τα κάτω στην ιεραρχία όπως σας έλεγα. Αντιμετωπίστηκαν διάφορα προβλήματα. Πρώτα απ' όλα ε, ήταν δύσκολο να βρεθούν ε, οι κατάλληλοι συνομιλητές στα όλα τα επίπεδα του συστήματος. Πρώτα απ' όλα έπρεπε να ενθαρρύνουμε το Υπουργείο Άμυνα να αναλάβει το ρόλο του, να παίξει το ρόλο του ω Υπουργείο Άμυνα. Βέβαια το ευτυχές είναι ότι τουλάχιστον όσον αφορά το Υπουργείο Άμυνα σημειώθηκε επιτυχία. Λειτουργεί πλέον ικανοποιητικά. Επίσης ήταν σημαντικό να διαχωριστούν οι αρμοδιότητες ανάμεσα στο Υπουργείο Άμυνα, στο πολιτικό προσωπικό και τις ένοπλες δυνάμεις στο στρατιωτικό προσωπικό και να είναι ξεκάθαρες οι αρμοδιότητες του ενός και του άλλου και στις δύο πλευρές. Ο στόχος είναι το, η νέα ιεραρχία, η, η, η νέα δομή να αρχίσει να λειτουργεί από το 2016. Αυτό λοιπόν όσον αφορά την παροχή συμβουλών για την στρατιωτική οργάνωση. Δεύτερος στόχος ήταν να δημιουργηθεί μια δικτύωση γιατί Όταν κάποιος προσπαθεί να δημιουργήσει μια αποτελεσματική στρατιωτική ιεραρχία, δεν αρκεί να απευθύνεται και να ασχολείται μόνο με τους στρατιωτικούς ή με το Υπουργείο Άμυνας. Πρέπει να συνεργαστεί και με άλλα πολιτικά πρόσωπα, όπως για παράδειγμα τον, τον Πρωθυπουργό, το Γραφείο του Πρωθυπουργού και άλλα Υπουργεία, έτσι ώστε οι ένοπλες δυνάμεις να ταιριάξουν με την υπόλοιπη πολιτική δομή που δημιουργείται στη χώρα. Γι' αυτό λοιπόν η αποστολή ε, φρόντισε να το κάνει αυτό και επίσης να έχει στενές σχέσεις με την αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη χώρα. Γιατί θα ξαναέρθω σε αυτό. Στο μέλλον η ε, αποστολή της Ένωσης ε, στη χώρα αυτή θα έχει πολύ σημαντικό ρόλο να παίξει στα επόμενα project, στα επόμενα σχέδια που έχουμε στρατιωτικής συνεργασίας. και επίσης υπήρχε και πολύ στενή συνεργασία με τις δυνάμεις του ΟΗΕ. Εξίσου σημαντικό. Ένα άλλο ζήτημα κρίσιμη σημασία για την αποστολή ήταν η διαχείριση των ανθρώπινων πόρων. Αντιλαμβάνεστε πόσο σημαντικό αυτό είναι για να υπάρξει πραγματική μεταρρύθμιση στον τομέα τη ασφάλεια. Για παράδειγμα, 7.300 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας ε, που είναι το σύνολο που, που, που, που μετέχουν στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας έπρεπε να ληφθούν από αυτά βιομετρικά δεδομένα να καταγραφούν και επίσης έγινε και μια ε, διαδικασία συνεργασία με τις τοπικές αρχές για ε, υποστήριξη για, τον, για παράδειγμα για τον τρόπο με τον οποίο οι, οι μαχητές που έχουν πλέον παραδώσει τα όπλα από την προηγούμενη σύγκρουση θα μπορούσαν να συμμετάσχουν αργότερα στις ένοπλες δυνάμεις. Προσπαθήσαμε λοιπόν να δημιουργήσουμε μια ε, λειτουργική δομή στις ενόπλες δυνάμεις παρήχαμε ε, εκπαίδευση στους αξιωματικούς και τους υπαξιωματικούς, ξεκινώντας φυσικά από το επαγγελματικό προσωπικό. Όσον αφορά α, την εκπαίδευση, τη μη επιχειρησιακή, α, αυτό πρέπει να έχει ήδη ξεκινήσει. Κάποια στιγμή τον Ιούλιο έγιναν σχετικά σεμινάρια. Ζητήθηκε λοιπόν από την αποστολή ε, συγκεκριμένα να παράσχει μια επιχειρησιακή εκπαίδευση. Και αυτό ανοίγοντας την πόρτα και για μελλοντικέ συνεργασίες. Έχουμε δύο συγκεκριμένε πρωτοβουλίες λοιπόν υποστήριξη αυτή τη μία επιχειρησιακή εκπαίδευση. Πρώτον, έχει σχέση με τις εγκαταστάσεις. Ε, ε, το, το, το, τα έπιπλα, τον εξοπλισμό. Δηλαδή χρειάστηκε πραγματικά να βρούμε καρέκλες, τραπέζια, πίνακες για να δημιουργήσουμε αίθουσες τις οποίες να μπορούμε να κάνουμε τα σεμινάρια. και παρά το μικρό του κόστου, αυτό το πρόγραμμα δεν προχώρησε. Επίσης ένα άλλο ζήτημα είναι η κάλυψη των εξόδων των εκπαιδευτών που θα έρθουν από ε, την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα μεταβούν στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, στον Πάνκι, για να κάνουν την εκπαίδευση. Και αυτό μπλοκαρίστηκε. Δεν είναι κρίση. είναι ένα ζήτημα το οποίο το έχουμε ξανασυζητήσει στο πλαίσιο της, της Επιτροπής εδώ για τα ζητήματα της εκπαίδευσης, ότι ο αποδέκτης των, της εκπαίδευσης στον τομέα της το στρατιωτικό και της ασφάλειας, αυτό σημαίνει ότι μια και ο αποδέκτης είναι οι ένοπλες δυνάμεις μια χώρα, δεν είναι επιλέξιμος σύμφωνα με την αξιολόγηση της νομικής υπηρεσίας της Επιτροπής, σύμφωνα με τη συνθήκη. Είναι ένα ζήτημα το οποίο το έχουμε συζητήσει πολλές φορές, είναι μια, ένα πρόβλημα διαρκές, το οποίο δεν ε, έχει, ε, μας έχει αποτρέψει από το να ολοκληρώσουμε ή να ξεκινήσουμε καν ε, προγράμματα εκπαιδευτικής συνεργασίας. Για τα 13 προγράμματα τα οποία έχουμε εν εξελίξη θα, χρειαστούν, ε, ε, θα χρειαστεί εξοπλισμός πολιτικής προέλευσης. Μιλάμε για τραπέζια και καρέκλες. Αυτά είναι απαραίτητα για να παρέχει κανείς αυτή την εκπαίδευση. Όλες αυτές οι πρωτοβουλίες, όλα αυτά τα αιτήματα έχουν απορριφθεί. Τώρα γίνεται μια ε, προσπάθεια από κοινού από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης για να βρεθεί μια λύση Τώρα δεν θέλω να πω στα θέματα του equip, θα ήταν μια ξεχωριστή συζήτηση. Είναι δύο ξεχωριστά ζητήματα εδώ. Πρώτον, πώς θα βρεθεί τρόπος να έχουμε στη διάθεσή μας ε, τα πολύ απλά και απαραίτητα ε, εργαλεία ή εξοπλισμό που χρειαζόμαστε ε, σε μια βραχυπρόθεσμη προσπάθεια ή ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο όπως αυτά που περιέγραψα στην ε, και Αφρικανική Δημοκρατία και το δεύτερο σε μεγαλύτερο βάθος χρόνου πώς μπορούμε ε, να ξεκινήσουμε και να λειτουργήσουν αποτελεσματικά προγράμματα τέτοια εκπαιδευτικά. Τα περισσότερα από αυτά τα προγράμματα καταφέραμε να τα ξεμπλοκάρουμε ως εξής την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, αξιοποιώντας την βοήθεια και τη γενεοδορία δύο κρατών μελών, το Λουξεμβούργο, το οποίο προσέφερε 300.000 ευρώ, και η Γαλλία, η οποία προσέφερε 50.000 ευρώ. Συνολικά 450.000 λοιπόν ήταν το κόστος που χρειάστηκε για να υλοποιηθούν αυτά τα δύο προγράμματα. αλλά τουλάχιστον μπορούμε να είμαστε ευτυχείς ότι θα καταφέρουμε να επιτελέσουμε το έργο μας. Να... Αυτό που μας έχει ζητηθεί να επιτελέσουμε εξάλλου. Αλλά Ε, αυτή η κατάσταση ε, ε, μας δείχνει ότι υπάρχει ένα πρόβλημα εδώ. Δεν μπορούμε να εξαρτώμαστε από τη γενεοδορία, από την καλή θέληση κάποιου κράτους μέλους κάθε φορά. Είναι ένα δομικό πρόβλημα, ένα συστημικό πρόβλημα που θα πρέπει να λυθεί. Ζητώ συγγνώμη για αυτή τη μικρή παρένθεση. Πιστεύω όμω είναι πάρα πολύ κέριο. Γιατί πρέπει να καταλάβουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση όλο και περισσότερο εμπλέκεται στο να δίνει να ενισχύει τι ικανότητε τοπικών παικτών, τοπικών αρχών σε διάφορα μέρη του κόσμου, ιδίω στην Αφρική. Αυτό μπορεί να αποτελέσει ένα μεγάλο πρόβλημα. Δεν θέλω να κατηγορήσω κανένα αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινεί με τον εαυτό μας και δούμε τι γίνεται σε σχέση με τις δικές μας εθνικές λύσεις, αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι οι εμπλεκόμενοι στην ανάπτυξη κάνουν τα ίδια πράγματα. Αυτό που θέλω να υπογραμμίσω εδώ είναι ότι αυτό που θέλουμε να πετύχουμε σε ό,τι αφορά την σωστή και προβλέψιμη λύση είναι να δώσουμε υποστήριξη σε μη στρατιωτικό εξοπλισμό, σε στρατιωτικούς οργανισμούς και αυτό είναι κάτι περισσότερο από αυτό που μπορούν να κάνουν τα κράτη-μέλη σε εθνικό επίπεδο. Πρέπει να δούμε λοιπόν τι διαδικασίε μα σε εσωτερικό επίπεδο για να δούμε πώ θα υποστηρίξουμε αυτή τη, αυτή τη διαδικασία. Κάτι ακόμα τώρα ο αντίκτυπος της κρίσης του τέλους Σεπτεμβρίου. Τι αποτέλεσμα έχει πάνω στην δραστηριότητα της αποστολής μας. Όπως ξέρετε στο τέλος Σεπτεμβρίου, 26 με 30 Σεπτεμβρίου, με τη βοήθεια της ε, γαλλικής δύναμης μπορέσαμε να επαναφέρουμε την τάξη και τον νόμο και να σταματήσουμε τις ταραχές παραμένουν βέβαια οι εντάσεις και εξακολουθούν να υπάρχουν επεισόδια σε τακτικό επίπεδο. Είναι σημαντικό λοιπόν να επανελθεί η εμπιστοσύνη η οποία έχει υπονομευτεί και υπάρχει η υπόνοια ότι πολλοί οι οποίοι βρίσκονται σε θέσεις έχουν συμμετάσχει σε αυτές τις ταραχές. Αυτό το οποίο λοιπόν διακυβεύεται εδώ και ο στρατηγός Λοζιάλ φυσικά το έχει υπόψη του είναι πράγματα για τα οποία προσπαθούμε να βρούμε μια λύση. Πρώτα απ' όλα είναι η ανάγκη να μην συμμετάσχει ο στρατός της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας της ε, ε, ταραχές. Πάνω από 400, περίπου 400 μόνο άτομα αυτού του στρατού έχουν συμμετάσχει στις ταραχές. Το μεγαλύτερο μέρος όχι, δεν το έκανε. Το να κατηγορήσουμε συμπούρμπουλο και σύνολο αυτόν τον οργανισμό λοιπόν θα ήταν απόλυτα άδικο. Και θα ήταν και αντιπαραγωγικό εξάλλου. Χρειαζόμαστε επίσης η ΦΑΚΑ να κάνει μια εσωτερική εξυγίανση των τάξεών της. Αυτοί οι οποίοι δεν έχουν ε, διαδραματίσει σωστά το ρόλο τους και αυτοί οι οποίοι ενεπλάξαν στις ταραχές ήταν πάρα πολύ λίγοι. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει μια κάθαρση του στρατού από αυτά τα στοιχεία για να μπορέσει να επανέλθει η εμπιστοσύνη και η αξιοπιστία αυτού του φορέα. Και είναι σημαντικό επίσης να επανέλθει η η τάξη και η πειθαρχία. Όταν είναι αργή και χωρίς κανένα αντικείμενο εργασίας οι στρατιώτες, είναι πολύ πιο πιθανό ότι θα εμπλακούν σε τέτοιες ταραχές και ενόπλες δυνάμεις. Αυτό που είδαμε λοιπόν το Σεπτέμβριο πρέπει να βελτιώσουμε και να επιταχύνουμε τη διαδικασία να τους ε, εκπαιδεύσουμε και να έχουν μια καλύτερη προοπτική για το μέλλον. Να τους ξαναδώσουμε λοιπόν την αξιοπρέπεια και την εμπιστοσύνη στο έργο τους. Και πρέπει να σου κρατήσουμε το χέρι και να τους μεταμορφώσουμε. Δεν μπορούμε να πούμε ότι τελείωσε το έργο μας και μετά τους αφήνουμε και φεύγουμε και τους αφήνουμε στην τύχη τους. Αυτό δεν είναι μια σωστή αντιμετώπιση. Και τώρα για την ε, κατάσταση που θα επικρατήσει μετά από το τέλος αυτής της αποστολής. Όταν δώσουμε λοιπόν αυτές τις συμβουλές, όταν βελτιωθεί η αλυσίδα διοίκησης και τα αρμόδια υπουργεία και το προσωπικό σε στρατιωτικό επίπεδο έχουν οργανωθεί με τον κατάλληλο τρόπο, είναι πολύ σημαντικό κάποιος να εκπαιδεύσει και το προσωπικό της ΦΑΚΑ. Δεν είναι πολλοί οι εθελοντές. Το έλεγξαμε αυτό και με τις δυνάμεις των Ηνωμένων Εθνών. Δεν υπάρχει καμία ιδιαίτερη προθυμία, αλλά δεν υπάρχει και επίδογνωμοσύνη σε επίπεδο θελοντών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει την εμπειρογνωμοσύνη και έχει και την εμπειρία. Αυτά κάνουμε και στο Μαλί και στην Σομαλία και αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε και στην Κέντρο Αφρικανική Δημοκρατία. Είναι τμήμα της ε, εμπειρογνωμοσύνη που μπορούμε να δώσουμε. Δεν μπορούμε να πούμε γυρίζουμε την πλάτη μας, κάναμε ό,τι μπορούσαμε και αυτό ήταν. Όχι, έχουμε μια μεγάλη ευθύνη να παραμείνουμε και να βοηθήσουμε να δημιουργηθεί ένα ε, σύστημα το οποίο θα υποστηρίζει μια δημοκρατική χώρα και θα έχει την απαραίτητη επαγγελματικότητα. Πρέπει λοιπόν να παραμείνουμε σε όλη τη διάρκεια της ε, διαδικασίας αυτής ώστε να φτάσουμε στο σωστό αποτέλεσμα. Στις 8 Οκτωβρίου εξάλλου ο πρόεδρος της μεταβατικής κυβερνήσεως ο Σαμποπάντα Πάντσα, έστειλε μια επιστολή στον, ε, στην ύπατη εκπρόσωπο ζητώντας από την Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσει συνέχεια στην αποστολή αυτή ώστε να υπάρξει λειτουργική, μάλλον επιχειρησιακή εκπαίδευση του προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων εκεί. Ξέρουμε ότι υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις για να γίνει κάτι τέτοιο προτού ξεπεράσουμε σε μια τόσο ευρύτερη ε, ενέργεια εκπαίδευσης. Είναι πολύ σαφές ότι η πρώτη προϋπόθεση είναι να έχουμε μια εκλεγμένη κυβέρνηση η οποία θα έχει την εξουσία. Δεν μπορεί μια μεταβατική κυβέρνηση να ξεκινήσει μια τέτοια διαδικασία. Πρέπει να είναι η νέα εκλεγμένη κυβέρνηση η οποία θα έχει περάσει από τη φυσιολογική διαδικασία εκλογών. Όλε αυτέ οι δράσει λοιπόν ήδη έχουν καθυστερήσει. Προβλεπόταν για τον Οκτώβριο και τώρα τον Δεκέμβριο. Ελπίζουμε ότι μπορούν να γίνουν αυτέ οι εκλογέ ή αλλιώ στην αρχή του επόμενου χρόνου. Είναι απολύτω σαφέ ότι μια νέα κυβέρνηση δεν μπορεί να αναλάβει τα καθήκοντά της πριν από το Μάρτιο του 2016 εγκαίρως και πάλι, γιατί η εντολή της ε, αποστολής μας τρέχει μέχρι τον Ιούλιο του 2016. Ιδανικά δεν θα πρέπει να υπάρξει ένα μεγάλο χάσμα μεταξύ της τρέχουσας ε, ε, αποστολής και της νέας μας παρουσίας στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία. Είναι επίσης σαφές ότι προτού ξεκινήσουμε οποιαδήποτε επικρισιακή κατάρτιση θα πρέπει να ολοκληρωθεί όλη η διαδικασία ελέγχου της ασφαλείας. Να γνωρίζουμε δηλαδή ακριβώς ποιον εκπαιδεύουμε. Να διασφαλίσουμε ότι όντως οι άνθρωποι εκπαιδεύουμε είναι έμπιστοι άνθρωποι. Πρέπει λοιπόν και αυτή η διαδικασία της διαπίστευσης του ελέγχου να ολοκληρωθεί. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να περάσει από τη διαδικασία αυτή το σύνολο των ενόπλων δυνάμεων. Πολύ σημαντική είναι η διαδικασία SSR, η μεταρρύθμιση τομέα της άμυνας. Πρέπει να δούμε εδώ πέρα ποιος κάνει τι, ποιες θα είναι οι ευθύνες που θα έχουν από τη μια ο στρατό και από την άλλη χωροφυλακή και αστυνομία. Είναι πολύ σημαντικό να γίνει δηλαδή μια οριοθέτηση αρμοδιοτήτων και καθηκόντων, γιατί ακριβώ η ασάφεια που υφίσταται αυτή τη στιγμή προκαλεί και εντάσει. Είναι επίση πολύ σημαντικό να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία αφοπλισμού, DDR. Και βέβαια με αυτό ασχολείται κυρίω η αποστολή των Ηνωμένων Εθνών, που ασχολούνται κυρίω με τον αφοπλισμό και την επανένταξη. Πώ μπορούμε δηλαδή να επανισάγουμε στον επίσημο στρατό τους α, συμμετέχοντες αυτή τη στιγμή σε παραστρατιωτικές οργανώσεις. Να περάσουν δηλαδή άνθρωποι αυτοί από έναν έλεγχο και σιγά σιγά να ενσωματωθούν στις επίσημες ενωπές δυνάμεις της χώρας. Και επ' αυτού τον πρώτο λόγο βέβαια έχει αποστολή των Ηνωμένων Εθνών και συνεργαζόμαστε με τους συναδέλφους μας στα Ηνωμένα Έθνη προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι όντως μπορούν να έχουν και τη δική μας τη βοήθεια. Επίσης, ο προπολογισμό και ο μελλοντικός ρόλος του επίσημου στρατού, του ΦΑΚΑ, και αυτό δεν έχει ακόμα αποφασιστεί. Επίσης, ξέρετε ότι η κεντροφερκανική δημοκρατία βρίσκεται σε ένα καθεστώς κυρώσεων των ΗΕ. Δεν μπορούμε δηλαδή να φέρουμε όπλα στη χώρα αυτή. Αλλά αυτό προκαλεί πρόβλημα, γιατί αν πραγματικά θέλουμε αυτή τη στιγμή να δημιουργήσουμε ένοπλε δυνάμει οι οποίε θα μπορέσουν να επιτελέσουν το έργο του, προφανώ οι δυνάμει αυτέ χρειάζονται και αμυντικό εξοπλισμό. Λοιπόν, όσον αφορά το χρονοδιάγραμμά μα και τα μελλοντικά βήματα, τον... στι 17 Νοεμβρίου θα έχουμε το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, το οποίο θα δώσει συγκεκριμένα καθήκοντα και αρμοδιότητες προκειμένου να ξεκινήσει ο στρατηγικός σχεδιασμός προκειμένου να έχουμε μια ευρωπαϊκή αποστολή κατάρτιση στην κεντροφροκανική δημοκρατία. Την επόμενη εβδομάδα λοιπόν θα ξεκινήσει η εργασία. Αυτή τη στιγμή ληφθεί η επίσημη απόφαση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και θα εκπονήσουμε ένα έγγραφο το οποίο θα είναι έτοιμο στα τέλη Ιανουαρίου. Πράγμα το οποίο θα μας επιτρέψει στη συνέχεια να αρχίσουμε την επιτόπου κατάρτιση των στρατιωτικών έτσι ώστε να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε με τις νέες μας αυτές αρμοδιότητες προτού ολοκληρωθεί η υφιστάμενη αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η EU MAMA. Αν έχω λίγο χρόνο κύριε Πρόεδρε, να πω και συγγνώμη να έχω μακρηγορήσει, σταματήστε με αν δεν υπάρχει χρόνος. Και όχι, μετά εδώ πέρα να σας ακούσουμε. Λοιπόν, να πω κάτι ακόμα, κυρία Πρόεδρε. Κάτι που κάνουμε για πρώτη φορά και είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Αφορά τη συνεργασία μα με τα Ηνωμένα Έθνη και αναφέρομαι εδώ πέρα σε αυτά την άντληση διδαγμάτων στην οποία αναφέρθηκα στην αρχή από την όλη εμπειρία που έχουμε στην κετοφρακανική δημοκρατία. Είπα ότι έχει ολοκληρωθεί η αρχική στρατηγική επιχείρηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση, η EU4, που έθεσε ένα πολύ θετικό παράδειγμα Θέλουμε εδώ πέρα να χρησιμοποιήσουμε την επιχείρηση αυτή ως μοντέλο πρότυπο για μελλοντικές στρατιωτικές επιχειρήσεις. Αυτή τη στιγμή σε η απόφαση να θεσπιστεί η EU4 CAR. Χρειάστηκαν 79 μέρες προτού στηθεί η όλη επιχείρηση. Είχαμε παραπονεθεί πάρα πολύ εμείς για αυτό το πράγμα, αλλά για τα Ηνωμένα Έθνη η όλη διαδικασία θεωρήθηκε ιδιαίτερα ταχεία. Ξέρετε ότι στις Ηνωμένα Έθνη χρειάστηκε ένας ολόκληρος χρόνος για να στήσουν τη δική τους την επιχείρηση. Βλέπουμε λοιπόν ότι όταν υπάρχει μια συμφωνία μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν όλες οι χώρες πούν ότι όντως πρέπει να πληχθούν οι στρατιωτικές δυνάμεις για να περισσώσουμε, να διασφαλίσουμε την ασφάλεια σε ορισμένες περιοχές όπως το Μπανκί, τότε μπορούμε να κινηθούμε πάρα πολύ γρήγορα. Μπορούμε δηλαδή να θεσπίσουμε μια προπαρασκευαστική επιχείρηση μέχρι να θεσπιστεί και να αρχίσει να λειτουργεί η επίσημη επιχείρηση των ΗΠΑ Ήδη λοιπόν από τον Ιανουάριο είχαμε μια διευθυντική συντονιστική επιτροπή Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένων Εθνών που συνεδριάζει μια φορά κάθε εξάμεινο και είπαμε ότι θα πρέπει να συνεργαζόμαστε για να αντλούμε διδάγματα, να μπορούμε να ξέρουμε πώς μπορούμε να συνεργαστούμε στο μέλλον για να γεφυρώνουμε το διάστημα αυτό το οποίο υπάρχει ανάμεσα στις δύο αυτές επιχειρήσεις, να μην προκύπτουν δηλαδή κενά. Και Είπαμε επίσης ότι για το 2015 μέχρι το 2018 έχουμε πλέον ένα επίσημο πρόγραμμα εργασία για τη συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένων Εθνών. Πολλά έγγραφα έχουν συνταχθεί, πολύ σύντομα θα έχουμε και τα αποτελέσματά τους. Στις αρχές Δεκεμβρίου θα έχουμε την επόμενη συνεδρίαση της Steering Committee και φαντάζομαι ότι μέχρι τότε θα έχουμε και το σχετικό έγγραφο έτοιμο. Να αναφερθώ και σε κάτι ακόμα που ενδεχομένω να σε ενδιαφέρει. Ποια είναι τα διδάγματα αυτά τα οποία έχουμε αντλήσει από την όλη εμπειρία μα μέχρι σήμερα και πώ θα μα εμπνεύσει αυτό για τη μελλοντική μα εργασία. Το πρώτο δίδαγμα έχει να κάνει με τη γενικότερη μεθοδολογία που χρησιμοποίησαμε. Όπω γνωρίζετε, αναφερόμαστε εδώ πέρα σε ένα τρίγωνο. Έχουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Αφρικανική Ένωση και τα Ηνωμένα Έθνη. Έτσι ξεκίνησε η όλη συνεργασία. Το αρχικό μας πρόβλημα ήταν ότι όταν αρχίσαμε να σχεδιάζουμε και να προγραμματίζουμε τη δράση μας από ευρωπαϊκής πλευράς, δεν γνωρίζαμε εκείνη τη στιγμή ότι θα έπρεπε να υποστηρίξουμε ή να γεφυρώσουμε, αν θέλετε, το επιχειρησιακό αυτό χάσμα που είχε προκύψει μέχρι να αρχίσει να λειτουργεί η επιχείρηση της, Ευρωπα... της Αφρικανικής Ένωσης ή της... των Ηνωμένων Εθνών. Αρχικά είχαμε πει ότι θα σχεδιάζαμε τη δική μας τη δράση σε σχέση με την ΜΙΣΚΑ, που ήταν η πρώτη επιχείρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προτού ξεκινήσει η EU MAMA. Ήταν πολύ σημαντικό λοιπόν να αρχίσουμε να εργαζόμαστε από πολύ νωρί και να είμαστε σε θέση να συντονιζόμαστε με τους άλλους εταίρους από τα πρώτα προπαρασκευαστικά στάδια, προκειμένου να καταφέρουμε να αποφεληθούμε από όλες τις πιθανές συνέργειες. Αυτό ακριβώς το πλαίσιο νομίζω ότι ε, θα πρέπει να ακολουθήσουμε και σε άλλες τέτοιες περιστάσεις που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε στην Αφρική. Να αρχίσουμε δηλαδή να συνεργαζόμαστε και στις υπόλοιπες περιοχές Αφρικής όπου έχουμε στρατιωτική παρουσία με τα Ηνωμένα Έθνη ακολουθώντα αυτή τη μεθοδολογία. Το ίδιο ισχύει και για τη συνεργασία μα με την Αφρικανική Ένωση. Ξέρετε ότι εκατομμύρια και δισεκατομμύρια έχουμε δαπανίσει προκειμένου να δημιουργηθεί το μέσο αυτό ειρήνευση στην Αφρική, το African Peace Facility Capacity. Θέλουμε λοιπόν να συνεχίσουμε και στο μέλλον να εργαζόμαστε σε αυτό το πλαίσιο, να ακολουθήσουμε αυτή τη διάρθρωση, να είμαστε σε άμεσο συντονισμό και με την Ηνωμένα Έθνη και με την Αφρικανική Ένωση. Και ένα άλλο ζήτημα τακτική φύσεω, η ανταλλαγή πληροφοριών. Ξέρετε ότι ε, δεν έχουμε τη δυνατότητα να δίνουμε στου συναδέλφου από Ηνωμένα Έθνη απόρριτε πληροφορίε Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε στη φάση του σχεδιασμού, ούτε στη φάση τη εκτέλεση. Καταλαβαίνετε ότι όμως αυτό μας προκαλεί πολλά προβλήματα. Αν δούμε την επιχείρησή μας, την EU-MAM και αναφέρομαι στα 60 άτομα τα οποία εργάζονται στα πλαίσια της επιχείρησης αυτής, τα οποία είναι τοποθετημένα σε ένα κτίριο το οποίο έχει ε, δημιουργηθεί με τη συνεργασία των Ηνωμένων Εθνών. Αν οι άνθρωποι λοιπόν αυτοί δεν μπορούν να διαβιβάζουν απόρριτες πληροφορίες, τότε τίθεται ένα σημαντικότατο ζήτημα ασφάλειας Πρέπει λοιπόν να επιληθεί το πρόβλημα αυτό. Και ξέρετε ότι αυτό δυσχεραίνει επίσης και οποιαδήποτε απόπειρα γίνεται για συνεργασία, για σχεδιασμό από κοινού ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Ηνωμένα Έθνη. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να δούμε τι θα κάνουμε με το ζήτημα αυτό, γιατί πολύ φοβάμαι θα το αντιμετωπίσουμε και σε άλλα θέατρα επιχειρήσεων. Ουσιαστικά, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης EU4 είχαμε εθνικές συνιστώσεις, εθνικές ομάδες δηλαδή στρατιωτών που α, ε, πολλές φορές τα Ηνωμένα Έθνη του ζητούσαν να παραμείνουν στην κεντροφρακανική δημοκρατία προκειμένου να συνεχίσουν την εργασία που κάνανε και στα πλαίσια της UN Minusca. Προφανώς δεν μπόρεσε όμως να γίνει τίποτα τέτοιο τα Ηνωμένα Έθνη θέλουν να χρησιμοποιήσουν για παράδειγμα τις ειδικέ δυνάμεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενδιαφέρει ιδιαίτερα να χρησιμοποιήσουν τις δυνάμεις της χωροφυλακής. Για πρώτη φορά εμείς είχαμε δυνάμεις της χωροφυλακής στα πλαίσια της στρατιωτικής μας αυτής επιχείρησης και οι άνθρωποι, οι συνάδελφοί μας από Ηνωμένα Έθνη θέλουν να κρατήσουν αυτές τις μονάδες χωροφυλακής επιτόπου προκειμένου να συνεχίσουν εκεί πέρα το πολύ θετικό του έργο. Δεν καταφέραμε όμως αυτό για διοικητικούς λόγους να το κάνουμε. καταφέραμε μόνο να συνάψουμε κάποιε συμφωνίε διοικητική φύση με τον ΕΕ ποιο θα αναλάβει τη μίσο του κτηρίου αφού εμεί αποχωρήσουμε κ.ο.κ. Νομίζω θα πρέπει όμω να έχουμε συνεργασία και για στρατιωτικά ζητήματα, όχι μόνο για διοικητικά. Και να αναφερθώ και σε κάτι ακόμα. Στη Γεωργία. Η Γεωργία είναι χώρα εταίρο η οποία διαδραμάτισε ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην στελέχωση τη όλη επιχείρηση και αναφέρομαι και στην EU-CAR και στην υφιστάμενη EU-MAMA. Μάλιστα, 169 στρατιώτες από τους συνολικά 850 που χρησιμοποίησαμε προέρχονταν από τη Γεωργία στα πλαίσια της EU4 CAR. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό συμβολή. Καταλαβαίνετε ότι συμμετείχαν προφανώς και άλλες χώρες όπως η Γαλλία και άλλες που υποστήριξαν χρηματικά την Γεωργία αλλά μην ξεχνάμε ότι η Γεωργία έστειλε πραγματικά στρατιώτες επιτόπου και συνέβαλαν κατά αυτόν τον τρόπο με προσωπικό, με εξοπλισμό στην κυτοφροκανική δημοκρατία. Αν δούμε και την επιχείρηση ISF, θα δούμε πάλι εκεί ότι ε, η συμβολή της ε, Γεωργίας ε, ήταν πάρα πολύ σημαντική. 1.600 άτομα είχαν συμμετάσχει στην επιχείρηση αυτή και μάλιστα κάναν και την πιο δύσκολη δουλειά εκεί πέρα. Δεν κάνανε διοικητική δουλειά σε κάποια γραφεία, αλλά πραγματικά επιτελούσαν την πιο δύσκολη στρατιωτική εργασία. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο του συμπεριλάβαμε και αυτούς ε, σε αυτή την αποτίμηση ε, άντλησης διδαγμάτων. Έτσι λοιπόν αυτή τη στιγμή δεν αναφερόμαστε μόνο στην εργασία που είχαμε με την Αφρικανική Ένωση ή την ΕΕ, αλλά αναφερόμαστε ρητά και στην πολύ θετική συνεργασία που είχαμε με τη Γεωργία. Ακούστηκαν κάποιες επικρίσεις αλλά εν γέννη εμεί είπαμε ότι ήταν πάρα πολύ σημαντικό το ότι ήδη από την αρχή όταν ξεκίνησαν οι επιχειρήσεις αυτές το 2003 και ξέρετε ότι είχαμε συνολικά 34 επιχειρήσεις στα πλαίσια της κοινή πολιτικής άμυνας και ασφάλειας, πάντα είχαμε και εταίρους. Είχαμε δηλαδή και τρίτε χώρε οι οποίε συμμετείχαν. Είναι πολύ σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ποιε είναι οι δυσκολίε των χωρών αυτών κάθε φορά που θέλουν να συμμετέχουν, να συμμετέχουν σε τέτοιε επιχειρήσει. Θα σταματήσω εδώ πέρα. Δυστυχώς έχω να πω και πολλά ακόμα, αλλά δεν προφθαίνω. Ευχαριστώ. Η επόμενη, το επόμενο θέμα σημερινής διάταξης είναι η δημόσια κρόαση για τη συνεργασία με άλλους φορείς και χώρες. Είναι πολύ καλή η παρουσίασή σας, είναι μια εισαγωγή σε αυτή την ακρόαση και πρωτού δώσω το λόγο στα μέλη. Θα ήθελα και εγώ να πω μερικά σχόλια για το θέμα αυτό. στις αρχές του 2015 ήταν η αποστολή μας στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία ήταν ουσιαστικά η τελική φάση της ε, δράσης της ε, επιχείρησής μας στο Μπαγκί και όλοι οι συνομιλητές μας ανέφεραν την θαυμάσια απόδοση της γεφυρωτικής αυτής αποστολής και τα μόνα σχόλια τα οποία έγιναν είναι ότι υπήρξαν κάποιες αμφιβολίες αν ήταν η σωστή χρονική στιγμή για να δοθεί η σκητάλη στη Μινούσκα. Και εγώ η ίδια είχα αμφιβολίες Όλα αυτά λοιπόν είναι μια διαδικασία μαθησιακού χαρακτήρα. Πρέπει να σκεφτούμε καλύτερα για το πιο μακροπρόθεσμο επίπεδο και αυτά αναφέρθηκαν και από τον διοικητή της ε, δύναμης χωροφυλακής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και μιλώντας με τους ε, συμμετέχοντες, τους στρατιώτες, της ε, δύναμης της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορώ να πω ότι ήταν πολύ πεπειραμένοι περισσότεροι από αυτούς, είχαν ε, ήδη συμμετάσχει σε αποστολές στο Αφγανιστάν. Ήταν διαθέσιμοι να παρέμβουν και να αναλάβουν τα καθήκοντά τους, όσο δύσκολη ήταν και αυτή η στιγμή, δεν εφοβούντο να βρεθούν στο, στην καρδιά των τεκτενομένων και να αντιμετωπίσουν τους αντιπάλους τους και συνέβαλαν ιδιαίτερα στο να υπάρξει η σωστή λειτουργία της αποστολής με την εντολή της Μινούσκα. Μετά από την έκρηξη των ταραχών έγιναν πολλά γεγονότα τα οποία ήταν ιδιαίτερα ατυχή και οδήγησαν στην ε, παρέτηση του πρεσβευτού Γκαϊέρ και τελικά ήταν απόφαση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ να αποδεχθεί την ε, παρέτηση αυτή. Ελπίζουμε λοιπόν να ξαναβρούμε την ε, ε, όθηση που απαιτείται για τα θέματα αυτά, αλλά αυτή η μεταφορά εξουσιών δεν ήταν ιδιαίτερα επιτυχής, τουλάχιστον να το πω έτσι. Η Μινούσκα δεν ήταν τόσο έτοιμη να παίξει το ρόλο της και ήταν πολύ δύσκολη στιγμή και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να ανακτήσουμε την όρμη που χρειάζεται. Κύριε Γκόμις, θέλετε να πείτε κάτι. Ε, όχι, Κύριε Κέλαμ, συγγνώμη, να δώσουμε πρώτα το λόγο στην κυρία Γκόμες. Ευχαριστώ. Θέλω ευχαριστώ κύριο Κλόντι για την τόσο ενδιαφέρουσα αυτή ενημέρωση. Ήταν μια ενδιαφέρουσα και πολύ επικοδομητική εμπειρία σε δύσκολες συνθήκες. Ναι, πράγματι έχουμε μια υποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία. Ξέρουμε ότι κάποια κράτη-μέλη παίζουν ένα πιο σημαντικό ρόλο εκεί. Υπάρχει μια έλλειψη λοιπόν αναλογίας και αυτό δυσκολεύει τα πράγματα. Τουλάχιστον υπάρχει αυτή η παρουσία. Εγώ εντυπωσιάστηκα από τις δυσκολίες που αντιμετωπίσατε και ελπίζω ότι θα μπορέσετε να ξεπεράσετε αυτές τις παράλογες νομικές αντιρρήσεις για την παροχή απαραίτητου εξοπλισμού. Μπορώ να φανταστώ λοιπόν ότι αυτή είναι μια ενδιαφέρουσα περίπτωση και για τον ΟΗΕ και ξέρω γιατί αυτή η περίπτωση μπορεί να αποτελέσει ένα παράδειγμα, ένα υπόδειγμα. Υπάρχουν βέβαια όλες αυτές οι πολύ σημαντικές προϋποθέσεις που αναφέρατε, ώστε να μπορέσουμε πράγματι να προχωρήσουμε προς μία πιο σημαντική κατεύθυνση. Για μένα η επιστολή αυτή που αναφέρεται, που ζητά να εκπαιδεύσουμε τους μελλοντικούς ε, Στρατιώτε της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας είναι πολύ σημαντική, αλλά χρειάζεται να υπάρχει το κατάλληλο πολιτικό πλαίσιο ώστε να γίνει πραγματικότητα. Αλλά όταν υπάρχουν αυτές τις προϋποθέσεις θα πρέπει να το πράξουμε. Και το ερώτημα προς εσάς είναι το εξή. Μήπως αυτό θα μπορούσε να γίνει ένα υπόδειγμα όχι μόνο για την Αφρική και τις αφρικανικές χώρες, αλλά και για μας τους ιδίους εν ώψη του παρελθόντος κάποια μέρα θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε καθήκοντα που δεν μπορούμε να τα απαρνηθούμε και η άρνησή μας για το θέμα αυτό ήταν ένας από τους λόγους που έφτασε η κατάσταση στη Λιβύη εκεί που έφτασε. Σε κάποιο σημείο θα πρέπει να κάνουμε αυτά τα απαραίτητα στη Λιβύη δεν μπορούν να γίνουν αυτά καθόλου χωρίς ευρωπαϊκή συμμετοχή και δέσμευση. Και το ερώτημά μου είναι, σε, κάποιο, σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι αυτό μπορεί να αποτελέσει ένα θετικό υπόδειγμα για τις διαφορετικές χώρες. Γιατί πολλά από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στην κεντροαφρικανική δημοκρατία έχουν μεγάλη σχέση με το μπάχαλο το οποίο δημιουργήθηκε στην Λιβύη και τα μηνύματα που προέκυψαν από εκεί. Ευχαριστώ, λέει πρώτος, κύριε Κέλλαμ. Σας ευχαριστώ για την τόσο καλά παρουσιασμένη θέση σας. Εγώ συμφωνώ με την προλαλή σας, κύριε Γκάμις, ότι το παράδειγμα της κεντροαφρικανικής δημοκρατίας θα μπορούσε να μεταλαμβαδευτεί και σε άλλες περιπτώσεις. Το ερώτημα παραμένει γιατί δεν έχει σταθεροποιηθεί ακόμα η κατάσταση. Η χώρα αυτή είναι σχετικά μικρή. Λιγότερα από 5 εκατομμύρια είναι κάτι το διαχειρίσιμο. Υπάρχει το πρόβλημα αυτό εδώ και πολύ καιρό. Υπάρχει βοήθεια που δίνεται στις εθνικές δυνάμεις. Υπάρχει υποστήριξη των προσφύγων και σε γειτονικέ χώρες, ειδικά προγράμματα για τα παιδιά και παρόλα αυτά ο μισός πληθυσμός χρειάζεται βοήθεια για να αντιμετωπιστεί η βία, ιδίως η βία που προέκυψε μετά το Σεπτέμβριο, η οποία ήταν πολύ ανησυχητική, δεν υπάρχει ακόμα προοπτική εκλογών. Με την εκτιθής από εσά λοιπόν εμπειρία, το ερώτημά μου είναι το εξή. Κατά τη δική σας άποψη, η βάση της δικής σας εμπειρίας, ποιο θα έπρεπε να είναι το σημαντικό στοιχείο για να αντιμετωπιστεί την αστάθεια. Μήπως υπάρχουν και εξωτερικοί συντελεστές που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Πώς αξιολογείτε εσείς την κατάσταση εκεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Έχετε το λόγο λοιπόν για να απαντήσετε. Ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις σας, ευχαριστώ πολύ και για τις παρατηρήσεις. Κοιτάξτε, όσον αφορά την επιστολή αυτή, δεν νομίζω ότι είμαι πλέον αρμόδιος για να σας απαντήσω. Ενδεχομένως οι αρμόδιοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ασχολούνται με την κεντροφρακανική δημοκρατία θα έπρεπε να σας δώσουν τις απαντήσεις αυτές. Εγώ θα ήμουν αρκετά υποκειμενικό στην τοποθέτησή μου. Όσον αφορά τώρα την χρηματοδότηση για την αγορά εξοπλισμού, να ξεκινήσω πρώτα με αυτό. Κοιτάξτε, είναι πολύ σημαντικό το ζήτημα αυτό και όντως θα πρέπει να επιληθεί. Κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μας επιτρέψει τελικά να σχεδιάσουμε και να εφαρμόσουμε επιτόπου τα καθήκοντα που έχουμε στη χώρα αυτή, για το σχεδιασμό δηλαδή εξοπλισμών. Προφανώς δεν μπορούμε τον αμυντικό κλάδο να τον αφήσουμε εκτός όλης αυτής προσπάθειας που γίνεται. Αν ο στόχος μας είναι να οικοδομήσουμε κράτη τα οποία θα λειτουργούν σωστά στην ε, Αφρική ή οπουδήποτε αλλού, προφανώς θα πρέπει να δίνουμε τη δυνατότητα στις τοπικές αρχές να έχουν συγκεκριμένε ικανότητες στους κέριους τομείς και ένας από αυτούς είναι και η άμενα. Αν φύσετε εκτός την άμυνα από τις προτεραιότητές σας, τότε προφανώς η χώρα μπορεί να καταρρεύσει, δεν θα μπορέσει να λειτουργήσει και ως αποτέλεσμα όλες οι υπόλοιπες επενδύσεις που θα έχετε κάνει στον υγειονομικό τομέα, στις υποδομές, στην παιδεία και αυτές θα καταρρεύσουν. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό να θεραπεύσουμε αυτό το πρόβλημα. Επίσης, βλέπω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταβάλει σημαντικές προσπάθειες προκειμένου να γίνουν αυτές οι επενδύσεις και ακόμα και αν είχαμε κάποια προβλήματα και σας εξέθεσα με απόλυτη ειλικρίνεια το πρόβλημα. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να πω ότι οι εθνικές πρακτικές δεν διαφέρουν πάρα πολύ. Εμείς ουσιαστικά περιμένουμε και από όλους αυτούς οι οποίοι φέρουν μια συγκεκριμένη ευθύνη όσον αφορά την χρηματοδότηση των προγραμμάτων που θέλουμε να εφαρμόσουμε στην κοινωνική δημοκρατία, θα πρέπει και αυτοί σε εθνικό επίπεδο να αλλάξουν τη στάση τους. Νομίζω ότι και αυτή είναι πολύ σημαντική πρόκληση και ως προς αυτό καταβάλλονται σημαντικές προσπάθειες. Αν δούμε για παράδειγμα την επιστολή προθέσεων του Προέδρου Γιούνκερ. Εκεί πέρα φαίνεται ξεκάθαρα ότι θέλει και αυτός να επιληθεί αυτό το πρόβλημα. Αναφέρεται και σε αυτό στα πλαίσια του προγράμματος εργασίας Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα επόμενα χρόνια. Τα πράγματα δεν είναι όσο απεσιόδοξο ενδεχομένω τα παρουσίασα στην αρχή. Προφανώ υπάρχουν και θετικά στοιχεία, προφανώ γίνονται θετικέ προσπάθειε, αλλά χρειαζόμαστε και τη δική σα τη συμβολή. Όσον αφορά τώρα το πρότυπο το οποίο ακολουθούν, μάλλον το αν θα μπορούσε η δική μα επιχείρηση να πούμε για τα Ηνωμένα Έθνη. Ναι, αυτό όντω ισχύει αυτή τη στιγμή. Δεν λέμε εμεί όμω ότι θα κάνουμε οτιδήποτε για να υποστηρίξουμε τα Ηνωμένα Έθνη, ούτε θα πρέπει αυτόματα να θεωρείται κάθε φορά που τα Ηνωμένα Έθνη θέλουν να κάνουν μια επιχείρηση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτόματα άμεσα θα πρέπει να στέλνει μια τέτοια γεφυρωτική επιχείρηση προκειμένου να καλύψουμε το κενό το οποίο προκύπτει μέχρι να αρχίσει να λειτουργεί επίσημα οι επιχείρηση των ΗΕ. Πάντα κατά περίπτωση θα λαμβάνονται αποφάσεις αυτές, αν και πότε θα βοηθούμε τα Ηνωμένα Έθνη και τα κράτη-μέλη θα το αποφασίζουν αυτό. Πιστεύω πάντως ότι θα πρέπει να θεσπιστεί ένα πρότυπο εργασίας, έτσι ώστε αν εγκριθεί μια τέτοια συνεργασία να μπορεί να ελοποιηθεί επιτόπου γρήγορα και άμεσα. Και ως προς αυτό λοιπόν πρέπει να κάνουμε σημαντική δουλειά. όσον αφορά τη Λιβύη στην οποία αναφερθήκατε και όσον αφορά τη μεταρρύθμιση τομέα άμυνας στη Λιβύη. Και αυτό μας έχει απασχολήσει ήδη από σήμερα και σχεδιάζουμε να κάνουμε κάτι τέτοιο. Βέβαια πρέπει να πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις, ίσονο σημασία ενδεχομένως, το ότι θα πρέπει να έχουμε επιτόπου ένα GNA το οποίο θα μας εκπροσωπεί πραγματικά. Ορισμένοι μπορεί να το ονομάσουν αυτό το Brook Scene, μη πείτε το όπως θέλετε. Πάντως είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει μια γενικότερη υποστήριξη από το κοινό για μια τέτοια επιχείρηση. Θα πρέπει επίσης να μας προσκαλέσει Λιβύη και να μας ζητήσει να στήσουμε μια τέτοια επιχείρηση. Αυτό δεν είναι δεδομένο αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή οι διάφορες παρατάξεις που έχουν την εξουσία στη Λιβύη από κοινού λένε ότι δεν θέλουν ξένη στρατιωτική παρουσία στη χώρα. Αν μας δοθεί όμως η άδεια να επέμβουμε στη χώρα και αυτή τη στιγμή ε, έχουμε ένα συγκεκριμένο σχέδιο στρατιωτικής επιχείρησης, θα πρέπει σε συνεργασία με την πολιτική και στρατιωτική επιχείρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δημιουργήσουμε μια τέτοια επιχείρηση η οποία θα έχει ως στόχο να εξετάσει τις ε, ανάγκες της Λιβύης και να δούμε επίσης τι υποστήριξη μπορούμε εμείς να τους δώσουμε και τι υποστήριξη μπορούμε να πάρουμε από αυτούς. Μόνο κατά αυτόν τον τρόπο μπορούμε να προχωρήσουμε και αυτό μπορούμε να κάνουμε σε ένα πρώτο στάδιο. Καταρχάς πρέπει να δούμε αν μας θέλουν, αν ενδιαφέρονται για την δική μας παροχή βοήθειας. Ασχολούμεθα πάντω με το ζήτημα της Λιβύης και θα πω και κάτι ακόμη. Μία βασική ανησυχία μας είναι πώς θα καταφέρουμε να περιορίσουμε τον ιό, αν θέλετε, το έτσι, του Ισλαμικού κράτους, να μην απλωθεί περισσότερο. Θεωρώ αυτή τη στιγμή ότι είναι ένα πραγματικό θαύμα το ότι ο Λίβανος λειτουργεί αυτή τη στιγμή φυσιολογικά σαν χώρα και δεν έχει ακόμα υποπέσει αν θέλετε στον ιό αυτό του Ισλαμικού κράτους. Στόχος μας λοιπόν είναι να βοηθήσουμε χώρες σαν το Λίβανο, να καταφέρουμε να δημιουργήσουμε τις απαραίτητες ικανότητες, ενδεχομένω να δώσουμε και χρηματοδότηση. Η Ορδανία μας λέει πολλές φορές ότι πρέπει να χτίσω περισσότερες υποδομές, έχουν καταφτάσει σε μένα πάρα πολλοί πρόσφυγες. Χρειάζομαι τη δική, δική σας την χρηματοοικονομική υποστήριξη. Πολλές φορές λοιπόν η υποστήριξη είναι καθαρά οικονομική, άλλες φορές όμως έχει να κάνει και με τη δημιουργία ικανοτήτων, με τη δημιουργία ε, ενός αστυνομικού τμήμα, ε, αστυνομικών δυνάμεων, δυνάμεων της χωροφυλακής. Κατά αυτόν τον τρόπο μπορεί να προβληθεί πολύ περισσότερο και η δραστηριότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό. Προφανώς πρέπει να δούμε και το θέμα των πόρων. Και αυτό μας απασχολεί. και πρέπει να δούμε και την ετοιμότητα των κρατών μελών εφόσον υπάρχει για να προσφέρουν στρατιώτες, να προσφέρουν άτομα τα οποία θα μπορούσαν να ασχοληθούν με την κατάρτιση. Αυτή τη στιγμή σας είπα ότι στην Συμβουλευτική Στρατηγική Αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην EUMAM, έχουμε 60 άτομα. Σε άλλες αποστολές έχουμε πολύ λιγότερα. Και πάλι θα πρέπει να ευχαριστήσουμε και τους Γεωργιανούς οι οποίοι μας στείλανε το προσωπικό το οποίο μας στείλανε και πέντε επιπλέον άτομα για την επιχείρηση αυτή. Σαφώς λοιπόν θα πρέπει να συντονίσουμε την ετοιμότητα που υπάρχει στα κράτη-μέλη και θα πρέπει να έχουμε την απαραίτητη φιλοδοξία προκειμένου να υποστηρίξουμε τεχνικά και οικονομικά όλες αυτές τις επιχειρήσεις και τις ανάγκες διαφόρων κρατών. Και Νομίζω ότι ε, οι συνάδελφοί μου που είναι πιο ειδήμονες στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα είναι σε θέση να σας πούνε περισσότερο τι πρέπει να γίνει προκειμένου να παραμείνει ενωμένη η κεντροφρικανική δημοκρατία και να καταλήξει να γίνει ένα βιώσιμο κράτος το οποίο δεν θα πλήττεται από συνεχείς συγκρούσεις. Εν γέννη πάντως, και μπορώ να σας πω κάποια πράγματα εφόσον πέρασε και την προηγούμενη εβδομάδα στη Σομαλία, μας απασχολεί πραγματικά το ζήτημα αυτό. Πώς μπορούμε χώρες οι οποίες φαίνονται να είναι δημιουργημένες με έναν τρόπο κάπως αυθαίρετο και τεχνητό, χώρες οι οποίες ε, πλήττονται από το ότι υπάρχουν πάρα πολλές διαφορετικές φράξεις ή ομάδες που αντιμάχονται μία την άλλη, πώς μπορούμε να ενισχύσουμε τις χώρες αυτές για να γίνουν πραγματικά κράτη και πώς μπορούμε μάλιστα να έχουμε και την απαραίτητη περιφερειακή συνεργασία προκειμένου να υπάρχει και από τι όμορε χώρες μια υποστήριξη προς τις χώρες αυτές προσπαθούν σιγά σιγά να σταθούν στα πόδια τους χρειάζεται μια συνεχής υποστήριξη σίγουρα και κάθε φορά που συζητάμε το ζήτημα της μετανάστευσης και φαντάζομαι ότι το συζητάτε κάθε μέρα πλέον στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το ζήτημα της ασφάλειας πάλι βρίσκεται στο κέντρο και του προσφυγικού και μετανευστικού ζητήματος και αναφέρομαι βέβαια και στις χώρες καταγωγής και στις χώρες διέλευσης και πρέπει να δούμε επίσης και ποιες είναι οι συνθήκες διαβίωσης όλων των προσφύγων. Όλα αυτά στοιχίζουν, σίγουρα στοιχίζουν, αλλά πραγματικά αξίζουν την προσπάθεια γιατί Υπάρχει κάποια άλλη εναλλακτική. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε και εμείς από την πλευρά μας για αυτή την εξαιρετικά ε, διεξοδική ανάλυση της κατάστασης και την παρουσίαση που μας κάνατε. Να σας ενημερώσω ότι η γραμματεία μας έχει ήδη ξεκινήσει να, ε, να προσπαθεί να καλέσει τον διοικητή της ε, EUMAM ε, να μιλήσει στην Επιτροπή μας κάποια στιγμή τη διάρκεια του 2016. Επομένω θα μπορέσουμε να ξεδάσουμε το ζήτημα ακόμη περισσότερο βάθους. βάθος. σε ευχαριστούμε. <laughs> Please stay. We have uh, next point of our agenda. Θα περάσουμε στο επόμενο σημείο της μερίσης διάταξής μας, που είναι μια δημόσια ακρόαση σε σχέση με την συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς και τρίτες χώρες στον τομέα της ε, κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας. Έχουμε τρεις ομιλητές. Ένας από αυτούς δυστυχώς έχει καθυστερήσει με τον έλεγχο ασφαλείας στην είσοδο του Κοινοβουλίου, αλλά ελπίζουμε ότι θα έρθει και αυτό σύντομα. Ladies Κυρίες και κύριοι, καθίστε παρακαλώ. Θα παρουσιάσω τη δημόσια ακρόαση την οποία διοργανώνουμε σήμερα για το θέμα της συνεργασίας με ε, διεθνείς οργανισμούς και τρίτες χώρες στον τομέα της κοινής πολιτικής, ε, εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής άμυνας. Έχουμε μαζί μας την κυρία Κλάρα Κάνσλαντ από την Υπηρεσία Εξωτερικής ε, υπεύθυνη για τον τομέα CSDP. Όσον αφορά τη συνεργασία με τρίτες χώρες και στρατιωτικό ε, ακόλουθο της ε, εκπροσώπησης μας στο Μαρόκο ο κύριος Αλαμαντίν, εάν ακούσουμε σωστά. Ο εκπρόσωπος του Γραφείου ε, Διασύνδεσης των Οργανισμών Ηνωμένων Εθνών με την Ευρωπαϊκή Ένωση Και τέλος, ο καθηγητής Κόψ, κοσμήτορας του Κολεγίου Βερσάλιους στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο των Βρυξελών. Νομίζω ότι με αυτούς τους ομιλητές θα έχουμε μια εξαιρετική εισαγωγή στο, μια ε, εξαιρετική συζήτηση για το ζήτημα αυτό. Η παρουσίαση του κύριου Ικλόντι σίγουρα ήταν μια πολύ καλή εισαγωγή στο θέμα αυτό. Έδωσε μία από τις πτυχές της ε, συνεργασίας και χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση θα δώσω το λόγο στην κυρία Κλάρα Κάρσπλαντ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση θα μιλήσω σήμερα λοιπόν για την συνεργασία με ε, τρίτους ε, στον τομέα της κοινή εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας. Αυτό είναι ένα στοιχείο ε, ουσιώδες και αλληλένδετο, γιατί γνωρίζουμε ότι κανείς δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις μόνος του, ιδίως όταν οι πόροι είναι περιορισμένοι. Γι' αυτό πρέπει να συνεργαζόμαστε Οποτεδήποτε συνεργαζόμαστε με κάποιον τρίτο ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αξιοποιούμε την ειδική του γνώση, την εμπειρία του, αλλά επίσης μας ε, βοηθάει να δημιουργούμε και σχέσεις με φορείς, με χώρες, με οργανισμούς και να τους φέρνει πιο κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάτι το οποίο επίσης αυξάνει και την νομιμοποίηση της ε, δράσης. Δεν λαμβάνεται μωρέως από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά στη συνεργασία με άλλους φορείς, άλλους οργανισμούς διεθνώς. Επιθυμούμε να ε, ενισχύσουμε τις συνεργασίες, ε, ιδιαίτερα με τον ΟΗΕ, με την Αφρικανική Ένωση, με τον ΝΑΤΟ και με τον ΟΣΑ. ΟΣΑ έχει ήδη ε, τονιστεί λοιπόν η σημασία που έχουν οι συνεργασίες αυτές στην πολιτική μας ε. η οποία δομείται γύρω από τους εξής πυλώνες. Πρώτον, η σχέση μας με περιφερειακά και διεθνή φόρα. Εδώ εμπίπτει η συνεργασία μας με τον ΟΑΣΕ, με την Αφρικανική Ένωση, με τον ΝΑΤΟ, με τον ΟΗΕ. Δεύτερος πυλώνας είναι η συμμετοχή τρίτων χωρών σε αποστολές μας και σε επιχειρήσεις μας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης δηλαδή. Τρίτος πυλώνας, εξίσου σημαντικός, είναι ο διάλογος για την ασφάλεια και την άμυνα που αναπτύσσουμε με άλλους και τέταρτος πυλώνας είναι η συνεργασία με τρίτους προκειμένου να βελτιωθούν οι δικές τους ικανότητες. Θα ξεκινήσω από τον πρώτο πυλώνα που ανέφερα. Την συνεργασία με το ΝΟΙΕ, με το ΝΑΤΟ, με την Αφρικανική Ένωση και τον ΑΣΕ. Όσον αφορά τα Ηνωμένα Έθνη, η συνεργασία με το ΝΟΙΕ είναι προφανώς ε, εξαιρετικά σημαντική για ε, οποιοδήποτε ε, επίπεδο, για οποιοδήποτε πολιτική. Στα αριστερά μου βρίσκεται ο συνάδελφος από το ΝΟΙΕ, επομένως εκείνος θα δώσει περισσότερο θέμα. Αυτό εγώ από την πλευρά μου θα ήθελα να τονίσω την σημασία που έχει αυτή η συνεργασία είτε είναι σε πολιτικό επίπεδο, είτε είναι σε επιχειρησιακό επίπεδο, είτε σε αποστολές επιτόπου. Η διμερής συνεργασία Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΟΗΕ έχει ενισχυθεί πολύ τα τελευταία χρόνια. Θα έλεγα ότι έχει γίνει πλέον τρόπο ζωής, έχει γίνει κάτι το σύνηθες έχουμε κοινέ αξίες και αρχές με τον Οϊέ και από πλευράς ε, ΚΕΠΑ θα μπορούσε κανείς να αναφερθεί στη συνεργασία στο Μαλί, στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία ως πολύ καλά παραδείγματα μιας συνεργασίας που λειτουργεί. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η παράδοση ε, από την Μινούσκα την, ε, δηλαδή την αποστολή του ΙΕΣ την αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κέντρο Φυσικανική Δημοκρατία. Προωθείται ε, μία ε, συμφωνία πλαίσιο για την συνεργασία των αποστολών αφενός και αφετέρου μία συμφωνία για την ανταλλαγή διαβαθμισμένων πληροφοριών. Δύο εργαλεία πολύ σημαντικά για να εμπεδοθεί και να εμβαθυνθεί αυτή η συνεργασία. Επίσης είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι εφαρμόστηκε με επιτυχία το σχεδιο δραση δράσης 2012-2014 για την υποστήριξη των ερευνευτικών αποστολών του ΕΕ και τώρα ξεκινάμε μια νέα στρατηγική συνεργασία την οποία κατέπτυσαν από κοινού η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο ΕΕ που εκείνα από το 2015 με 7 περιοχές προτεραιότητες στις οποίες θα εστιάσουμε έως το 2018. Οι προτεραιότητες αυτές είναι εξής, η άμεση ανταπόκριση, η υποστήριξη των ερευνητικών διαδικασιών στην Αφρική, η διευκόλυνση της συμμετοχής των ευρωπαϊκών κρατών σε αποστολές στο ΙΕ, μεταρρύθμιση του, ε, ασφάλειας, ε, από κοινού υποστήριξη και ανταλλαγή πληροφοριών κάθε έξι μήνες ε, χάρη στο ομάδα EU Steering Committee ε, για τη συνεργασία μεταξύ ΟΗ και ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε πληροφορίες από την ΟΗΕ και σύντομα θα συναντηθούν εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Γενικού Γραμματέα για να συζητήσουν περισσότερο συνεργασία. Συμμετείχε η Ευρωπαϊκή Ένωση στις 28 Σεπτεμβρίου στην ε, Σύνοδο Κορυφής για ζητήματα ερνευτικών αποστολών του ΙΕ που οργάνωσε ο πρόεδρος Ομπάμπα. Τώρα περνώ στη συνεργασία με το ΝΑΤΟ, όπου φυσικά ε, εδώ ε, επηρεάζεται σημαντικά από τον τρόπο με τον οποίο μεταβάλλεται το περιβάλλον ασφάλειας και στην, στην περιοχή της Ευρώπης. Εδώ εστιάζουμε στο να παρέχουμε συγκεκριμένες στρατιωτικές ικανότητες ε, και να τις παρέχουμε αυτές στο, στο ΝΑΤΟ ή σε αποστολές του ΕΕ. Επίσης υπάρχει μια ε, διαρκή συνεργασία για το ζήτημα της ασφάλειας στη θάλασσα, της αντιμετώπισης των κυβερνοεπιθέσεων και της εκπαίδευσης στα στρατιωτικά θέματα στρατιωτικής συνεργασίας. Παραμένουν όμως κάποιες πολιτικές δυσκολίες. Και αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν πολύ, καλά, πολύ καλές επαφές σε ανεπίσημο επίπεδο μεταξύ στελεχών και φέτος συμφωνήθηκε να γίνονται τακτικές συνεργασίες, ε, τακτικές συναντήσεις. στο Ουαλία του 2014, στη Βαρσοβία του 2015, στις συνόδους κορυφής του ΝΑΤΟ, η παρουσία μας εκεί μας έδωσε τη δυνατότητα να ενισχύσουμε τη συνεργασία μας με τον ΝΑΤΟ. Όσον αφορά την Αφρικανική Ένωση. Και εδώ εστιάζουμε κυρίως στην βοήθεια προς τα κράτη της Αφρικής στον τομέα της ασφάλειας και την ενίσχυση της λεγόμενης αρχιτεκτονικής για την ασφάλεια στην Αφρική, άψα. προσπαθούμε να βοηθήσουμε στον τομέα της εντεμokratiας. Αυτό είναι κέρια σημασία για την εταιρική σχέση μεταξύ Αφρικανικής Ένωσης και Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της ασφάλειας. Επίσης, πέρα από αυτό το γενικό πλαίσιο, υπάρχουν και πιο συγκεκριμένες περιφερειακές ε, στρατηγικές, τοπικές στρατηγικές. Η συνεργασία μας εστιάζεται σε τρεις πτυχές. Πρώτα απ' όλα, να ε, ενισχυθεί ο διάλογος ανάμεσα στην πολιτική ε, ασφαλείας ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος είναι να φτάσουμε σε πλήρη επιχειρησιακή εφαρμογή της άψα και τρίτον να βελτιωθεί η χρηματοδότηση σε πρόσφατη σύνοδο, ε, συνάντησή μας ε, στην Αφρική είχαμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε τα ζητήματα αυτά περισσότερο σε βάθος. Τώρα, όσον αφορά τον ΟΑΣΕ, εστιάζουμε κυρίως αντιμετωπίση κρίσεων και υπάρχει στενή συνεργασία με τις ε, αποστολές του ΟΑΣΕ στη Γεωργία, στο Κόσοβο και την Ουκρανία. Κύριε Πρόεδρε, προχωρώ λίγο πιο γρήγορα, όσο πιο γρήγορα γίνεται, γιατί έχουμε και χρονικού περιορισμού και τα θέματα είναι πολλά που θα έπρεπε να καλύψω. Θα προσπαθήσω να το κάνω όσο το δυνατό πιο γρήγορα. Ωστόσο, δεν μπορεί κανεί να ξεχάσει τη σημασία του πάνελ για την Ανατολική Γειτονία. Για την Ανατολική Εταιρική Σχέση, μάλλον, τη ε, ΚΕΠΑ. Εδώ λοιπόν κάθε έξι μήνες στις Βρυξέλλες προσκαλούμε τους ηγέτες, ε, ε, του, μάλλον σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων γίνονται συναντήσει με τις ε, έξι χώρες ε, της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης και προσπαθούμε να δούμε προς, ε, πώς προχωρούν τα διάφορα θέματα που καλύπτει ο πολυμερής διάλογος στον οποίο συμμετέχουν εδώ η Αρμενία, το Ζερβαϊτζάν, η Λευκορωσία, η Γεωργία, η Μολδαβία και η Ουκρανία, καλύπτοντας θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Για παράδειγμα, πώς μπορούν εκείνες οι χώρες να συμμετέχουν σε ε, αποστολές αντιμετώπισης κρίσεως, κρίσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναφέρθηκε ήδη η πολύ σημαντική συμμετοχή της ε, Γεωργίας στην αποστολή στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, ένα παράδειγμα. Επίσης, ασχολόμαστε με ζητήματα που αποσχολούν τις χώρες εκείνες, όπως για παράδειγμα πώς εξελίσσεται η πολιτική γειτονίας, ή οι στρατηγικές επικοινωνίες, ποια θα είναι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτό το θέμα. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν συνεργαζόμαστε με τις χώρες της ανατολικής εταιρικής σχέσης. Άλλα πολυμερή φόρουμ τώρα. Συμμετέχουμε στο Περιφερειακό Φόρουμ ΑΖΕΑΝ. Θα γνωρίζετε ότι έχει ε, δημιουργηθεί και μια ομάδα επαφής ειδικά για την καταπολέμηση της πειρατείας ε, στις ακτές της Σομαλίας. Δεν θα πω όμω περισσότερε λεπτομέρειε τώρα εδώ. Μίλησα για τέσσερι πυλώνε και κάλεσα μόνο τον πρώτο μέχρι στιγμή. Συνεχίζουμε λοιπόν με τον δεύτερο για τη συμμετοχή τρίτων χωρών σε ε, μα. μας. Το εργαλείο το έχουμε για αυτή τη συνεργασία λέγεται το οι συμφωνίες πλαισίου για την συμμετοχή. 18 τέτοιες συμφωνίες έχουμε υπογράψει με 18 αντίστοιχες χώρες μία συμφωνία μία χώρα. Και έχουμε ως νούπο την συμφωνία με τη Δημοκρατία της Κορέας που θα λειτουργήσει και έχουμε και καλές προοπτικές με το Μαρόκο και ελπίζω ότι θα έχουμε και περισσότερες ειδήσει σχετικά με τα θέματα αυτά. Αυτές οι συμφωνίες εταιρικής πλαισιακής σχέσης. Είναι πολύ σημαντικές για να προωθήσουμε τη συνεργασία μας και να κάνουν εφικτό να υπάρχει η συμμετοχή και η εισφορά από όλες αυτές τις χώρες. Είναι με άνευ αυτοματισμό όμως αυτές οι συμφωνίες. Όταν έχουμε συγκεκριμένες απόστολες πάντα πρέπει να ληφθεί μια απόφαση από τα κράτη-μέλη κατά πόσο στη συγκεκριμένη δράση αυτή είναι μέσα στις επιθυμίες και τους πόθους τους να συμμετάσχουν. Τα μέλη της Πολιτικής ε, και Ασφαλείας Επιτροπής συζητούν και αν οι εταίροι το επιθυμούν να συμβάλλουν. Τα κράτη-μέλη θα δεχτούν αυτήν την συνεισφορά ή όχι. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τη συμμετοχή Έχουμε το 2014 15 χώρες συμμετέσχαν με περίπου 560 άτομα, 8% του συνολικού αριθμού των δυνάμεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό ήταν πολύ σημαντικό. Τα πιο πρόσφατα παραδείγματα ανέφερα ήδη την Γεωργία με την U4RCA η Σερβία επίσης ε, ειδικεύεται στην παροχή υγειονομικού προσωπικού στη Σομαλία, το Μαλί και την ε, Κεντροαφρικανική Δημοκρατία. Η Τουρκία, η Ελβετία και η Χιλή αναπτύσσουν μαζί μας στη Βοσνία αναπτύσσουν καλύτερα μαζί μας στην ε, Βοσνία δυνάμεις και το Μαρόκο έχει συμβάλει σημαντικά στο παρελθόν. Και έχουμε και σημαντική συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών και της ε, Τουρκίας στο Κόσοβο. Επέκεινα αυτή τη άμεση συμμετοχή έχουμε την Κολομβία που έχει συμμετάσχει τα τελευταία, τις τελευταίες εβδομάδες στην Αταλάντα και είχαμε πολύ καλή κατανομή αρμοδιοτήτων με άλλους εταίρους όπως είναι Κίνα και η Ιαπωνία και η Κορέα στο κέρας της Αφρικής θα είναι πολύ σημαντικές βομπτυχές στο μέλλον στις στρατηγικές μας ε, αναθεωρήσεις και τις θέσεις που πρέπει να αναλάβουμε. Για το διάλογο τώρα που έχουμε. Τις διάφορες μορφές διαλόγου είναι πολύ σημαντικές για να μπορέσουμε να εξετάσουμε την ενδεχόμενη συμμετοχή των χωρών αυτών στις ενεργειές μας, αλλά όπως είπα προηγουμένως αποτελούν και ένα μέσο περαιτέρω ανάπτυξης των σχέσεών μας σε θέματα ασφαλείας. Μας επιτρέπει επιπλέον να συζητήσουμε θέματα κοινού ενδιαφέροντος όπως είναι η εκπαίδευση, η κατάρτιση, οι βέλτιστες πρακτικές και παρόμοια θέματα. Αν στραφούμε προς το μέλλον τώρα και τις μελλοντικές προοπτικές. Σας είπα ότι έχουμε τη συμφωνία με την Κορέα που έχουμε ήδη υπογράψει, υπογράψει αυτή τη συμφωνία και περιμένουμε την κύρωσή της. Η Ελβετία θα μας δώσει τη δική της συνεισφορά και έχουμε και περισσότερες δυνατότητες για το μέλλον η ενίσχυση τώρα της ε, ικανότητας των εταίρων μας. Ο στόχος μας είναι να υποστηρίξουμε τους τοπικούς και περιφερειακούς εταίρους για να μπορέσουν να αναλάβουν την ευθύνη της διαχείρισης και της αντιμετώπισης των κρίσεων, καθώς και της πρόληψής τους. Νομίζω ότι έχει πει η ο διευθυντής μου για την, ε, ε, το training and Equip και την κοινή επικοινωνία. Ε, κάποια μέλη είναι νεόφυτα εδώ πέρα και δεν ξέρουν να μπορείτε να τα πείτε, να τα πείτε πάρα πολύ σύντομα. Υπήρξε μια κοινή επικοινωνία μεταξύ της ΥΠΑ εκπροσώπου και της Κομισιόν τον Απρίλιο για το πώς θα ενισχύσουμε την ικανότητα των εταίρων μας στα θέματα ασφάλειας και άμυνας. Και τώρα συνεχίζεται η δραστηριότητα αυτή. Δύο στόχους έχουμε σε αυτήν την κοινή προσέγγιση. Καταρχήν η ενίσχυση της ικανότητας για τα θέματα ασφάλειας βασιζόμενη σε όλα τα εργαλεία που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση προς την κατεύθυνση αυτή και να προχωρήσουμε προς μια πραγματικά εταιρική σχέση βοηθώντας τις χώρες αυτές για να μπορέσουν να προλάβουν και να διαχειριστούν κρίσεις. εστιάζουμε περισσότερο στην Αφρικανική Ήπειρο προς το παρόν, αλλά εμείς είμαστε πεπισμένοι ότι το έργο αυτό που έχει τον τίτλο Train and Equip, εκπαιδεύστε και εξοπλίστε, μπορείτε να, μπορεί να μεταλαποδευτεί και σε άλλες περιοχές του κόσμου. we can Ναι, μπορούμε να σταματήσουμε σε αυτό το σημείο για να δώσουμε και το λόγο στους επόμενους ομιλητές και μπορείτε να επανέλθετε στο δεύτερο γύρο, εάν συμφωνείτε. Ο κύριος Αλάμι Χαμαντάν έχει τώρα το λόγο. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καταρχάς να σας ευχαριστήσω για την πρόσκλησή σας στην ακρόαση αυτή, η οποία θα μου επιτρέψει να σας παρουσιάσω σύντομα τον ρόλο που διδραματίζει το Μαρόκο στα πλαίσια της κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας Ευρωπαϊκής Ένωσης και να αναφερθώ επίσης και στις μελλοντικές προοπτικές. Είδαμε αυτή τη στιγμή ότι ενισχύεται ο ρόλος της κοινή πολιτικής ασφάλειας και θα αποτελεί πλέον πυλώνα στην ευρωπαϊκή οικοδόμηση και επομένω επηρεάζει πάρα πολύ την άμυνα και την ασφάλεια και στην περιοχή της Μεσογείου. Έτσι λοιπόν τα κράτη εταίροι θα πρέπει βάσει μιας κοινή συμφωνίας να δούνε πώς μπορούν στην πράξη και επικρισιακά να συνεργαστούν στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουν όλες τις προκλήσεις που βαρύνουν την περιοχή της Μεσογείου. Το Μαρόκο ανέκαθεν θεωρούσε ότι ε, είναι πολύ σημαντικό να λαμβάνουν υπόψη όλες οι αμυντικές προκλήσεις των ε, εταίρων στη Μεσόγειο θα πρέπει να υπάρχει ένας επικοδομητικός διάλογος προκειμένου να υπάρχει πραγματικά μια αδιέρετη περιφερειακή πολιτική ασφάλειας η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική και θα πρέπει να λάβει υπόψη της όχι μόνο τη στρατιωτική αλλά και την ανθρωπιστική, οικονομική και κοινωνική πλευρά. Δεν θα πρέπει λοιπόν να δώσουμε βάρος μόνο σε μια πτυχή εις βάρος κάποιων άλλων. Στα πλαίσια λοιπόν αυτής της περιφερειακής αλληλεγγύης και συνειδητοποιώντα ότι έχουμε κοινέ προκλήσει, το Μαρόκο ανταποκρίθηκε θετικά στο αίτημα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, στέλνοντα κατά αυτόν τον τρόπο ένα τμήμα του στρατού του στα πλαίσια της επιχείρησης Αλτέα στη Βοσνία Αρζεγοβίνη. Ήταν η πρώτη αυτή σημαντική στρατιωτική επιχείρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία κατέδειξε ότι όντως υφίσταται ένας πολύ σημαντικός μια πολύ σημαντική σχέση συνεργασίας ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Μαρόκο. Το Μαρόκο όμως συμμετέχοντας στην επιχείρηση Αλτέα κατέδειξε τελικά ότι όντως ενδιαφέρεται για την αμυντική και στρατηγική πλευρά της σχέσης που έχει με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με τις όμορες του χώρες. Και κατά αυτόν τον τρόπο συμμετείχαμε και σε επιχείρηση του ΝΑΤΟ στο Κωσυφοπέδιο στην ε, Αϊτή, στην ακτή ε, του Ελεφαντοστού και στην ε, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Το Μαρόκο, συμμετέχοντας κατά αυτόν τον τρόπο σε όλες αυτές τις στρατικές επιχειρήσεις, έγινε ο εταίρος με την πιο σημαντική συμβολή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και χαίρεται ιδιαίτερα για το γεγονός ότι έχουν ευωδοθεί θετικά όλες αυτές οι στρατιωτικές επιχειρήσεις και μάλιστα υπήρξε μια πολύ επικοδομητική συνεργασία ανάμεσα στους Μαρακινούς και Ευρωπαίους στρατιώτες. Κατά αυτόν τον τρόπο βλέπουμε ότι όντως υπάρχει μια διαλειτουργικότητα η οποία είναι πολύ σημαντική για την επιτυχία οποιασδήποτε επιχειρησιακή στρατιωτικής επιχείρησης. Αν δούμε λοιπόν ακριβώς πώς είχε η συμμετοχή του Μαρόκου στο παρελθόν, πιστεύουμε ότι θα μπορέσει να αποτελέσει και σημείο αναφοράς για μελλοντικές τέτοιες συνεργασίες στα πλαίσια της κοινή ευρωπαϊκής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας. Η συμμετοχή των στρατιωτικών δυνάμεων του Μαρόκου σε επιχειρήσεις διατήρησης της ειρήνης αλλά και σε ανθρωπιστικές επιχειρήσεις μας οδήγησαν στο να αντλήσουμε τα εξή διδάγματα. Πρώτον, ότι μπορούμε να συνεργαστούμε επικοδομητικά με στρατούς άλλων χωρών. Δημιουργήσαμε πολύ θετικές σχέσεις. Μιλάμε αυτή τη στιγμή για πραγματικούς ε, συντρόφους που μας επέτρεψαν τελικά να έχουμε ακόμα και πολιτιστικές ανταλλαγές μεταξύ των δύο ε, στρατιωτικών δυνάμεων. Επίσης, οι συνδυασμένες αυτές επιχειρήσεις επέτρεψαν στρατιώτες του Μαρόκου να συνειδητοποιήσουν τι θα πει να δεσμεύεται κανείς σε, μια διεθνή επιχείρηση και ότι δεν συμμετέχουμε στο ΝΑΤΟ, συμμετείχαμε πολύ επικοδομητικά σε όλες αυτές τις πολυεθνικές πολυμερείς επιχειρήσεις. όλοι οι στρατιώτες μας ε, που πήγανε στο Κοσφοπέδιο και στην Βοσνία Ζεγοβίνη κατέδειξαν τον επαγγελματισμό τους και πραγματικά έδειξαν ότι μπορούν να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και των μελλοντικών περιστάσεων. Όσον αφορά τώρα τη συμμετοχή σε επιχειρήσεις των Ηνωμένων Εθνών, οι ε, μαροκινοί στρατιώτες έχοντας πολυετή εμπειρία κατάφεραν να συμβάλλουν αλλά να κερδίσουν και αυτοί πάρα πολλά πράγματα ε, στις σχέσεις που είχαν με τους ε, άλλους στρατιώτες και κατάφεραν επίσης να συμβάλλουν πολύ όσον αφορά την ανθρωπιστική διάσταση τη διαχείριση των κρίσεων. Είχαμε επίσης στρατό του Μαρόκου που συμμετείχε στη Βοσνία και στο Κοσμοπέδιο στα πλαίσια πολυεθνικών δυνάμεων και κατά αυτόν τον τρόπο συμβάλαμε στην μείωση της βίας, στην πάυση των συγκρούσεων και στο να επανακατασταθεί εκ νέου η ειρήνη και η ευημερία και πέρα από τις νέες προκλήσεις ε, που αντιμετωπίζουμε στον χώρο της ε, Μεσογείου και ιδίω όσον αφορά την ε, διάδοση των ε, όπλων μαζικής καταστροφής, όσον αφορά την εμπορία ανθρώπων και γενικότερα την τρομοκρατία. Όσον αφορά λοιπόν όλες αυτές τις προκλήσεις, θα ήθελε το Μαρόκο όλοι οι εταίροι στην περιοχή της Μεσογείου και της Ευρώπης να συμμετέχουν προκειμένου να συμβάλλουν στην καταπολέμηση όλων αυτών των προκλήσεων στα πλαίσια της γενικότερης έννοιας ότι η άμυνα είναι αδιαίτερη και μας αφορά όλους. Πρέπει λοιπόν να συνειδητοποιήσουμε ότι υποβαθμίζεται η κατάσταση της ασφάλειας στην περιοχή της Μεσογείου και στην περιοχή του Σαχέλ. Αυτό μας ανησυχεί όλους ιδιαιτέρως και είναι πολύ σημαντικό να αντιμετωπίσουμε όλες αυτές τις νέο αναδιόμενες προκλήσεις που προέρχονται από διάφορες τρομοκρατικές οργανώσεις, οι οποίες υποφελούνται από το γεγονός ότι πάρα πολλά κράτη στην περιοχή είναι ιδιαίτερα ασθενή και κατά αυτόν τον τρόπο απλώνουν όλο και περισσότερο τις τρομοκρατικές και εγκληματικές τους δραστηριότητες. Το Μαρόκο επιθυμεί λοιπόν να συμβάλλει θετικά προκειμένου να επιληθούν όλες αυτές οι κρίσεις, να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις και να δημιουργηθεί πραγματικά ένας ενιαίος μεσογειακός χώρος ασφάλειας και ελευθερίας. Έχουμε λοιπόν πλέον μια συμφωνία πλαίσιο με την Ευρωπαϊκή Ένωση που διαρθρώνει τη συμμετοχή του Μαρόκου στις επιχειρήσει διαχείριση κρίσεων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε την συμμετοχή αυτή και το Μαρόκο πρέπει να το πούμε είναι η πρώτη και μοναδική χώρα αυτή τη στιγμή από τη Μεσόγειο και γενικότερα από την Αφρικανική Ήπειρο που έχει συνάψει μια τέτοια συμφωνία. Στη συμφωνία αυτή τίθενται συγκεκριμένα οι αρμοδιότητες που θα αναλάβει το Μαρόκο, το ο ρόλος που θα δραματίσει και η σχέση που θα έχει με τις υπόλοιπες χώρες που συμμετέχουν σε μια τέτοια επιχείρηση. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα μας επιτρέπει πολύ γρήγορα και ομαλά να συμμετέχουμε σε τέτοιες επιχειρήσεις στο μέλλον χωρίς να χρειάζεται κάθε φορά να διαπραγματευόμαστε και μια νέα συμφωνία συνεργασίας. Θα συμβάλλει λοιπόν αυτή η συμφωνία στη διαχείριση κρίσεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν μετά από αρκετού μήνες διαπραγματεύσεων υπέγραψε τη συμφωνία αυτή με το Μαρόκο. Αυτό αποτελεί πραγματικά αναγνώριση του, της συμβολής του Μαρόκου καθώς επίσης και της πολιτικής βούλησης που διαθέτει το Μαρόκο προκειμένου να συμβάλλει σε τέτοιες επιχειρήσεις. Χαιρόμαστε λοιπόν πάρα πολύ για την δυνατότητα αυτή που μας δίνει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να συμμετέχουμε σε δράσεις ΚΕΠΑ. Μέσω τη συμφωνία αυτή επισημοποιείται λοιπόν η συμμετοχή του Μαρόκου στη διαχείριση των κρίσεων και αυτό αποτελεί ένα πολύ σημαντικό νέο κρίκο στι στρατηγικέ αυτέ εταιρικέ σχέσει που θέλει να συνάψει το Μαρόκο με την Ευρωπαϊκή Ένωση βλέπουμε κατά αυτόν τον τρόπο ότι όντω υπάρχει μια κοινή κατανόηση και εμπιστοσύνη μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Μαρόκου, όπω άλλωστε έχουμε δει πάρα πολλέ φορέ στο παρελθόν. Στα πλαίσια λοιπόν τη αναθεωρημένη πολιτική γειτονία τη Ευρωπαϊκή Ένωση, το Μαρόκο θεωρεί ότι θα πρέπει ο πηγησιακό διάλογο να ενδυναμωθεί όσον αφορά το ζήτημα των κοινών προκλήσεων και αναφέρομαι εδώ πέρα στη μετανάστευση, την παράνομη μετανάστευση, τη διαχείριση των κρίσεων, την παράνομη, το λαθρεμπόριο χημικών ραδιενεργών όπλων, την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Είναι πολύ σημαντικό να καταφέρουμε από κοινού να δείξουμε αλληλεγγύη και να έχουμε μια κοινή δραστηριοποίηση για να καταπολεμήσουμε τις κρίσεις αυτές. Αυτό όμως μπορεί να γίνει μόνο αν έχουμε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο στα πλαίσια του οποίου θα μπορεί το κάθε κράτος μέλος και ο κάθε εταίρος Ευρωπαϊκής Ένωσης να λαμβάνει συγκεκριμένη δράση. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Thank you, sir. Uh, και εμείς σας ευχαριστούμε. Θα δώσω το λόγο τώρα. Στον κύριο Ρορική. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι και είναι μεγάλη τιμή για μένα να παρεμπτύσκουμε σήμερα εδώ μιλήσω στην εκ μέρου των Ηνωμένων Εθνών, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ξεκινώ λέγοντας ότι είμαι επικεφαλής ε, γραφείου του ΟΗΕ της Βρυξέλλες, το οποίο εκπροσωπεί το Τμήμα Πολιτικών Υποθέσεων της Γενικής Συνέλευσης, το Τμήμα των ε, Ειρηνευτικών Αποστολών και το τμήμα υποστήριξη ε, των επιτόπιων αποστολών. Δημιουργήθηκε το 2011 στι Βρυξέλλε και ο στόχο ήταν ε, να δημιουργηθούν ε, σχέσει στι Βρυξέλλε κυρίω με την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και άλλου φορεί. Και πιστεύω ότι η δημιουργία του γραφείου αυτού δείχνει την σημασία που αποδίδουν τα Ηνωμένα Έθνη στις σχέσεις τους με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με χαρά λοιπόν αποδέχτηκα την πρόσκλησή σας για να συζητήσουμε με τους φίλους εδώ στο πάνελ και με τα μέλη της Επιτροπής σας τη σχέση αυτή Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΟΗΕ. Πρώτα απ' όλα να πω ότι θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα ε, κατάλληλη χρονική στιγμή για να συζητούμε τη σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΗΕ για πολλούς λόγους. Μια αποστολή της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και της Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων επισκέφτηκε την έδρα των Ηνωμένων Εθνών την προηγούμενη εβδομάδα και ε, εκείνοι τους οποίους συνάντησαν ε, μου μετέφεραν ότι ε, έκανε ιδιαίτερα που είχαν πολύ ψηλού επίπεδου και ψηλής ποιότητας συζητήσεις με εκπροσώπους του ΟΗΕ και εκπροσώπους του Γενικού Γραμματέα. Προφανώ ο ΙΕ παρακολουθεί με μεγάλο ενδιαφέρον τα τεκτενόμενα στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το ψήφισμα την προηγούμενη εβδομάδα ε, για την, ε, τη, τη σημασία του ρόλου του ΙΕ ε, είναι κάτι το οποίο το καλωσορίζουμε και νομίζω ότι διευκολύνει και τη συνεργασία μας. Όπως γνωρίζετε στον ΟΗΕ το προηγούμενο έτος ήταν έτος αναστοχασμού. Προετοιμάστηκαν ε, διάφορες εκθέσεις ανάμεσα στις οποίες και μια αξιολόγηση ε, των ειρηνευτικών αποστολών ε, τα τελευταία 15 χρόνια. Η προηγούμενη σχετική εκθέση ήταν έκθεση Ιμπραχήμη, σίγουρα γνωρίζετε. Ενώ ταυτόχρονα η Ευρωπαϊκή Ένωση και εκείνη ξεκινάει την παγκόσμια, ε, μια αναθεώρηση της στρατηγικής της όσον αφορά την εξωτερική πολιτική της, το Global Strategy, επομένως μπορούμε αυτές τις δύο διαδικασίες κάπως να τις συνδυάσουμε. Θα ήθελα να σας δώσω μια αίσθηση των δυσκολιών και του πλαισίου μέσα στο οποίο κινούνται σήμερα τα Ηνωμένα Έθνη. Τι σκεπτόμαστε σε σχέση με αυτές τις προκλήσεις και το πώς μπορεί η σχέση ΟΗΕ-Ευρωπαϊκής Ένωσης να ενισχυθεί. Οι παρευρισκόμενοι στην αίθουσα φαντάζομαι είναι ειδικοί στα ζητήματα, στα, τεκτενόμενα στον κόσμο. Επομένω, δεν χρειάζεται εγώ να σας πω ότι ευξάνονται οι ενόπλες συγκρούσεις. 28 είναι ερευνητικέ αποστολές ε, ε, του ΟΗΕ που είναι, ε, έχουν αναπτυχθεί αυτή τη στιγμή ανά τον κόσμο. Βλέπετε που βρίσκονται αυτές στο χάρτη που εμφανίζεται αυτή τη στιγμή στην οθόνα. Υπάρχουν στα αριστερά οι παραδοσιακές αποστολές ανοκράνων και στα δεξιά οι αποστολές πολιτικού χαρακτήρα που ε, είτε πρόκειται για ε, παροχή κανόνων υπηρεσιών του Γενικού Γραμματέα, είτε για άλλου είδου πολιτικέ ε, διαδικασίε διευκόλυνση πολιτικού διαλόγου. Επίση υπάρχουν και οι ειδικοί απεσταλμένοι του Γενικού Γραμματέα με συγκεκριμένε αρμοδιότητε ο καθένα του. Γνωρίζουμε όλοι, για παράδειγμα, το έργο του κυρίου Λεόν στην Λιβύη ή του ειδικού απεσταλμένου στην Συρία. είναι αυξάνεται ο αριθμός των κρίσεων και των συγκρούσεων, αλλά αυξάνεται, αλλάζει επίσης και ο χαρακτήρας τους. Γίνονται όλο και περισσότερο περιφερειακές οι συγκρούσεις. Το οποίο σημαίνει ότι χρειάζεται και μια περιφερειακή ανταπόκριση σε αυτές, με λιγότερο περιορισμό στα ε, εθνικά σύνορα, στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε, αντιδρούμε σε αυτές. Ενώ επίσης η ανταπόκριση μας πρέπει να προσαρμοστεί και στον ασύμετρο χαρακτήρα των ε, νέων κρίσεων. Και φυσικά η όποια ανταπόκριση στην κρίση δεν ε, υφίσταται σε ένα πολιτικό κενό, πρέπει να, γίνει, πρέπει να εντάσσεται σε μια γενικότερη στρατηγική. Αναφέρθηκα ήδη στους ειδικούς απεσταλμένους στη Λιβύη και τη Συρία. Ε, υποστηρίζουμε την ε, μετάβαση στο Μαλί, στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία υποστηρίζουμε τη μεταβατική κυβέρνηση που προετοιμάζει τις επικείμενες εκλογές και στο Νότιο Σουδάν συνεχίζεται η υποστήριξη σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη και εύθραυστη ε, ειρηνευτική διαδικασία. Στην διαφάνεια που βλέπετε εδώ. Όπως έλεγα, χρειάζεται η ανταπόκρισή μας να, γίνεται, να είναι πιο ενισχυμένη εξαιτίας της αλλαγής στο χαρακτήρα των κρίσεων και των συγκρούσεων. Έχει τονίσει ο Γενικός Γραμματέας την σημασία που έχει τα ανθρώπινα δικαιώματα να, ξεκινούν, ε, ξεκινάει η περάσπιση τους ήδη από την αρχή μιας ειρηνευτικής ε, ιδιαίτερα όσον αφορά την προστασία των αμάχων. 28 Σεπτεμβρίου 2015, λοιπόν, διοργανώθηκε υπό την αιγίδα του Πρόεδρου Ομπάμα μια σύνοδος κορυφή για τι ειρηνευτικέ αποστολέ, Με χαρά διαπίστωσα ότι οι Ευρωπαϊκέ χώρε δεσμεύτηκαν ουσιαστικά να προσφέρουν ε, αυτό που μπορούν να προσφέρουν ε, στην σύνοδο αυτή. Το βλέπουμε ήδη στο Μάλι, στο Μαλί αλλά και σε άλλες αποστολές ειρηνευτικές του ΟΗΕ που υποστηρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό είναι μια θετική εξέλιξη νομίζω. Είπα επίσης ότι το 2015 ήταν έτος αναστοχασμού. Τον Απρίλιο του 2015 ο Γενικός Γραμματέας ε, δημοσιοποίησε την έκθεσή του με τίτλο ε, «Μια εταιρική σχέση για τις ειρηνευτικές αποστολές, Partnership Peacekeeping», λέγοντας πόσο σημαντική είναι η συνεργασία με τρίτους οργανισμούς για σε αυτές τις αποστολές και ιδιαίτερα στην γρήγορη ανταπόκριση σε κρίσεις. Ομάδες άμεσης ε, αντίδρασης, άμεσης επέμβασης ή ιδιαίτερα όσον αφορά την προστασία των αμάχων και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτές οι μονάδες ε, άμεσης επέμβασης πιστεύω ότι θα έχουν πολύ σημαντικό ρόλο να παίξουν συνεργαζόμαστε με την ε, Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και άλλα κρατημέλη για να δούμε πώς μπορεί η Ένωση να συμμετέχει, συμμετάσχει σε αυτές τις ομάδες. Τρεις προτεραιότητες είναι την άποψή μας οι πιο σημαντικές, συνθεματολογικά θα έλεγα άνθρωποι, people, πολιτική, politics και partnerships, συνεργασίες. Όσον αφορά του ανθρώπου σημαίνει ότι πρέπει να δίνουμε μεγαλύτερη έμφαση στη διαμεσολάβηση και στην πρόληψη των συγκρούσεων. Όσον αφορά την πολιτική, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να, να, να, να, οποιαδήποτε ενέργεια του ΟΗΕ να εντάσσεται σε μια γενικότερη στρατηγική πολιτική η οποία να μπορεί να έχει διάρκεια και ε, σταθερότητα. Και τέλος, partnerships, συνεργασίες. Στην έκθεση του Γενικού Γραμματέα αναδεικνύεται ότι χρειάζεται να συνεργαζόμαστε με οργανισμούς όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους, γιατί τα προβλήματα είναι περίπλοκα και δεν μπορεί κανείς να τα αντιμετωπίσει μόνος του. Χαίρομαι να... Με χαρά διαπιστώνω ότι η συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι υποδειγματική και μπορεί βέβαια να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο. Και το ανέφερε και η Κλάρα, δεν θα δώσω ακόμα περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά θα ήθελα Ευχαριστώ την προσοχή σας στο έγγραφο Strategic Partnership, το οποίο αναφέρεται σε αυτές τις στρατηγικές συνεργασίες. Ε, σε ποιους τομείς θα εστιαστεί η στρατηγική συνεργασία, δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΙΕ, τα επόμενα τρία χρόνια, ως το 2018. Το κυριότερο για εμάς είναι η άμεση ανταπόκριση μετά το, την, την υπερψήφιση ενός ψηφίσματος του Συμβούλου Ασφαλείας του ΟΗΕ να ξεκινά όσο το δυνατόν πιο γρήγορα η, η επέμβαση, η ανταπόκριση, η αποστολή μιας ε, δύναμης ό,τι χρειάζεται. Επίσης, Καλωσορίζουμε το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ανακοινώσει ότι θα αναλάβει πρωτοβουλία στον τομέα του capacity building της βελτίωσης των ικανοτήτων ε, των κρατών στον τομέα της ασφάλειας. Τώρα, όσον αφορά τους μηχανισμούς που έχουμε στη διάθεσή μας για τον πολιτικό διάλογο, υπάρχουν πολλοί και διάφοροι τέτοιοι μηχανισμοί. Σας έδωσα το παράδειγμα της, από, της ε, ε, ε, επίσκεψης των εκπροσώπων της ΑΦΕΤ την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά πολύ συχνά έχουμε και συνεργασία με την Αντιπρόεδρο Μογκερίνη πολύ συχνά τα μέλη της PSC, της, Πολιτικής και, ε, ε, της Επιτροπής Πολιτικής και Ασφαλείας, επισκέπτονται την έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Ε, αντιστρόφως, ο Γενικός Γραμματέας Περιφερειακών Οργανισμών του ΟΗΕ, ο κ. Λασσός, συχνά έρχεται στην, ε, στις Βρυξέλλες για να ενημερώσει. Όσον αφορά την πρόληψη συγκρούσεων, έχει δημιουργηθεί ένα εργαστήριο, ένα, μιας συνάντηση ετήσια ε, στην οποία συζητάμε από κοινού ε, εκπρόσωπο του ΙΕ και εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ανοιχτά θέματα πρόληψης συγκρούσεων. Και επίσης άλλα όργανα τα οποία ήδη αναφέρθηκαν. Θα έλεγα λοιπόν ότι έχουμε στη διάθεσή μας πολλούς μηχανισμούς πολιτικού διαλόγου και χρειάζεται αυτός ο ουσιαστικός πολιτικός διάλογος, γιατί θα διαπιστώνεται διαπιστώνει κανείς απλώ κοιτώντα τι προτεραιότητες των ΜΕΝ και των ΔΕ ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο ΙΕ συνεργάζονται ή εργάζονται μάλλον σε παράλληλε ή τι ίδιε προτεραιότητε πολύ συχνά. Ένα παράδειγμα καλή συνεργασία ήταν η εργαζονται μαλλον σε παραλληλε η τις ιδιε προτεραιοτητες πολυ συχνα ενα παραδειγμα καλη συνεργασιας ηταν η κεντροαφρικανικη δημοκρατια Το ίδιο στο Μαλί, εδώ συνεργαζόμαστε για την μεταρρύθμιση του τομέα της ασφάλεια. Και εδώ λειτουργούν τα πράγματα πολύ καλά και στη Σομαλία βρέθηκε μια πολύ ενδιαφέρουσα ε, συνεργασία που εμπλέκει και την Αφρικανική Ένωση. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμες και οι παράλληλες αποστολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και οι αποστολές γέφυρα όπως στην περίπτωση της Κεντροαφρικανικής ε, Δημοκρατίας αλλά επίσης και οι, αποστολές, οι περιπτώσεις στις οποίες μια αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραδίδει σε μια αποστολή του ΟΗΕ. Αυτοί είναι οι τρεις τρόποι με τους οποίους συνεργαζόμαστε ε, επί τόπου. Το παράδειγμα της κεντροαφρικανικής δημοκρατίας που ήδη το ε, συζητήσατε δεν θα ε, το ξανααναφέρω, αλλά είναι κατά την άποψή μου μια περίπτωση όπου τα πράγματα λειτουργήσαν πολύ ορθά. ορθά. Κλείνω λέγοντα, κύριε Πρόεδρε, ότι έχει στρατηγική σημασία για εμά η σχέση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι ένα τομέα αυτό στον οποίο θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε περισσότερο. Σε πολλού τομεί, μάλλον, θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε περισσότερο. Ένα κρίσιμο ζήτημα είναι το ζήτημα τη χρηματοδότηση. Πώ μπορούν να βοηθηθούν οι αποστολέ του ΟΗΕ, οι οποίε ανταποκρίνονται σε μια επίγουσα κρίση επιτόπου. Ε, και εδώ η συνεισφορά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορεί να είναι πολύ σημαντική. Επίση η αποστολή παρατηρητών σε εκλογέ είναι ένα τομέα στον οποίο μπορούμε να συνεργαστούμε. Ή η αξιοποίηση των καλών υπηρεσιών του, του, του ε, προκειμένου να διοργανωθούν εκλογε Και αυτό είναι ενα τομεα στον οποίο θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε. Η συμμετοχή ευρωβουλευτών στι αποστολέ παρατήρηση εκλογών, όπω είπα. Σήμερα είναι η πρώτη φορά που ο εκπρόσωπος ε, του γραφείου του ΟΕΑ, στο οποίο προείσταμε, ε, έρχεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να κάνει μια παρουσίαση. Χαίρομαι ιδιαίτερα για αυτή την πρόσκληση και ελπίζω να επαναληφθεί κάτι τέτοιο και στο μέλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Μπορεί να υπάρξει ένα δεύτερο γύρο, αλλά θα είναι πολύ σύντομο. Καθηγητά κόψε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ για αυτή την πρωτοβουλία της ε, πρόσκλησης και της δικής μου. Είναι ένα πολύπλοκο θέμα. Το βασικό ερώτημα είναι πώς μπορεί να χρησιμοποιήσει καλύτερα αυτές τις εταιρικές σχέσεις η Ευρωπαϊκή Πολιτική Άμυνας και Ασφάλειας. Έχουμε κάνει πολλή έρευνα τα τελευταία τέσσερα χρόνια για αυτό το ζήτημα. Να σας πω καταρχήν ότι υπάρχουν δύο οπτικές γωνίες που έχουμε για το θέμα αυτό την οπτική γωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θέλει να ενισχύσει την πολιτική ασφάλειας και άμυνας, να έχει σημαντικό αντίκτυπο, να κινητοποιεί τα κράτη-μέλη υπέρ των ε, κοινών θεμάτων συμφέροντος. Αυτό μπορεί να μην οδηγήσει σε συμμετοχή των κατών μελών, αλλά τουλάχιστον αυτή είναι η κύρια κατεύθυνση που πρέπει να έχουμε για να έχουμε μια σωστή πολιτική και άμυνας και ασφάλειας και υπάρχει και μια μη ευρωπαϊκή γενική προσέγγιση που αφορά το άλλο μου κασκέτο δεν είναι αυτή καθεαυτή η πολιτική άμυνα και ασφάλεια τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά πρέπει να αντιμετωπιστεί μέσα σε μια παγκόσμια ε, λειτουργία διακυβέρνηση τη άμυνα και τη ασφάλεια, ενίσχυση των πολυπολικών και παγκόσμιων οργανισμών και να προσπαθήσουμε να εξασφαλίσουμε τον παγκόσμιο μακροχρόνιο διάλογο. Δεν είναι πάντα σε ε, αρμονία τα, οι δύο αυτοί στόχοι μπορεί να υπάρχουν πάντα στρατηγικά συμφέροντα των κρατών μελών τα οποία δεν συνάδουν με αυτό το οποίο είναι το καλύτερο για την, ε, για τη συνολική δράση των άλλων φορέων που είναι τέλει. Πρέπει λοιπόν να έχει κανείς εξ αρχή στο μυαλό του ότι υπάρχουν τέτοιου είδους εντάσεις. Η επόμενη τώρα διαφάνεια. Παρακαλώ. Η CSDP αυτή καθε αυτή όπως ελέγχθη τονίζει ότι η διατήρηση της ειρήνης είναι μια εταιρική σχέση από τα γενοφάσια της. Η πολιτική άμυνας και ασφάλειας ξεκίνησε γιατί είχε πραγματικά ενσωματωμένα τα στοιχεία της στρατηγικής εταιρικής σχέσης τόσο στρατιωτική ε, διάσταση όσο και στην πολιτική διαχείριση κρίσεων. Ξεκίνησε με τη συνεργασία Ευρωπαϊκής Ένωσης ΝΑΤΟ για πολλούς λόγους λοιπόν που δεν έχει επιτευχθεί πλήρως αλλά υπήρξε περισσότερη πολιτική επιρροή ορισμένων σκεπτικιστών που θέλουν τον ΝΑΤΟ να είναι ο κύριος χώρος για την ευρωπαϊκή στρατιωτική δράση και όχι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εν πάση περιπτώσει ήταν σημαντική αυτή η διαδικασία για μεταλαμπάδευση γνώσεων και για πολιτικούς λόγους. Το ίδιο και με τον ΟΗΕ η δράση των αστυνομικών δυνάμεων του ΟΗΕ τη Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν πάρα πολύ σημαντική και εκεί το Μαρόκο υπήρξε της Αποστολή τη Ευρωπαϊκή Ένωση στην Βοσνία γιατί προηγουμένω ήταν στον ΟΗΕ, στην αποστολή του ΟΗΕ και έτσι υπήρξε μια ε, ομαλή μετάβαση. Είχε κάθε συμφέρον να περάσει και στι δραστηριότητε που στη συνέχεια πέρασαν στην ηγεσία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Μου ζητήσα να μιλήσω για τα κράτη-μέλη και του φορείς, τις δύο αυτές πτυχές. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπογραμμίσω ότι το επίπεδο θεσμοποίηση των αυτονόμων οργανισμών είναι αξιοσημείωτο στην περίπτωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν υπάρχει κανένας άλλος τέτοιος περιφερειακός οργανισμός ο οποίος σε τόσο έντονο και σε τόσο πλήρες επίπεδο έχει θεσμοποιήσει τη σχέση που έχει μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ενωμένων Εθνών και επίσης την πολύ στενή συνεργασία με τον ΝΑΤΟ. Ξέρουμε ότι υπάρχουν και πολιτικά προβλήματα. ή άτυπες σχέσεις βέβαια είναι πάρα πολύ σημαντικές σε διαδρομικό επίπεδο. Υπάρχουν τροποποιήσεις σε αυτή την πολιτική και όταν μιλάμε για πολιτική άμυνας και ασφάλειας πάντα θα έχουμε το αγκάθι του ΝΑΤΟ που κάποτε πρέπει να αντιμετωπιστεί και όχι με τρόπους που είναι απλώς και μόνο άτυποι. Μία μικρή παρατήρηση, μία εταιρική σχέση μπορεί να και πηγή ισχύω και αδυναμίας. Στη δική μας περίπτωση φαίνεται ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για να υπάρξει συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε θέματα ασφάλειας, να υποστηρίξουν την κοινή πολιτική αμήνας και ασφάλειας, να έχουμε στατικές σχέσεις, των οποίων η πολιτική άμυνας και ασφάλειας είναι ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Υπάρχει και αυτή η δυνατότητα να έχουμε ενίσχυση των κοινών πρακτικών. Ε, Επίση μπορεί να το δει κανεί και ω αδυναμία, ότι μόνη της η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να κινητοποιήσει αρκετά κράτη-μέλη ακούσαμε στο προηγούμενο πάνελ τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο ΟΕΕ Εθνών για να μπορέσουν να, να υπάρξουν συνεισφορές στρατιωτικών δυνάμεων εν γέρος. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα, όπως ξέρετε. Το να υλοποιηθεί μια εντολή και να οδηγήσει σε παρουσία στρατευμάτων είναι ακόμα πιο δύσκολο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μια πρόκληση λοιπόν και για μας και όχι μόνο για τον ΟΗΕ. Επόμενη διαφάνεια τα τελευταία 12 χρόνια. Αναφέρθηκαν συμφωνίε πλαισίου, εταιρικέ συμφωνίε πλαισίου με 18-17 χώρε. Αν δούμε τώρα όλε αυτέ τις αποστολέ είναι σχεδόν 50 κράτη εκτό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. κάποια τώρα είναι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε ήταν έξω, έχουν συμβάλει σε αποστολέ άμυνα και ασφάλεια. Είναι σημαντικό ο αριθμό. και δείχνουν τη σημασία της ΕΠΑ, της πολιτικής άμυνας και ασφάλειας. Έχουμε την Γιοφόρ στην Βοσνία, εκεί υπήρχε μια διάδοχη αποστολή στην αποστολή του ΝΑΤΟ και οι διάφορες χώρες άλλαξαν τα ρούχα τους και τα έβαλαν αλλιώ από τον ΝΑΤΟ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ή υπάρχουν χώρες όπως η Νορβηγία που υποστηρίζει ιδιαίτερα την ΕΠΑ, όχι μονάχα με στρατεύματα, αλλά και με την συμμετοχή της στο σχηματισμό μάχης των σκανδιναμικών χωρών. Σημαντικό είναι αυτό που δέχουμε ένα μέλος που δεν είναι μέλος του ΟΗΕ. Έχουμε τον Καναδά και τη Ρωσία που έχουν συμμετάσχει. Είχαν προβλήματα στρατηγικής αερομεταφοράς και χωρίς τα Αντώνο της Ρωσίας δεν θα μπορούσε να τα καταφέρει. Ενώ συγχρόνως η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ρωσία ήταν σε μεγάλη ένταση λόγω της κρίσης γεωργίας. Αυτό δείχνει ότι μπορεί να υπάρξει μια διαδικασία διαχωρισμού παρά τις δυσκολίες υπάρχουν χώρες που είναι έτοιμες να συμβάλλουν σε τέτοιες ε, επιχειρήσεις. Σημαντικό είναι και η παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών στην διαχείριση κρίσεων και σε αποστολές ε, εκπαίδευσης στο Μάλι, στην ε, Σομαλία και στην Λέξη του Κωσυφοπεδίου. Επόμενη διαφάνεια. Υπάρχουν διάφορες διαστάσεις συνεργασίας με τρίτες χώρες. Υπάρχει η τεχνική και επιχειρησιακή πλευρά που αναφέρθηκε προηγουμένως. Υπάρχει η δυνατότητα οι χώρες αυτές να φέρουν στρατεύματα, ειδικέ ε, εμπειρογνωμοσύνες, τη δυνατότητα στρατηγικής αερομεταφοράς, αλλά υπάρχει και η πολιτική πτυχή συμμετοχή στη διαδικασία αυτή που φυσικά είναι τμήμα του οράματος ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης δείχνει επίση ότι οι στρατηγικέ εταιρικέ σχέσεις οι οποίες ξεκινούν για άλλους λόγους, παραγωγικά χάρη Κορία, Κορέα και η Ιαπωνία, ξεκίνησαν μέσω του Ελεύθερου εμπορίου και ακολουθούν με την συνεργασία σε δράσεις ε, ΕΠΑ. Αυτό δείχνει το πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει μια πλήρη εταιρική σχέση η οποία δεν αφορά μόνο το εμπόριο αλλά και άλλες πτυχές συνεργασίες πολιτικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πολύ σημαντικό να εξασφαλίσει την ορατότητα, να είναι εύστοχες οι ενέργειες της ΕΠΑ και να υπάρχει ευρύτερος αντίκτυπος, να υπάρχουν ευρύτεροι ευρωπαϊκοί συνασπισμοί χωρών έξω και από το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης επόμενη ο διαφάνεια. Οι χώρες αυτές μπορούν να καλύψουν σημαντικά κενά, αλλά επίσης μπορούν να επιτύχουν πιο πολυμερείς αποστολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορούν να αυξήσουν τον περιφερειακό χαρακτήρα, ήταν σημαντική η αλθέα η αποστολή αυτή που έπαιξε σημαντικό ρόλο υποστήριξε την αποστολή του ΟΙΑ και είχαν επίσης και χώρες όπως η Νότια Αφρική, η Βραζιλία ως περιφερειακή εταίροι οι οποίοι συνέβαλαν πάρα πολύ στην αποστολή αυτή και της έδωσαν μια πολυμερή διάσταση. Αλλά βέβαια δεν είναι ο καλύτερος πάντα τρόπος να συμμετέχουν ε, περιφερειακές δυνάμεις οι οποίες μπορούν να έχουν και δικές τους υστεροβουλίε. Το 2005 η ΑΣΕΑ ήταν πολύ σημαντική όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση έστειλε μια αποστολή στο Άτζε στην ε, Ινδονησία και οι άλλες χώρες επίσης συμμετέσχαν σε αυτήν την ε, διαδικασία. Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχει και μια μεγαλύτερη δυνατότητα γεωγραφικής εμβέλειας των ενεργειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα από τις συνεργασίες με τις χώρες αυτές. Ανέφερα ήδη τα την κληρονομιά της συνεργασίας Ευρωπαϊκού, ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης ΝΑΤΟ. Επόμενο σημείο. Ποιες είναι οι προκλήσεις ως ε, μηχανισμός. Έχουμε ένα υψηλό επίπεδο επισημοποίησης αυτών των μορφών ε, συνεργασίας. Έχουμε διευθύνσεις επιτροπές που συνδέουν την Ευρωπαϊκή Ένωση με το ΝΟΗΕ. Έχουμε τους αξιωματικούς σύνδεσης που είναι μια μεγάλη επιτυχία. Υπάρχει σταθερή διασύνδεση μεταξύ των φορέων, μοιράζονται την κοινή επιχειρησιακή κουλτούρα για αυτές τις αποστολές. Νομίζω ότι είναι πολλά που μπορεί να γίνουν σε αυτό το επίπεδο και οι δύο φορείς έχουν δείξει μια μεγάλη δέσμευση και προσήλωση στο να ενισχυθεί η διασύνδεση μεταξύ τους και δεν είναι απλώς πολιτική ρητορική. Νομίζω σε θεσμικό επίπεδο και οι δύο πλευρές έχουν κοινέ αξίες και κοινά θεματολόγια. Όλα αυτά όμως θα πρέπει να οδηγήσουν σε κοινού πόρους, σε πολιτική υποστήριξη, στα κράτη-μέλη να συμμετέχουν περισσότερο. Αυτό είναι το πρόβλημα. Μπορείτε να έχετε όση θεσμοποίηση θέλετε, αλλά τελικά οι πόροι όλων αυτών των οργανισμών θα πρέπει να τίθενται από κοινού. Ορισμένες φορές υπάρχουν διαφορές σε στατηγικό επίπεδο μεταξύ κρατών μεταξύ φορέων μπορεί τα κρατημένα να ακολουθούν διαφορετικές ατζέντε μέσα στους φορείς, αλλά ποτέ δεν είναι τόσο σημαντικές αυτές οι διαφορές ώστε να θέσουν ένα φιβόρο τις αποστολές. Είναι δύσκολη βέβαια η διαδικασία συντονισμού, είναι μεγάλο το άχθο το οποίο εμπλέκεται, ιδίω αν είναι χώρε οι οποίε είναι τρίτε. Υπάρχουν συζητήσει που πρέπει να γίνουν για χρηματοδοτικά θέματα, για νομικά θέματα και τελικά θα στείλουν 5-6 φαντάρου και η παρά, αλλά μακροχρόνια έχει σημασία το αποτέλεσμα. Η Τουρκία, η Τουρκία ήταν πάντα ένα σημαντικό εταίρο για το ΝΑΤΟ. Υπάρχουν άλλα κράτη τη Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν θέλουν να ενισχύσουν ιδιαίτερα τη συνεργασία με την Τουρκία, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο ίσω μπορεί να αντιμετωπιστεί τώρα με το τροποποιούμενο στρατηγικό και πολιτικό κλίμα. Ενδιαφέρον να δούμε ότι η υπηρεσία εξωτερικής δράσης μπορεί να κάνει και μια ιεράρχηση των εταίρων μέσα στις εταιρικές σχέσεις και να δώσει έμφαση σε αυτούς που θέλουν να συνεργαστούν ακόμα περισσότερο από τις 50 αυτές χώρες. Κάτι που είναι επίσης σημαντικό είναι να έχουμε μαθήματα τα οποία βγάζουμε από αυτές τις εταιρικές σχέσεις. Ο ΙΕ έχει πολύ μεγάλη εμπειρία στις εταιρικές σχέσεις. Από τη δεκαετία του 1960 αντλεί εμπειρία γιατί χρειάστηκε να ε, συνεργαστεί με διάφορες φορείς, με τον Οργανισμό Αφρικανικών Κρατών παραδείγματος χάρη. Είναι σημαντικό να μιλήσουμε και με την ε, Αφρικανική Ένωση. Δεν έχουμε στεγανά μεταξύ των διαφόρων αυτών οργανώσεων. Έχουμε διάφορα φόρα όσο δύσκολο φαίνεται, όπου τα διδάγματα μπορούν να αντλούνται εν κοινό μεταξύ διαφόρων φορών. Επόμενη διαφάνεια. όλοι ξέρουμε και το αναφέρατε ότι πρέπει να υπάρχει μια συνολική προσέγγιση, περιεκτική προσέγγιση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επενδύσει πολύ κεφάλαιο στο να έχει την σωστή θεματολογία και τη σωστή ρητορική και αυτό είναι πολύ σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω τώρα. Εκεί που μπορεί να επιτευχθεί η μεγαλύτερη πρόοδος και θυμάμαι αυτά που είχε οργανώσει ο κύριος Φαν Όρδεν το 1912, είναι η συνεργασία με την Αφρικανική Ένωση. Είναι σημαντική ικανότητα, αλλά δεν υπάρχει ακόμα μια συντονισμένη δραστηριότητα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μια εξισορροπημένη ίσως προσέγγιση. Ο ΙΕ προσπαθεί να συνεργαστεί με την Αφρικανική Ένωση και το ΝΑΤΟ επίσης και εδώ μια καλύτερη συνεργασία μεταξύ όλων των φορέων είναι πολύ καλή. Τώρα, Ναι, ναι, νομίζω τα έχω πει τα περισσότερα, μπορούμε να περάσουμε πιο στο επόμενο. Και νομίζω, ναι, ναι, ναι, εντάξει. Για να κλείσω λοιπόν. Εντάσεις μεταξύ μέσα στην ΕΠΑ θα πρέπει και αυτές να αντιμετωπιστούν. Θα πρέπει να ξέρουμε ότι δεν έχουμε εδώ μία πλήρως αυτοματοποιημένη διαδικασία ενίσχυση τη ΕΠΑ. Είδαμε τα τρία-τέσσερα χρόνια να υπάρχει έλλειψη ενδιαφέροντος σε αυτές τις πολιτικές, ιδίως σε σχέση με την κεντροαφρικανική δημοκρατία. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον ΟΗΕ μιλάμε πάντα για την όρεξη περιορέξεως των κρατών μελών. Αυτό πολλές φορές ε, ε, οδήγησε καλύτερη συνειδητοποίηση στου πολιτικού για το πώ πρέπει να δαπανώνουν τα χρήματα αυτά. Αυτή πρέπει να μια ευρύτερη συζήτηση, η οποία θα είναι απλώ τεχνική. Πού πάμε, ποια είναι τα κέρια θέματα, ποιε είναι οι βασικέ στρατηγικέ ιδέε, τι θέλουν τα κρατημέλη, τι θα πρέπει να κάνουμε και θα πρέπει να υπάρξει και μια γενικότερη αναθέωση τη ευρωπαϊκή πολιτική ασφάλεια και άμυνα σε μια συζήτηση που διαδραματίζεται εδώ και 12 χρόνια και εδώ επιτέλου να το αντιμετωπίσουμε με τον σωστό τρόπο. Και θα ήθελα επίση να πω κατά δεύτερο και δευτερεύοντα λόγο ότι είμαστε εδώ πέρα σε μια διαδικασία, όπω είπατε προηγουμένω, αναφερθήκατε στι διασκέψει κορυφή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να εξασφαλίσουν οι Ευρωπαίοι ότι μέσα στα όρια τα οποία έχουν, τα οποία είναι περιοριστικού χαρακτήρα, θα πρέπει να τηρούν τι υποσχέσει του. Πολλέ φορέ εγώ ω ακαδημαϊκό δεν εντυπωσιάζομαι ιδιαίτερα το το ακριβώ αντίθετο με αυτέ τι συνεισφορέ που δίνουν οι χώρε αυτέ όπω είναι η Γερμανία, παραδείγματο χάρη, και θα ήθελα να βλέπω από την πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση να χρησιμοποιήσει καλύτερα αυτέ τι ευκαιρίε, όχι μόνο από την πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση, να υπάρχει εκπροσώπηση ω φορέα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά να δούμε τα κέρια ευρωπαϊκά κράτη, όχι του ε, Συνήθις υπόπτους να προχωρούν σε σημαντικότερες συνεισφορές προς τη διατήρηση ειρήνης από το ΡΟΙΑ, είτε εμπλέκεται η ΕΠΑΑ ή όχι. Και έχουμε και ένα μεγάλο ελεφαντάκι στο δωμάτιο που είναι η Κίνα. Πώς θα μπορέσει η Κίνα να μεταφέρει τη δύναμή της σε μια πραγματικότητα με το να αντιμετωπίσει το θέμα της ταχείας αντίδρασης. Θα δημιουργήσουν μια δύναμη ταχεία αντίδρασης 8.000 και θα δώσουν και δισεκατομμύρια δολάρια για την αφρικανική συνεργασία. Μπορούμε λοιπόν να έχουμε καλύτερες στρατηγικές ε, σχέσεις και με την Κίνα θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση μας με τον ΟΗΕ να δει πώς θα πρέπει να αντιμετωπίσει την Κίνα και να την εμπλέξει ώστε να η συμμετέχει στις ε, δεσμεύσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν θα πρέπει να δούμε σαν μια παγκόσμια εταιρική σχέση την ΕΠΑ. Πρέπει να ενισχύσουμε και τον ΟΗΕ και πρέπει να δούμε και τι γίνεται έξω και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Μία διαφάνεια μόνο θέλω να δείξω ακόμα όσον αφορά τη συμβολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω ότι γίνονται τόσο σημαντικές προσπάθειες όσον αφορά τη δημιουργία όλο και περισσότερων εταιρικών σχέσεων στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας. Πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να ενδυναμώσουμε την ΕΠΑ με τους εταίρους, πώς οι εταίροι μπορεί να ενδυναμωθούν από την ΕΠΑ Νομίζω ότι είτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης θα πρέπει να δημιουργήσουν περισσότερο ένα φόρουμ, ένα κόμβο ανταλλαγής πληροφοριών, ανταλλαγής θετικών διδαγμάτων από όλε αυτές τις εμπειρίες. Είναι πολύ σημαντικό επίσης να δώσουμε μια νέα όθηση στη σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ. Αντιμετωπίσουμε προβλήματα στη σχέση αυτή εδώ και 11 χρόνια και είναι πολύ σημαντικό κάποια κράτη-μέλη να συμβάλλουν προκειμένου να αναζωογονηθεί η σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ. Σας ευχαριστούμε κύριε καθηγητά. Το λόγο τώρα έχουν οι ευρωβουλευτές. Πρώτος ο κύριος Όρντεν. Σας ε, ευχαριστώ πρόεδρε. Να ευχαριστήσω καταρχάς όλους τους συμμετέχοντες στο πάνελ για τις εξαιρετικές τους παρουσιάσεις. Εγώ αυτή τη στιγμή Προετοιμάζω μια έκθεση για την υποεπιτροπή μας όσον αφορά την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Αφρικανική Ένωση, τα Ενωμένα και όλους τους άλλους διεθνείς οργανισμούς στους οποίους αναφερθήκαμε. Θα ήθελα λοιπόν προτού φύγετε να μιλήσω και μαζί σας διμερώς για να ανταλλάξουμε κάποιες ιδέες, γιατί είμαι σίγουρο ότι μπορώ να μάθω πολλά πράγματα από σας. Κάποιες ερωτήσεις βέβαια θα ήθελα να θέσω σαφώς. Ένα από τα προβλήματα που έχουμε αντιμετωπίσει είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί όλο και περισσότερο να σταθεί στα πόδια της και να γίνει ένας αυτόνομος παράγοντας στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας, προσπαθεί να προσδώσει τον εαυτό της όλο και νέους ρόλους, μολονότι ε, δεν μπορεί να βρει πάντα τους απαραίτητους ή τους κατάλληλους εταίρους. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν κάποιες δραστηριότητες τις οποίες θα μπορούσε να επιτελέσει πολύ πιο καλά και αποτελεσματικά η Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να καταρρύψουμε αν θέλετε οποιοδήποτε διαχωρισμό αυτή τη στιγμή μπορεί να καταρρυψουμε αν το οποιοδηποτε διαχωρισμο αυτη ανάμεσα στην στρατιωτική και μη στρατιωτική πτυχή και να αναλάβει δράση η Ευρωπαϊκή Ένωση στους τομείς εκείνους που μπορεί πραγματικά να αποφέρει μια προστιθέμενη αξία. Μια ερώτηση προς τον κύριο Κίνα ποιος είναι αυτός ο βασικός παράγοντας που διέπει τη λογική των Ηνωμένων Εθνών όταν αποφασίζει αν μια ειρηνευτική αποστολή θα είναι καθαρά αποστολή Ηνωμένων Εθνών ή αν θα είναι μια αποστολή που τελικά θα ανατεθεί σε κάποιον εξωτερικό παράγοντα, τοπικό ή ακόμα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρετε ότι ε, πολλές φορές δυσκολευόμαστε να καταλάβουμε σε διάφορες περιοχές του κόσμου όπως ε, στην Κεντροφρικανική Δημοκρατία ή στο Τσάντ, ποιος κάνει ακριβώς τι και πώς έχουν αντεθεί τελικά οι αρμοδιότητες, πώς αποφασίζει τελικά ο Οργανισμός των Μένων Εθνών για το αν θα αναθέσει σε κάποιον εξωτερικό παράγοντα μια συγκεκριμένη επιχείρηση. Και μια ερώτηση για την κυρία Γκάνστλαντ όσον αφορά τις συνεργασίες και τις εταιρικές σχέσεις. Ποια είναι η σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες της, παράκτης χώρες της Βόρειας Αφρικής. Ξέρετε, αυτή τη στιγμή έχουμε την έκτακτη αυτή κατάσταση του προσφυγικού ζητήματος και αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να λάβουμε κάποιες αποφάσεις για να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση στη Μεσόγειο. Αυτό προφανώς θα επηρεάσει και τις χώρες της Βορείου Αφρικής. Μήπως θα μπορούσατε να μας φωτίσετε λίγο περισσότερο ως προς αυτά. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Καν έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ. Να σας ευχαρώ και εγώ για τις παρουσιάσεις σας. Αναμφίβολα ο κόσμος αλλάζει και εξελίσσεται και είναι θετικό να έχουμε ως το δυνατόν περισσότερη συνεργασία. Μόνο έτσι θα καταφέρουμε να επιτύχουμε σε όλες αυτές τις προσπάθειές μας. Μία ερώτηση τώρα θα ήθελα να θέσω προς τον κύριο Αλάμι Χαμεντάνη, ο οποίος αναφέρθηκε στην τρομοκρατία, στην περιφερειακή διάσταση τρομοκρατίας. Γνωρίζουμε ποιες είναι οι παγκόσμιες επιπτώσεις του Ισλαμικού κράτους και συμφωνώ μαζί σας ότι πρέπει να έχουμε μια κοινή ενιαία προσέγγιση, όχι μόνο όμως στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Μόνο κατά αυτόν τον τρόπο θα καταφέρουμε να καταπολεμήσουμε το Ισλαμικό κράτος, αν έχουμε μια κοινή κατανόηση και κοινή προσέγγιση όσον αφορά την πρόκληση αυτή. Το Μαρόκο προφανώς έχει μια πολύ μεγάλη πλούσια ιστορία, έχει κάποιους πολύ σημαντικούς θεσμούς που θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε. Πώς μπορεί λοιπόν να διαρθρωθεί η συνεργασία με το Μαρόκο, πώς μπορείτε εσείς να συμβάλλετε προκειμένου να επέμβουμε σε όλη αυτή την περιοχή για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που έχουμε εκεί. Πρόεδρο, σας ευχαριστούμε. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να θέσω δύο ερωτήσεις, να κάνω μάλλον δύο παρατηρήσεις. Η πρώτη προς την κυρία Γκάγκσλαντ, όσον αφορά την ανατολική εταιρική σχέση. Υφίστανται διαφορές και ανάμεσα στις χώρες της αντολικής εταιρική σχέσης όσον αφορά τις συγκρούσεις που έχουμε σε διάφορες περιοχές, όπως για παράδειγμα στην Ουκρανία. Ξέρετε ότι η Λευκορωσία είχε συμμετάσχει σε κάποιες στρατιωτικές ασκήσεις οι οποίες βασικά στρέφονταν εναντίον της ε, παρουσίας κάποιων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, από την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, χωρών της ε, Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης. Νομίζω λοιπόν ότι κάποιες χώρες θα μπορούσαμε να τις αντιμετωπίσουμε κάπως ξεχωριστά. Στον τομέα πάντως της άμυνας και της ασφάλειας, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να αξιολογήσουμε τις υφιστάμενες απειλές εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή την παρατήρηση κάνω και προς τον κύριο Ρόρι Κίνα. Είχαμε μια ανταλλαγή απόψεων με τον κύριο Ίγντορ πριν από λίγο και καταφέραμε να αποτιμήσουμε την κατάσταση στην κεντροφρικανική δημοκρατία και αυτό μας κάνει να σκεφτόμαστε λίγο τα χρονοδιαγράμματα της ανάπτυξης των στρατιωτικών δυνάμεων επιτόπου. Δηλαδή αυτές, αυτή η γεφυρωτική επιχείρηση από ό,τι φαίνεται θα επιμηκυνθεί αυτή τη στιγμή ακριβώς επειδή πρέπει να κερδίσουμε λίγο χρόνο προτού ολοκληρωθεί η επιχείρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω λοιπόν ότι και αυτό το παράγοντα θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Να δούμε δηλαδή πώς λειτουργούν αυτές οι γεφερωτικές επιχειρήσεις και για αυτές ήταν πολλές φορές δύσκολο να εξασφαλίσουμε τη συμβολή των κρατών μελών. Ποια είναι λοιπόν η δική σας η άποψη όσον αφορά την ταχύτερη ανάπτυξη των μάχημων μονάδων σε τέτοιες καταστάσεις, σε τέτοιες περιστάσεις, ενώ περιμένουμε δηλαδή να θεσπιστεί μία επίσημη επιχείρηση, να ξεκινήσει η πρώτη επιχειρησιακή φάση μίας επιχείρησης των Ηνωμένων Εθνών. Νομίζω ότι αυτό που έχουμε δει στην πράξη είναι ότι στο εφιστάμενο πλαίσιο δυσκολευόμαστε πολύ να συντονιστούμε ήδη στα πρώιμα στάδια δεν ξέρω λοιπόν αν θα καταφέρουμε όντω να εφαρμόσουμε το δικό σα το σχέδιο των ΗΕ για τι ερωτικέ επιχειρήσει. Ενδεχομένω να είναι κάπω πρόημο. Λοιπόν, μπορείτε να απαντήσετε με τη σειρά αυτή στι ερωτήσει που έθεσα, αλλά είστε σύντομοι, παρακαλώ πολύ. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και τα... τους... εκείνου που έθεσαν ερωτήματα. Για τον κύριο Βανότεν. θέτει το ερώτημα για τις ε, σχέσεις μας με τις παράκτης ε, χώρες της Βόρειας Αφρικής. Στη σημερινή συγκυρία. Το πρώτο που μπορώ να πω είναι ότι κάνουμε μεγάλες προσπάθειες να αναπτύξουμε σχέσεις με αυτές τις χώρες μέσω των αντιπροσωπιών μας εξηγώντας τους τα διάφορα στάδια των επιχειρήσεων και το ίδιο ισχύει και για τον διοικητή της επιχείρησης Σοφία ο οποίος ίσως έχει κάνει επαφές με αυτές τις χώρες. Πιο συγκεκριμένα για την, με την Τινησία και με την Αίγυπτο θα ζητήσουμε να μας δώσουν την έγκρισή τους όταν κατά τη διάρκεια της φάσης 2 υπάρχει πιθανότητα να ε, σταματώνται πλοία τα οποία φέρουν τη σημαία τους γιατί προφανώς ε, ε, τα πλοία αυτά θα βρίσκονται υπό τη δική τους δικαιοδοσία. Ένα παράδειγμα μιας κάποιων συγκεκριμένων επαφών που έχουμε με τις χώρες αυτές. Επίσης, τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ έχουν ενημερωθεί και έχουμε συχνά επαφές με την ομάδα πολιτικού συντονισμού του ΝΑΤΟ για την επιχείρηση Σοφία. Σχέση με το δικό σας ερώτημα, κυρία Πρόεδρε. Συμφωνώ πλήρως ότι ε, πρέπει να υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση ανάμεσα, απέναντι στις διαφορετικές χώρες της ανατολικής εταιρικής σχέσης. Δεν είναι όλες το ίδιο. Εμείς στον τμήμα στο οποίο εργάζομαι βρισκόμαστε σε συνεχή επαφή με τους συναδέλφους που ασχολούνται με τον πολιτικό διάλογο με τις χώρες αυτές, έτσι ώστε να γνωρίζουμε πώς εξελίσσεται αυτός ο πολιτικός διάλογος και έχουν και προσωπική εμπειρία στο πάνελ που διοργανώσαμε για να συζητήσουμε ζητήματα ασφαλείας με τις χώρες της ανατολικής εταιρικής σχέσης διαπίστωσα ότι ήταν πολύ χρήσιμο να κάνουμε αυτή τη συζήτηση να έχουμε ένα διάλογο μαζί τους να τους εξηγήσουμε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση βλέπει τα πράγματα και πως κινείται και τελικά αυτός ο διάλογος να εστιαστεί σε πιο πρακτικά ζητήματα αυτό είναι πολύ τιμό, νομίζω. Ευχαριστώ. Μεσολαμή. Ας συνεχίσουμε με τη σειρά την προηγούμενη, λέει η Πρόεδρος. Απαντώ σε ένα ερώτημα του κ. Χάνιν. Το Μαρόκο έχει μια προσέγγιση τριπλή, δηλαδή που αφορά και την ασφάλεια και τα κοινωνικο-οικονομικά ζητήματα και την θρησκεία. Όσον αφορά το πρώτο, προσπαθούμε να ενισχύσουμε τους δικαστικούς θεσμούς και δημιουργήθηκε ένα ειδικό τμήμα για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας. Συνεργαζόμαστε ιδιαίτερα με την Ισπανία και την Γαλλία για την ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά τα κοινωνικο-οικονομικά θέματα. Δημιουργήθηκε από το 2007 μια πρωτοβουλία για την καταπολέμηση της ανεργίας και τη βελτίωση των συνθήκων ζωής σε όλους τους τομείς. Και τρίτον, και κατά την άποψή μου σημαντικότερο, είναι το θέμα της ε, θρησκείας, όπου έχουμε προσπαθήσει να ε, κρατήσουμε μακριά τις ε, ψεύτικες ιδέες που οδηγούν στην ριζοσπαστικοποίηση. Εμείς προωθούμε ένα Ισλάμ το οποίο βασίζεται στην ανεξιθρησκεία και σέβεται μάλλον την ανεξιθρησκεία και την... Ε, και σε κέντρο για την εκπαίδευση ημάμιδων Έχουμε ε, ήδη πάνω από 400 ε, ε, ε οι οποίοι συμμετέχουν σε, σε εκπαιδευτικά προγράμματα από όλη την Αφρική. Με αυτές τις τρεις λοιπόν προτεραιότητες προσπαθούμε να συνεισφέρουμε και εμείς στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας στην Αφρική. Ευχαριστώ πολύ για το ερώτημα. Για τον κύριο Βανόρντεν, σας ευχαριστώ πολύ και προσβλέπω στην έκθεσή σας η οποία είναι υπό επεξεργασία τώρα. Από τη δική μας οπτική γωνία στα Ηνωμένα Έθνη, όταν αναφέρεστε στο θέμα της προστέμενης αξίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εμείς βλέπουμε την προστέμενη αξία σε διάφορες πτυχές της ε, ΕΠΑ. Και σίγουρα είναι το έργο σας για την ε, εκπαίδευση στον τομέα της ασφάλειας, ε, στον τομέα της ε, επιβολής του νόμου, την δημιουργία γενικά ικανοτήτων. Όλα αυτά ήταν πάρα πολύ επιτυχή και εμείς το είδαμε αυτό και στην Ευρωπαϊκή Αποστολή Εκπαίδευση στο Μαλί. Για το άλλο ερώτημά σας, για το πώς τα πράγματα αυτά ε, αντιμετωπίζονται σε ό,τι αφορά την αλλαγή των πύλων το ριχάτιν, δηλαδή την αλλαγή ε, και την ε, ε μετάδοση της κοιτάλης από μία ομάδα σε μία άλλη. Πολλές φορές βλέπουμε στον ΟΗΕ όταν γίνεται συζητήσει μεταξύ του Γενικού Γραμματέα και του ε, Συμβουλίου Ασφαλείας υπάρχουν τα θέματα της πολιτικής θέλησης και της ταχύτητας που είναι πάρα πολύ σημαντικά και πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ίσως μια σωστή αντιμετώπιση εδώ πέρα είναι να βλέπουμε συγκεκριμένα παραδείγματα. Συζητήσαμε προηγουμένως το θέμα της κεντροαφρικανικής δημοκρατίας όπου λόγω της ε, σοβαρότητας της κατάστασης πήγε πολύ ε, πρώιμα η ευρωπαϊκή αποστολή και μετά η αποστολή του ΟΗΕ πήγε να βοηθήσει για να εξασφαλίσει την ασφάλεια στο αεροδρόμιο και σε ορισμένα κέρια σημεία. Και έτσι δημιουργήθηκε η ευκαιρία για μένα πια μια ευρύτερη και πολυμερή αποστολή του ΟΗΕ που επέτρεψε λοιπόν σε, στα θέματα που ήταν εκεί να τεθούν υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών. Και έρχομαι στο ερώτημα της πρόεδρος μας τώρα. Νομίζω ότι η αποστολή EU4 ήταν σημαντική σε προσθέμενη αξία γιατί μπήκε σε ένα κρίσιμο σημείο εκείνη την ε, εποχή και έδειξε μια πάρα πολύ κέρια ευκαμψία γιατί η αρχική εντολή της ήταν μοναχά 6 μήνες και μετά από τη, μια διαδικασία διαλόγου με τα Ηνωμένα Έθνη η Ευρωπαϊκή Ένωση συμφώνησε να παρατείνει την ε, αποστολή αυτή για ένα σύνολο 9 μηνών για να εξασφαλίσει ότι η γεφύρωση λειτουργούσε και, και υπήρξε και κάποια δύναμη που θα ήταν στο τέλος της περίοδου γεφύρωσης. Το ερώτημα τώρα είναι γιατί αυτό θα ήταν πιο εύκολο με, μία, με ένα σχηματισμό μάχης. Αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον και αυτό πιστεύω είναι γιατί όπως ανέφερε και ο κύριος Ικλόντι προηγουμένως η, η δημιουργία μιας δύναμης επιτόπου είναι κάτι το οποίο είναι χρονοβόρο. Για τους σχηματισμούς μάχης δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα γιατί δεν υπάρχει μια διαδικασία τέταρτης γενιάς όπως λέγεται με ένα σχηματισμό μάχης. Η ομάδα αυτή υπάρχει και απλώς είναι μια απόφαση ανάπτυξης αυτής της ε, μονάδας του σχηματισμού μάχης. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι λαμβάνουν υπόψη τα κράτη-μέλη. Καταρχήν αν υπάρχει η πολιτική θέληση να γίνει κάτι τέτοιο και δεύτερον αν υπάρχει η απαραίτητη χρηματοδότηση γιατί κοστίζουν οι σχηματισμοί μάχης. και στο διάλογο αυτό για την ταχεία ανάπτυξη θα πρέπει να συζητήσουμε για αυτά τα δύο ζητήματα, το θέμα της πολιτικής θέλησης και της χρηματοδότησης και να δούμε αν μπορούμε να βρούμε ένα κοινό έδαφος. Τέλος, να πω επίσης ότι, ότι με το σενάριο των ε, σχηματισμών μάχης ο σχεδιασμός ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει αρχίσει να ευθυγραμμίζεται πλήρως με αυτή τη λογική και θα πρέπει να πω ότι ο Γενικό Γραμματέα εκτιμά ιδιαίτερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και χαίρεται για τι προσπάθειε που καταβάλει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όποτε μπορεί ε, πάντα να είναι στι Βρυξέλλες είναι πάντα πρότιμο να έλθει ενώπιον τη Ολομέλεια και ο αναπληρωτής Γενικό Γραμματέα έχει παρουσιαστεί σε συνεδριάσεις τη ε, ΑΦΕΤ και τη Επιτροπή Εξωτερικών ε, Ανθρωπινών Δικαιωμάτων πριν από πέντε μήνες. Ευχαριστώ πολύ καθηγητά, καθηγητά Coops, για το θέμα το οποίο έθεσε ο κύριο Φανόρντο για το αν η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να επιληθεί όλων αυτών των καθηκόντων που αναφέρουν και διαγράφουν τα επίσημα έγγραφα. Ξέρω ότι υπάρχουν συζητήσει για το κατά πόσο η ΕΠΑ θα πρέπει να περιοριστεί στις κέρδη, στα κέρια καθήκοντά της, κάτι το οποίο θα αντιβαίνει στην ιδέα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να διαδίδει το πλήρες φάσμα δυνατοτήτων και να παραμένει ανοιχτή σε όλα τα εργαλεία. Εδώ θέλω να έρθω στην ιδέα που υπάρχει σε πολλά εγγραφά και τις συνθήκες ότι η ενίσχυση φορέων όπως ο ΙΕ ως στοιχείο πολιτικής, εξωτερικής πολιτικής δεν είναι αντίθετο με τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βλέπουμε τώρα με την κρίση των προσφύγων που υπάρχει ο κίνδυνος να γίνει στρατιωτικοποιημένη κρίση. Είναι σημαντική η στιγμή η Ευρώπη να εστιάσει και στις αιτίες αυτού του προβλήματος και η συνεργασία με τον ΟΗΕ σε αντιμετώπιση κρίσεων δεν είναι μονάχα αλτρουιστικό, είναι και το ίδιο συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια φάση όπου μια κρίση έχει φτάσει πια στο κατόφλι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το να υποστηρίξουμε τις στρατηγικές δράσεις του ΟΗΕ τώρα και στο μέλλον θα σήμαινε ότι σε τελική ανάλυση η σταθερότητα και η ασφάλεια της ευρωπαϊκής περιφέρειας θα ενισχυθεί. Ευχαριστώ πολύ, λέει και η πρόοδος, πρόεδρος. Ένα σχόλιο για αυτά που είπε ο κύριος Κίντ. Ξέρω πόσο καλή είναι η ευρωπαϊκή δράση στην κεντρική, στην κεντροαφρικανική δημοκρατία. Δεν ήταν θέμα, γιατί η UFO θέμα χρόνου και ανάπτυξης, ήταν κάπως αντίστροφη η κατάσταση από ό,τι στην περίπτωση της Μινούσκα. Το ερώτημά μου ήταν πώς φαντάζεστε τους πολυδάπανους αυτούς σχηματισμούς μάχης να παίζουν το ρόλο της γέφυρας εκεί. Δεν θέλω λοιπόν να τα διαφυσβητήσω αυτά, αλλά ήμουνα παρούσα εκεί και είδα πόσο καλά λειτουργήσε η EU4. Ε, και λοιπόν, Δεν έχω το χρόνο να ε, συνοψίσω. Θέλω να ευχαριστήσω όμως τα μέλη του πάνελ για την εξαίρετη συνεισφορά τους και βασιζόμαστε πάντα σε τέτοιου συζητήσεις για να βελτιώσουμε την έκθεση του Jeffrey Van Orden για θέματα όπως αυτό. Θα συνεχίσουμε λοιπόν αυτή τη συζήτηση που είναι πάρα πολύ σημαντική, είναι έγκυη επίκαιρη και σημαντική. Σας ευχαριστώ πολύ. Η επόμενη μας συνεδρίαση θα είναι στις 30 Νοεμβρίου και να σας πληροφορήσω επίσης ότι στις 3 Δεκεμβρίου έχουμε μια έκτακτη συνεδρίαση της ΣΕΔΕ που αφορά δύο θέματα. Η αξιολόγηση μαζί με την ΑΦΕΤ και την διακοινοβουλευτική αντιπροσωπεία με την Ουκρανία μια αξιολόγηση της εφαρμογής της ε, συμφωνίας του Μίνσκ και δεύτερον ανταλλαγή απόψεων μάλλον μια ακρόαση για την, τις ε, εταιρείες παροχής τις ιδιωτικές εταιρείες παροχής ασφάλειας.